La séance est ouverte. Άρχεται η συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω τον πρέσβη και πρόεδρο Μάριο Μόντι, τον γερουσιαστή συγγνώμη και τον κύριο Μάριο Μόντι, ο οποίο θα κηρύξει και την έναρξη τη ε, ακρόαση. Μα τιμάει η παρουσία σα, κύριε Μόντι. Είδατε την ημερήσια διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση να σας δώσω καταρχάς μια πληροφορία για την ε, μυρίσκεται σε μια πρόταση. Προβλεπόταν για απόψε ε, μια σειρά ακροάσεων στο πλαίσιο της Προσωρινής Επιτροπής ΤΑΞ. Είχαν προβλεφθεί μεταξύ άλλων ο κύριος Μέρφη, ο οποίος όμως έχει ένα πρόβλημα ε, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τα τρένα, δεν ξέρει αν θα φτάσει και πότε αν φτάσει. Αν δεν φτάσει την ώρα που προβλέπετε, θα φτάσει αργότερα, δεν είναι όμως ούτε αυτό σίγουρο. Επίσης, συγκρίσιμο πρόβλημα έχει και ο κύριος ε, Σκοτ, που ήταν ο προηγούμενος επικεφαλής ε, για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου tax ruling ε, από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, που δεν μπορεί καθόλου να παραστεί. Προτείναμε όμως να έρθει σε μια μεταγενέστερη συνεδριασή μας, ε, μάλλον στις 23 ε, Ιουνίου. Όμως, έχουμε την επιβεβαίωση της παρουσίας της κυρίας ε, Ρέντιν και του κυρίου Ντελτούρ. Άρα, τι σας προτείνω. Να ακούσουμε ευθύ αμέσω τον πρόεδρο Μόντι και τις ανακοινώσεις του Προέδρου, οι οποίε είναι σημαντικές για τη συνέχεια των εργασιών μας και μπορούν να δείξουν σε μια ανταλλαγή απόψεων, να τις μεταφέρουμε για το πέρας των ακροάσεων, στο τέλος δηλαδή της μερικής διάταξης, αν συμφωνείτε. Να σας πω ότι για τις λοιπές ακροάσεις γνωρίζετε όπως συνήθως ότι είναι δημόσια συνεδρίασή μας, πόσο μάλλον αυτό πρόκειται για ακρόαση και επομένως όλες οι χρήσιμες γλώσσες για τα μέλη της Επιτροπής μας και για τους ακροατές μας ή για τους, ε, τα μέλη ε, του πάνελ διατίθενται. Υπάρχει λοιπόν ταυτόχρονη μετάφραση. Και έχουμε και τα έγγραφα εργασία στις γλώσσες αυτές. Κύριε Γερουσιαστά, αγαπητέ Μάριο Μόντι, από την αρχή των εργασιών μας ήδη η Επιτροπή μας είχε θεωρήσει ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια ανταλλαγή απόψε μαζί σας και πρέπει να σας πω ότι εσείς είχατε ο ίδιος προτείνει να έρθετε πριν κάτι σας προσκαλέσω. Η παρουσία σας, η μαρτυρία σας είναι πάρα πολύ πολύτιμες διότι γνωρίζουμε ότι εσείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που είχατε στα τέλη της δεκαετίας ε, του 90 και στις αρχές ε, της δεκαετίας του 2000, εσείς ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχατε δρομολογήσει την όλη διαδικασία που είχε ως στόχο να τεθεί ένα τέλος σε κάποια στοιχεία αφύσικων, ανταγωνισμού μεταξύ των τότε κρατών μελών σε σχέση με την φορολογία των επιχειρήσεων όταν είχαμε την εντύπωση ότι είχαμε προχωρήσει σε εναρμόνιση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των κανονισμών που αφορούσαν τον οικονομικό βίο. Είχαμε λοιπόν ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό, τη νομική βάση για τον ενιαίο χώρο, αν θέλετε. Όταν λοιπόν θεωρούσαμε ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, εισήχθηκε το ενίο νόμισμα ένα ακόμη στοιχείο που μας επέτρεπε να καταργήσουμε εξάπαντος ε, μία μορφή ιδιαίτερος ε, ύπουλου θα έλεγα ανταγωνισμό, αυτό δηλαδή τον νομισματικό ανταγωνισμό στις δημόσιες ε, πολιτικές ε, παρέμενε ένα μεγάλο ερωτηματικό που ήταν η για τον επιχειρήσεων και με τη δική σας όθηση και παρότρινση ελήφθησαν σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες τότε. Σήμερα το 2014-2015 διαπιστώνουμε ότι πόρο απέχουμε του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και καλό είναι να ξαναγίνει μια ισχυρή πολιτική πρωτοβουλία σε ένα πλαίσιο που έχει μεταβληθεί και από οικονομικής πλευράς και σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Ένωσης, γιατί είμαστε 28 πλέον χώρες μέλη και από πολιτικής πλευράς βλέπουμε επίσης αλλαγές, ιδίως με ορισμένε αποκαλύψεις του τύπου που έριξαν τους προβολείς δημοσιότητας τα αριθμητικά στοιχεία, τα αποτελέσματα της κατάσταση. και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, στις οποίες πρέπει να δοθεί μια πολιτική απάντηση. Γι' αυτό και η μαρτυρία σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, Ιδίω εφόσον δεν υπήρξατε απλά και μόνο ο αρμόδιος επιτροπός για αυτά τα θέματα πριν από κάποια χρόνια, αλλά στο μεταξύ έχετε ασκήσει σημαντικές ε, αρμοδιότητες στη χώρα σας και πιστεύω ότι σας επιτρέψει να πάρετε και, και άλλες γνώσεις και εμπειρίες ως υπεύθυνο για τη διαχείριση σημαντικών χαρτοφυλακίων. Άρα είναι ακόμα πιο πολύτιμη η μαρτυρία σας. Έχουμε την Ελίζα Φερέιρα, την συνεισηγήτρια που είναι παρούσα ε, και τον Μικάλ Τόιρερ που είναι συνεισηγητής αλλά έχει και αυτός κάποιο πρόβλημα να φτάσει. Θα έρθει όμως ε, ο Σονούπο. Αν συμφωνεί η Ελίζα Φεραίρα, να δώσουμε καταρχά το λόγο στον πρόεδρο Μόντι και έπειτα εκπρόσωποι των ομάδων μπορούν να πάρουν το λόγο. Κύριε Μόντι, έχετε το λόγο, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ άλε μεγάλη μου τιμή που εμφανίζομαι εδώ μπροστά σας. Αποκαλύψατε ότι είχα αναλάβει την πρωτοβουλία ελάχιστα διπλωματική βέβαια, να σας προτείνω ότι θα αποδεχόμουν ενδεχόμενη πρόσκληση να εμφανιστώ στην Επιτροπή σας. Όλα αυτά δείχνουν ότι δέχθηκα τη σύσταση αυτής της Επιτροπής σαν κάτι πολύ σημαντικό πλευράς θεσμικής και πολιτικής. Όσον αφορά την πολιτική και φορολογική πολιτική, αλλά και την πολιτική γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολούθησα και από μακριά και εκ του σύνεγγυ της ακροάσεις σας, τις αρχικές σας δραστηριότητες όλους αυτούς τους μήνες. η ιδιαιτέρως από μία πτυχή που είμαι σίγουρος ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπικότητα και τη δραστηριότητα του Προέδρου. Ήτι, χρησιμοποίησατε πολύ συναισθηματισμό που δημιουργήθηκε στο κοινό λόγω κάποιων αποκαλύψεων και κάποιων γεγονότων και ταυτόχρονα είχα τη δυνατότητα να χειριστείτε αυτό το κύμα που δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο που έχω την εντύπωση ότι μεγιστοποιείτε τις πιθανότητες οι εργασίες σας να καταλήξουν συγκεκριμένες και χρήσιμες προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη σύγκρουση που θα, που θα ήταν στήρα αν ακολουθούσα προσέγγιση. Κάτι που ήθιστε, δυστυχώς, στις πολιτικές δραστηριότητε. Όχι μόνο στις χώρες μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πνευματική και πολιτική διάβια δέχτηκα λοιπόν αυτή την πρόσκλησή σας. Με τον πρόεδρο Λαμασούρ Είχαμε υπόψη μας και θα παραμείνω στα πλαίσια των σκέψεών του ότι τα λίγα λεπτά που ακολουθούν θα μπορούσα να τα αφιερώσω σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία των αρχικών πρωτοβουλειών των αρχικών ημερών του φορολογικού συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η οπτική γωνία που θα ακολουθήσω είναι η πολιτική. Πώς προσπαθήσαμε με κάποια επιτυχία, περιορισμένη βέβαια, να αμφισίσουμε ζωή και δύναμη ίσως στον δυσχερέστερο όλων των τομέων της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ίσχυε τότε και όπως ισχύει άλλωστε και τώρα, η φορολόγηση βρίσκεται παγιωμένη στο βασίλειο της ομοφωνίας. Είναι πολύ εύκολο κάθε κράτος μέλος να θέσει τροχοπέδι στην πορεία των προσπαθειών. το πρόβλημα της ομοφωνίας εξακολουθεί να υπάρχει. Και κάποια θέματα έχουν γίνει πιο επιτακτικά και πιο κατεπήγοντα. Ίσως λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κάποιους τομείς που περικλείονται από το, τα ισχυρά τείχη της ε, ομοφωνίας. Όταν ο πρόεδρος Σαντέρ το 1995 με ανέθεσε μαζί με την ενιαία αγορά και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη φορολογική πολιτική, όλα τα φορολογικά μέτρα ήταν μπλοκαρισμένα ουσιαστικά. Ήταν πολύ φιλόδοξη η αρχική γραμμή, αλλά τελικά τα αποτελέσματα ελάχιστα. Θεωρήσαμε τότε ότι ίσως θα χρειαζόταν μια νέα στρατηγική. Δηλαδή, να μειώναμε το επίπεδο των στόχων μας, να έχουμε πιο μετριοπαθείς στόχους που θα ανακοινώναμε, ταυτόχρονα να γίνει όλο και πιο δύσκολο και πιο ενοχλητικό για τους υπουργούς οικονομικών να αρνούνται να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα ζητήματα. Πώς αντιμετωπίσαμε λοιπόν το θέμα. Υπήρχε ένα τμήμα της στρατηγικής το οποίο μας έδινε κάποια, κάποια άνεση, μας καθησύχαζε και κάποια άλλο που μας έφερε σε δύσκολη θέση. Το καλό κομμάτι ήταν ότι δεν τους λέγαμε ότι είμαστε εδώ για να απαλλαγούμε από την φορολογική σας κυριαρχία. Όχι. Επιχειρηματολογήσαμε χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που χρησιμοποίησαμε και για την νομισματική κυριαρχία πριν από κάποια χρόνια. Ότι υπήρχε μια επίφαση κυριαρχίας που διεφύλασαν, διότι κανείς δεν μπορούσε να την ασκήσει μεμονωμένα την κυριαρχία. Και αυτή η φορολογική κυριαρχία χανόταν καθημερινά λόγω των αγορών, λόγω της αυξανόμενης ολοκληρώσεως των ευρωπαϊκών αγορών. Ίσως θα ήταν επικοδομητικό για τη συνοχή της ενιαίας αγοράς, αλλά και κάτι που θα βοηθούσε και τα διάφορα Υπουργεία Οικονομικών και τα Ταμεία των Κρατών Μελών, αν υπήρχε μεγαλύτερο συντονισμός. Χαμηλώσαμε το λάβαρο λοιπόν της εναρμονίσεως και ψώσαμε το πιο παθές λάβαρο του συντονισμού. Σημειολογικό ίσως, αλλά λιγότερο απειλητικό, πιο καθησυχαστικό σαν μέτρο. Όμως, παρόλα αυτά, ακόμα και με μικρότερες φιλοδοξίες που ανακοινώθηκαν, οι Υπουργοί Οικονομικών, που ήταν μόνο 15 τότε, αρνήθηκαν να ασχοληθούν με ένα δύσκολο θέμα και να το εξετάσουν σοβαρά. Οπότε χρησιμοποίησαμε και την αρνητική πλευρά της στρατηγικής, αυτή που έφερε τους υπουργούς οικονομικών σε δύσκολη θέση. Πώς μπορούσαμε να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, τους πολιτικούς. Πώς θα μπορούσαμε να τους φέρουμε σε δύσκολη αν συνεχώς ειρνούντο να συνεργαστούν για φορολογικό συντονισμό. Η πραγματικότητα μας το έδειξε και το χρησιμοποίησαμε εμείς. Ποιο? Έναν κόμβο πάρα πολύ ενοχλητικό στο όλο θέμα. Ήδη τότε, παρόλο που ήταν 10 χρόνια πριν τη μεγάλη κρίση του 2007 και των επομένων ετών, υπήρχε ένα αυξανόμενο πρόβλημα ανεργίας και ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. Ήδη τότε ήταν σαφές ότι κάθε χρόνο λόγω ελλείψης φορολογικού συντονισμού υπήρχε μια αλλαγή όσον αφορά την δομή των φορολογικών εσόδων στην Ευρώπη και στα κάτι μέλη που ευνοούσε περισσότερο τους πιο κινητούς φορολογουμένους όπως το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις εις βάρος των λιγότερο κινητών φορολογικών βάσεων, κυρίως εργατικό δυναμικό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό πιο συγκεκριμένα. Όχι τους μεγάλους επαγγελματίες της Φόρμουλα 1 και τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να μετακινούνται εύκολα φορολογικά, αλλά μιλώ τώρα για τους ανειδίκευτους εργάτες, Αν το κόστος χρήσεως της πιο, του ε, δυναμικού που υπάρχει χρησιμοποιείς τα εργατικά χέρια περισσότερο και τους άλλους ε, παράγοντες παραγωγής τους μειώνεις μέσω της φορολογίας, αυτό δεν αντιμετωπίζει την ανεργία, αντιθέτως μάλιστα. Αυτό ήταν κάτι που ήταν πολύ ενοχλητικό κοινωνικά. Τους έφεραν σε δύσκολη θέση, τους Υπουργούς Οικονομικών. Διότι αρχή κρατών κυβερνήσεων και κρατών και υπουργοί οικονομικών δεν μπορούσαν να συνεχίσουν έτσι, ατιμωρητοί, να λένε ότι πολεμούν υπέρ της απασχόλησης και να αρνούνται να ε, αντιμετωπίσουν το θέμα του, της φορολογίας. Θα έλεγε κανείς ότι αισθάνονται πιο άνετα βρίσκονται σε, λιγότερη, σε μικρότερη θέση ε, όσον αφορά το ότι δεν κάνουν κάτι, αλλά έχουν και το όπλο της ε, ομοφωνίας. Μπορούσαν να το κάνουν, δεν το έκαναν όμως. Γιατί? Ξεκινήσαμε μια εκπαιδευτική και πολιτική διαδικασία. Ξεκίνησε κατόπιν ετήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί Ιταλικής Προεδρίας του 1996 σε ένα άτυπο συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ στη Βερόνα. Και λίγο αργότερα καταλήξαμε σε κάποια ευρωπαϊκά ε, πρότυπα την 1η Δεκεμβρίου του 1997. Ξεκίνησε η προσπάθεια με την Ιταλική Προεδρία και ολοκληρώθηκε επί Λουξεμβουριανής Προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 1997. Ετοιμάσαμε ένα πακέτο λοιπόν φορολογικού συντονισμού. απετελείτο από τρία στοιχεία. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Οι αρχές μιας μελλοντικής οδηγίας για την ε, φορολόγηση των αποταμιεύσεων, των καταθέσεων. Μία οδηγία όσον αφορά τη φορολόγηση των τόκων και των διαφόρων ε, δικαιωμάτων και ξεκίνησε ένας συντονισμός όσον αφορά τη φορολόγηση των εταιριών, διότι θεωρήσαμε ότι τουλάχιστον τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι έτοιμα να κινηθούν επί της βάσης εξετάσεως του θέματος από μότιμους φορείς και επί εθελοντικής αναθεωρήσεως των διαφόρων υφισταμένων φορολογικών μηχανισμών. Το πακέτο βεβαίως όπως σε πολλές πολιτικές διαπραγματεύσεις έχει ένα όφελος, ένα πλεονέκτημα αν παρουσιαστεί προσεκτικά και αν προωθηθεί προσεκτικά στις διαπραγματεύσεις. Ένα πακέτο μπορεί να εξαλείψει τις κόκκινες γραμμές. Πολύ συχνά, κυρίως στην ευρωπαϊκή πολιτική, παραλύουμε λόγω της ιδέας ότι κάποια χώρα είτε είναι μεγάλη είτε μικρή έχει αυτές τις κόκκινες γραμμές. Έχω την άποψη, ίσως να είμαι υπερβολικά αισιόδοξο, ότι οι κόκκινες γραμμές δεν υπάρχουν. Διότι πάντα μπορεί να βρει κανείς συνθήκες, μπορεί να βρει κανείς συνθήκες υπό τις οποίες εκείνος που προασπίζεται μια κόκκινη γραμμή μπορεί να αλλάξει τη θέση της κόκκινης γραμμής ή να μην θεωρεί πλέον ότι είναι τόσο ζωτικό το συμφέρον που υπερασπίζεται βάσει τη κόκκινη γραμμή. Βέβαια, θα πρέπει να μπουν θέματα σε πακέτο, τόσο ώστε κάποια στοιχεία του πακέτου να είναι ελκυστικότερα σε κάποιους και άλλα στοιχεία ελκυστικότερα σε άλλους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα μικρό παράδειγμα όσον αφορά τον μικρό κόσμο της Benelux, που είναι ένας πλούσιος κόσμος και περίπλοκος. Το Βέλγιο ήθελε τότε διακαώς να εισθεσπίσει μια οδηγία για την φορολόγηση των καταθέσεων διότι δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα ότι πλούσιοι Βέλγοι, οδοντίατροι, ίσως και κάποιες άλλες κατηγορίες, ε, κατέθεταν τις οικονομίες του στο Λουξεμβούργο και έτσι ε, πέτυχε έναν φοροδιαφυγή. Το Λουξεμβούργο δεν διαμαρτυρόταν καθόλου για την όλη κατάσταση, αλλά διαμαρτυρόταν πολύ χειρά λέγοντας ότι το Βέλγιο προσέφερε πολύ θετική φορολογική αντιμετώπιση στις πολυεθνικές που είχαν την έδρα τους στο Βέλγιο. Αυτές είναι μόνο δύο χώρες από τις 15 ε, που είχαμε τότε αλλά αρχίζετε να βλέπετε ότι αν βάλετε σε ένα πακέτο την οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και κάποιες αρχές για την φορολόγηση των επιχειρήσεων ταυτόχρονα, μπορεί να προσελκύσεις ακόμα και χώρες ε, οι οποίες δεν θα είχαν προσελκυστεί από αυτά τα μέτρα. Ακολουθήσαμε την προσέγγιση του πακέτου λοιπόν Και υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφέρω που ίσως να ενδιαφέρει και κάποιες καινούριες σημερινές ε, πρωτοβουλίες κατά το παρελθόν. Όλα τα φορολογικά θέματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπιζόταν σε τεχνικά επίπεδα. Γενικοί διευθυντές για την άμεση φορολόγηση, γενικοί διευθυντές για έμεση φορολογία Φερρυπίν, τα συζητούσαν. Αυτή είναι η καλύτερη συνταγή, ούτω ώστε να έχεις μεγάλες γνώσεις εκείνο που ασχολούνται με τα θέματα, αλλά και να μην αλλάζει και τίποτα ουσιαστικά. Ποια ήταν η ιδέα. Μια μετριοπαθής ιδέα, να αλλάξουμε κάπως τα πράγματα, έπρεπε να εμπλακούν περισσότερο Υπουργοί Οικονομικών. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια ομάδα φορολογικής πολιτικής υπό την Προεδρία και το υπογραμμίζω αυτό και έντονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι από το Συμβούλιο όχι από την χώρα που είχε την Προεδρία, από τον ε, Επίτροπο Αρμόδιο για την ε, φορολόγηση. Και κάθε Υπουργός Οικονομικός εκαλείτο να διορίσει έναν ε, προσωπικό εκπρόσωπό του και είχαμε μεταβλητή γεωμετρία. Και βεβαίω και ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας. Σε άλλε περιπτώσεις θυμούμε την περίπτωση του Βελγίου. Ήταν ο υπουργό Οικονομικών τη εποχή εκείνη στην βελγική κυβέρνηση που όρισε έναν Βέλγο βουλευτή, ε, Βέλγο ευρωβουλευτή ε, υψηλών ικανοτήτων και που έχερε τις απολύτω εμπιστοσύνη του Υπουργού και ούτω καθεξής. Και διεξήχθησαν ε, τακτικές συναντήσεις του οργάνου αυτού που δεν θα είχαν γίνει με τους Υπουργούς Οικονομικών. Σαφώς όμως επρόκειτο για ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν σε κάποια χρονική στιγμή εφόσον είχαν πιστεί να προτείνουν στους υπουργούς τους να αλλάξουν ορισμένα πράγματα από αυτά που θα είχε προτείνει αφεύκτος η ηγεσία του Υπουργείου του των Οικονομικών. Έτσι λοιπόν, την 1η Δεκεμβρίου του 1997 ε, προέκυψε ομόφωνη συμφωνία στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ μεταξύ των 15 τότε χωρών μελών. Όχι βεβαίως ότι όλες οι προσωπικότητες εκείνες υπεχώρησαν, δηλαδή ότι ε, συμφώνησαν όλοι εύκολα. Είχαμε για παράδειγμα τον Gordon Brown και άλλους οι οποίοι συνέβαλαν σε μια ζωηρότατη συζήτηση. Πάντως εδώ θα ήθελα να σημειώσω διότι αυτό συνδέεται κύριε Πρόεδρε και με μία από τις απαρχές της δικής σας ειδική Επιτροπής Ποιος ήταν ο πρόεδρος στο δεύτερο μισό του 1997, όχι στην προεδρία του Tax Policy Group, ήταν ο Επίτροπος, αλλά στην πραγματική προεδρία του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ ήταν υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου και το όνομά του ήταν και πρωθυπουργός. Το όνομά του λοιπόν Jean-Claude Juncker. Σημειώνω λοιπόν ότι η δέσμη μέτρων για τα φορολογικά που εγκρίθηκε στην πρώτη η του 1997 και που γενικώ θεωρείται ως το βασικό θεμέλιο για τις ε, μετέπειτα εξελίξεις στον συντονισμό για τα φορολογικά αλλά και για τις ρυθμίσεις της Κομισιόν για τις κρατικές επιδοτήσεις αλλά και για τις λεγόμενες tax rulings ήταν κυρίως αποτέλεσμα των διαπραγματευτικών ικανοτήτων και της αποφασιστικότητας του σημερινού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το προηγούμενο Βέβαια όλοι σας λίγο πολύ υπήρξατε Υπουργοί Οικονομικών στις χώρες σας αλλά αν εξετάσω την στάση του κυρίου Γιούνκερ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιρρώνει αυτά που λέω τώρα. Και γι' αυτό είμαι πλήρης ελπιδός ότι η Επιτροπή Γιούνκερ θα δράσει με αποφασιστικότητα στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Και έχω δει άλλωστε τις ακροάσεις ε, στις οποίες προσκαλέσατε την κυρία Βέστερ και τον κύριο Μοσκοβισή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ έχω συνομιλήσει μαζί τους και μου φαίνονται το ίδιο αποφασιστικοί όπως και ο πρόεδρος σας για να επιτελέσουν πρόοδο. Ας ε, μου επιτρέψετε τώρα να ολοκληρώσω σύντομα στην βάση του ψηφίσματος του Συμβουλίου και του κώδικα διοντολογίας που είχαν εγκρίνει χώρες μέλη του Συμβουλίου. Μετά από αυτό ακολούθησαν άλλα βήματα και αυτό ήταν ένα θετικό spillover από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πήγε και σε άλλα όργανα. Και μάλιστα ήταν και πλευρό γιατί ο ΣΑ, αν εξετάσετε τις ημερομηνίε, έφτασε στον ορισμό της ε, επιβλαβούς, του επιβλαβούς μάλλον φορολογικού ανταγωνισμού λίγο μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό σε μια προσπάθεια να είναι όσο γίνεται πιο συνεκτικές οι στάσεις των οργάνων αυτών. Και άλλη μια συνέπεια ήταν ότι υπήρχε πλέον η βάση πάνω στην οποία να βασιστεί μια μακρά και δύσκολη πορεία και συνεργασία με άλλες μη μέλη χώρες. Και θυμούμε μια ημέρα του Ιουνίου του 1999, όπου ως Επίτροπος Αρμόδιος για τη Φορολογία πήγα μαζί με τον εκπρόσωπο της Γερμανικής τότε, τότε Προεδρίας στην Βέρνη για μια πρώτη, πρώτη, πρώτη επαφή με τον Ελβετό Υπουργό Οικονομικών για να συζητήσουμε φορολογικά θέματα. Και το ίδιο το απόγευμα είδαμε και τον Υπουργό του Λίχτενστάιν. Σε άλλα κατοπινότερα βήματα της ευρωπαϊκής μου πορείας. Βέβαια και οι Ιταλοί φορολογούμενοι δεν θα ξεχάσουν το 18 μήνο όπου ρύθμιζα τα φορολογικά τους θέματα, αλλά για τα επόμενα πέντε χρόνια όταν είχα την ευθύνη του ε, χαρτοφυλακίου για τον ανταγωνισμό εξετάσαμε προσεκτικά πώς οι κανόνες των κρατικών επιδοτήσεων μπορούσαν να εφαρμοστούν στην τυπολογία των δημοσιονομικών κρατικών επιδοτήσεων. Και όπως θα σας είπε και η Νίνα Αρμοδία Επίτροπος, ξεκινήσαμε μια δραστηριότητα η οποία ήταν συμπληρωματική με το έργο που διεξήγεται στο Συμβούλιο από τις χώρες μέλη. γιατί είχαμε τους μοχλούς της πολιτικής της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε και ελήφθησαν τελικώς 15 αρνητικές αποφάσεις. Πιο πρόσφατα, αλλά βέβαια πάλι εδώ και μια πενταετία, όταν ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, μου ζήτησε να του υποβάλω έκθεση για το μέλλον της ενίας αγοράς, Είχα εκεί περιλάβει και ένα κεφάλαιο για την φορολογική διάσταση της ενιαίας αγοράς και επιγράφεται συνεργασία για να διασωθεί η φορολογική κυριαρχία που φαίνεται σαν να είναι καταρχήν κάτι φιλικό προς τους Υπουργούς Οικονομικών. Και εγώ πρότεινα τότε εκεί ότι θα μπορούσε να γίνει μια επανεκκίνηση των προσπαθειών για να υπάρξει μια εναρμονισμένη φορολογική βάση για τον εταιρικό φόρο που έχει βεβαίως το μέγα διανοητικό πλεονέκτημα ότι θα πρέπει να είναι κανείς υπέρ της εναρμόνισης της φορολογικής βάσης και εάν θέλετε τον εναρμονισμό των συντελεστών, αλλά και αν τον μισείτε τον εναρμονισμό των συντελεστών. Διότι αν αγαπάτε, αν σας αρέσει ο εναρμονισμό των συντελεστών, θα, δεν θα έχει νόημα να εναρμονίσετε πράγματα τα οποία θα εφαρμόζονται σε διαφορετικά πράγματα και όχι σε κάτι το οποίο υπάγεται σε ένα κοινό ορισμό. Εάν δεν απεχθάνεστε το, τον εναρμονισμό των φορολογικών συντελεστών, διότι σας αρέσει ο φορολογικός ανταγωνισμός, θα θέλετε τότε οι χώρες μέλη να παίξουν το παιχνίδι του φορολογικού ανταγωνισμού σε μια διαφανή βάση και οι εταιρείε να μπορούν να γνωρίζουν ποια χώρα προσφέρει τον πιο ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή. Πάλι εκεί χρειάζεται ένας κοινό ορισμός του εταιρικού κέρδους. Και στην έκθεσή μου προς τον πρόεδρο Μπαρόσο είχα προτείνει ότι ίσως μια tax policy group θα ήταν χρήσιμο να ιδρυθεί και είδα στα όσα παρουσίασε ο Επίτροπος Μοσκοβισή στην Επιτροπή σας, ο οποίος έχει λάβει τώρα αυτή τη θέση, είδα λοιπόν ότι είναι λίαν αποφασισμένος όσον αφορά την ε, φορολογία των επιχειρήσεων. Και το τελευταίο βήμα είναι ένα βήμα το οποίο εσείς κύριε Πρόεδρε και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους οι οποίοι εμπλέκονται εμπλεκόμεθα σε ένα εγχείρημα Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για κάτι το οποίο δεν είναι κάθε αυτό φορολογία αλλά είναι οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πιστεύω λοιπόν ότι οι, οι συνέργειες και διανοητικά και τεχνικά και πολιτικά ανάμεσα στον χώρο του χειρισμού των εθνικών φορολογικών πολιτικών. Η έκταση και οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων της διαμορφώσεώς τους, αλλά και η μελλοντική διαμόρφωση του κοινοτικού προϋπολογισμού, όλα αυτά θα συναποτελέσουν ένα αντικείμενο πολλά υποσχόμενο. Σας ευχαριστώ για την μεγάλη υπομονή σας και την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. για την πολύ καλοδεχούμενη αυτή υπενθύμηση του παρελθόντος. Πολύ ποιοτικέ οι απόψεις, πολύ ποιοτική και η σύνθεση, μας εντυπωσιάσατε. Να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές για να κάνουν τις ερωτήσεις τους και αφού απαντήσει ο κύριος Μόντι θα δώσω στη συνέχεια το λόγο στους εκπροσώπους των ομάδων. Η Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Γερουσιαστά Μόντι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Ε, άκρος σημαντικά και όσα κάνατε και όσα προτείνατε και όλες σας οι σκέψεις για αυτά τα θέματα είναι σημαντικές και ελπίζω να παρακολουθείτε το έργο της Επιτροπής μας, της δικής αυτής Επιτροπής, για να μπορέσουμε και εμείς να αποφεληθούμε από τη σοφία σας και την εμπειρία σας. Ε, έρχομαι στην ουσία του θέματος. Στις 5 Μαΐου συνομιλήσαμε με τον κύριο Νόλς και αποκόμισαμε την εντύπωση, για να το πω ομά, ότι μετά από την αρχική αυτή όθηση η ομάδα για το... ομάδα επαφή για τον κώδικα ε, έχασε το δυναμισμό τη, ε, για να το θέσω έτσι, και είναι σαφέ ότι δεν παρέχει τι απαντήσει, τι ευρωπαϊκέ απαντήσει που χρειαζόμαστε σήμερα. Αυτό που ξεκίνησε πριν ε, από 4-5 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία άκρος ήπια συμφωνία κυρίων που δεν έχει καμία δύναμη επιβολής και με τη σημερινή κατάσταση αλλά και πολύ πριν ε, τα Lux Leaks, Offshore Leaks, ε, Swiss Leaks κτλ. κατάσταση είναι πολύ δραματική και πολύ άδικη για τους πολίτες. Άρα δεν μπορούμε να δεχθούμε πλέον μια τέτοια τόσο ήπια προσέγγιση και πάνω από όλα αυτά, αυτό που πολύ ορθά εσείς θεωρείτε ένα μεγάλο πρόβλημα για την εσωτερική αγορά, δηλαδή τα διαφορετικά επέμφωλικών συντελεστών, αυτό πλέον έγινε και εθνικό πρόβλημα, διότι στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα έχουμε την οικονομική διακυβέρνηση, τις τρόικες, άρα ε, κάποια κράτη-μέλη ελέγχουν τον προπολογισμό άλλων κράτων, κρατών Κάτι που δεν υπήρχε πριν. Και από την άλλη πλευρά, κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη σαφώς ακολουθούν άκρος ε, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Αυτό το επιβεβαιώσαμε με τις επισκέψεις μας σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, κάτω χώρες, Ελβετία. Και ναι, μεν έχουμε καλά επιχειρήματα, να προβάλλουμε, όπως είπατε, όχι μόνο στο καταστατικό επίπεδο, στο επίπεδο των φόρων, αλλά σε ό,τι αφορά και τη διάβρωση ε, των ε, εισοδημάτων ή των ε, φοροϊκών εσόδων. Έχουμε δίκτυα διμερών συμφωνιών, έχουμε φορολοτεχνικούς, συμβούλους και αυτά τα φαινόμενα ε, οδηγούν σε μια πραγματική ζούγκλα ε, πολύ επιθετικές ε, φορολογικές πρακτικές, άρα επίγει, είναι κατεπήγον μάλιστα, ε, να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση για το πρόβλημα αυτό. Έχουμε κάποια στοιχεία στην ημερήσια διάταξη. Μιλήσατε για το CCTB, την ενωπημένη δηλαδή βάση, τι φορολόγηση, αυτές τις αλλαγές αποφάσεις τύπου tax ruling. Όλα αυτά πρέπει να τα προωθήσουμε στη βάση των προτάσεων της Κομισιόν και από ό,τι ανακαλύψαμε δεν έχει υπάρξει καμία ανταλλαγή πληροφόρων μεταξύ των διοικήσεων μέχρι τώρα. Ελάχιστες και πολύ συγκεκριμένες οι εξαιρέσεις. Και το επιχείρημα είναι, μα δεν ζήτησε κανεί αυτέ τι πληροφορίε. Ναι, φυσικά είναι απόρριτο και δύσκολα μπορεί κανεί να ρωτήσει συγκεκριμένα. Επειδή όμω κανεί δεν ρώτησε, δεν δώσαμε τι πληροφορίε, λένε. Και εμεί δεν τι ζητήσαμε τι πληροφορίε γιατί δεν τι χρειαζόμαστε. Άρα αυτό οδηγεί ε, στην απουσία φορολόγησης και οδηγούνται τα χρήματα σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως έλεγα λοιπόν έχουμε αυτή την ε, βάση, την ενωπημένη βάση, έχουμε την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα, την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ίσως και άλλα στοιχεία, τα ξέρετε. Όλα αυτά τα έχουμε, αλλά εσείς τι μας συμβουλεύετε. Τι στρατηγική μπορούμε να υιοθετήσουμε για να αντιμετωπίσουμε Κάτι το οποίο πραγματικά γίνεται αφόρητο από πολιτικής πλευράς και έρχομαι στο τελευταίο αίτημά μου ε, και στο τελευταίο μου σχόλιο. Δύο επιχειρήματα πολιτικού χαρακτήρα. Όταν αντιμετωπίζουμε τα κράτη-μέλη, τους υπουργούς οικονομικών και τους αναφέρουμε την παράβαση βασικών κανόνων ανταγωνισμού και ηθικών αρχών ή αρχών διοντολογίας, μας απαντούν είμαστε πολύ μικροί ως χώρα, όπως λέει το Λουξεμβούργο το Βέλγιο για παράδειγμα. Είμαστε στην περιφέρεια, άλλοι, όπως ε, λένε οι κάτω η κυρλανδια η Ελβετία. Αυτά οι είναι τα επιχειρήματα. Άρα, ε, τι να πω, από πολιτικής πλευράς περίεργα τα επιχειρήματα. Μήπως πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά τα θέματα. Και ένα τελευταίο επιχείρημα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε γιατί σε διεθνέ επίπεδο έχουμε πάρα πολύ άγριο ανταγωνισμό και ανταγωνισμό τους φορολογικού παραδείσους με τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κόνγκ και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλο. Και ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε πλέον την Ευρώπη αλλά όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι ένα είδος ε, σύνθεσης ε, των μέχρι τώρα εντυπώσεων που έχουμε αποκομίσει. Με βάση την εμπειρία σας, ποιος είναι ο δρόμος αν θέλουμε να αναστρέψουμε γρήγορα την κατάσταση αυτή, γιατί όπως είπα γίνεται αφόρητη και από πολιτικής και από οικονομικής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ Ελίζα. Στο μεταξύ ήρθε και ο συνεισηγητής Μικάλ Τόιρερ, στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γερουστά, Γερουσιαστά, ευχαριστώ για την έλευσή σας εδώ. Στην ομιλία σας θυμήσατε την σύναψη του πρώτου τότε κειμένου υπό την ηγεσία του τότε Πρωθυπουργού Jean-Claude Juncker. Θα ε, τονίσω και εγώ τα όσα είπε η συνεισηγήτριά μου κυρία Φερέιρα και τις επισκέψεις σε χώρες μέλη όπως η Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και κάτω χώρες που υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες και αυτά που ακούσαμε εκεί είναι ότι υπάρχει αύξουσα υποστήριξη για, την προτινό, για τις προτινόμενες μάλλον νομοθετικές ρυθμίσεις ιδίως στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κυβερνήσεις και κοινοβούλια των χωρών αυτών αναμένουν αναθεωρημένες προτάσεις για το CCCTB επίσης για διάφορα δικαιώματα, royalties κλπ. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν εξετάσετε τα πακέτα αυτά, τα μέτρα αυτά, θεωρείτε ότι επαρκούν για να διασφαλίσουν μια, έναν έντιμο φορολογικό ανταγωνισμό, διότι ακούσαμε και σε ορισμένα κοινοβούλια και από ορισμένου εμπειρογνώμονες να ισχυρίζονται ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι σημαντικός, ίσως και αναγκαίος για μικρές ιδίως χώρες για να μπορέσουν αυτές να αντιμετωπίσουν τις δημοσιονομικές τους αναγκαιότητες. Αλλιώς, μας είπαν ορισμένοι βουλευτές ή και εμπειρογνώμονες, ότι χωρίς τον φορολογικό ανταγωνισμό δεν θα είναι δυνατόν μικρές ή περιφερειακές χώρες να προσελκύσουν ε, επιχειρήσεις. Και σήμερα, μάλιστα, στην εφημερίδα Financial Times ακούμε ότι μία από τις έξι διεθνείς ε, εταιρείε έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους ή έχουν εκεί θηγατρική πλήρωση ιδιοκτησία τους. Και αυτό που ήταν ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιρλανδία και στην Ολλανδία, στις επισκέψεις που κάναμε δηλαδή, ορισμένοι μας είπαν, μάλλον ορισμένοι εκεί κατηγορούν την άλλη χώρα ή ακόμη και το αμερικανικό φορολογικό σύστημα για, τα, για όλα τα φτεξίματα. Εμπειρογνώμονες στην Ιρλανδία μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται κατά εσφαλμένου στόχου, γιατί το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το δικό τους, ας πούμε, ελλανδικό ή Ολλανδικό φορολογικά συστήματα, αλλά το Αμερικανικό των Ενωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να σχολιάσετε στην βάση της πείρας σας ε, το θέμα αυτό. Μάθαμε επίσης, για παράδειγμα, ότι το Double Irish δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα σε συνδυασμό με το Dutch sandwich. Και μόνο έτσι γίνεται τελικός φορολογικός παράδεισος. Ένας Ολλανδός βουλευτής μας είπε ότι η Ολλανδία δεν είναι φορολογικός παράδεισος. Είναι πύλη για φορολογικούς παραδείσους, για κάποιον που δεν είναι για κάποιον που δεν έχει μητρική γλώσσα, γλώσσα τα αγγλικά, οι λέξεις tax haven και tax heaven μοιάζουν πάρα πολύ. Πάντως η ε, Κομισιόν προτείνει έναν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, τουλάχιστον τον μελετά όταν συζητεί για μια πρόταση CCCTB. Θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλλει και ένας ανώτατος φορολογικός συντελεστής έτσι ώστε να μειωθούν τα ποσοστά φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Η τελευταία, η τελευταία ερώτηση που σας απευθύνω μετά από την εμπειρία σας στην Επιτροπή ο ΦΠΑ νομίζουμε ότι έχει λύσει τα προβλήματά του. Όμως οι αποκαλύψεις των διαρροών του Λουξεμβουργού μας δείχνουν, αν εξετάσουμε την περίπτωση του Amazon, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι με ναι, τζίρο παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ που προέρχονται από τη Γερμανία, ο ΦΠΑ που ε, πληρώνει στο Λουξεμβουργό είναι της τάξης των 40-50 εκατομμυρίων. Είναι πάρα πολύ χαμηλός ο συντελεστή αυτός. Και ο κόσμος στη Γερμανία εξακολουθεί να έχει την ψευδέστηση ότι αν αγοράσει ένα βιβλίο στο Amazon πληρώνει ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ όμως επιστρέφεται όταν ο τζίρος φορολογείται στο Λουξεμβούργο. Ελπίζουμε ότι με τις νέες ρυθμίσεις αυτό θα πάψει για το μέλλον. Αλλά ποια είναι η δική σας εντύπωση. Θεωρείτε ότι αυτό το αποτέλεσμα μόχλευσης, αυτό είχε προβλεφθεί όταν συζητούσατε με τις χώρες μέλη την επιβολή του πρώτου φορολογικού πακέτου ή δεν είχε προβληθεί κάτι σχετικό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γερουσιαστά. Thank you very much to both rapporteurs. Ευχαριστώ και τους δύο που πήραν το λόγο και τους δύο συγγητές. Ελπίζω να μην υπάρχει μια τραγική παρεξήγηση. Δεν είμαι ειδικό για τα φορολογικά. και η ομορφιά της θέσης μου ως Επιτρόπου Υπευθύνου για τα φορολογικά ήταν ακριβώς αυτή ότι μπορούσα να βασίζομαι σε εμπειρογνώμονες αλλά μπορούσα να διαβλέπω νέες προσεγγίσεις. Το λέω αυτό ιδιαίτερα όσον αφορά αυτά που μου είπε ο κ. Τόιραρ. Ακριβέστατες ήταν οι ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω την τελευταία για τα φαινόμενα μόχλευσης, τα αποτελέσματα μόχλευσης. Δεν θυμάμαι να το είχαμε συζητήσει τότε αυτό. Εδώ και 18 χρόνια δηλαδή. 18 χρόνια. Και αν κάποιος τότε μου είχε αναφέρει μετά το τέλος των πολύ μακρών εξαντλητικών συνεδριάσεων για το Ολλανδικό σάντουιτς με Ιρλανδικές νότες, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, τότε θα το είχα δεχτεί. Ελάχιστος φορολογικός συντελεστής. Δεν είναι τόσο εύκολο να καθορίσουμε τι είναι δίκαιο ποιος είναι ο δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός. Στη φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι αξιοσημείωτο το ότι ο δοντολογικός μας κώδικας και μετά αυτός του ΩΣΑ έδιναν ακριβείς ενδείξεις περί του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού έναντι του αθέμητου και αυτό το επεξεργαζόταν η αρμόδια ομάδα. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι από τον δεντολογικό κώδικα. Δεν νομίζω ότι τροποποιήθηκε εν μεταξύ. Τα φορολογικά μέτρα που καλύπτονται τον κώδικα καλύπτουν νόμους και κανονισμούς σε διοικητικό επίπεδο και πρακτικές και εντός του πεδίου που αναφέρεται στην παράγραφο α τα φορολογικά μέτρα τα οποία προβλέπουν σημαντικά επίπεδο φορολόγηση, συμπεριλαμβανομένου μηδενικού επίπεδου φορολόγηση και εκείνα τα ποσοστά που συνήθω ισχύουν στον λόγο κάτω μέλο θα πρέπει να θεωρούνται ως ενδεχομένως επιβλαβή επίπεδα και καλύπτονται συνεπώς από τον κώδικα αυτό. Τέτοιο επίπεδο φορολόγησης μπορεί να λειτουργήσει βάσει του ονομαστικού ποσοστού φορολόγησης ή άλλων σχετικών παραγόντων και παρατίθεται ένας κατάλογος μετά πέντε παραγόντων για τους οποίους λέγει ότι όταν γίνεται αξιολόγηση κατά πόσο τέτοια μέτρα είναι επιβλαβή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων κλπ. κλπ, κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ακόμα χρήσιμο να κρατήσουμε αυτή την έννοια του θεμητού και του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού αν μη τι άλλο διότι αν αυτό καταργηθεί και γίνει μία επίθεση επί όλου του φορολογικού ανταγωνισμού τότε θα υπάρχει πολύ πιο μεγάλη αντίσταση σε αυτό και θα υπάρχει λαϊκή επίκριση που θα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μεταξύ άλλων, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων λέει ότι έχει το καθήκον να εμποδίζει και να καταργεί τα καρτέλ, τώρα βοηθά ένα καρτέλ κρατών μελών να εκμεταλλεύεται τους φορολογούμενους. Θα υποθούν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό, σε ένα φιλελεύθερο πνεύμα, κύριε Τόιρερ, πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός και να μην καταδικάζει κάθε φορολογικό ανταγωνισμό διότι είναι αληθές ότι σε διεθνές επίπεδο η Ευρώπη κατά μέσο όρο επιβάλλει μεγαλύτερη φορολογία από τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, διότι έχουμε και προτιθέμεθα να εξακολουθούμε να έχουμε και κάποιο κοινωνικό μοντέλο που δεν έχουν άλλες χώρες. Η ιδέα λοιπόν ότι κάποιος ανταγωνισμός μπορεί να βοηθά μπορεί να υποχρεώσει χώρες να ελέγξουν τα δημοσιονομικά τους αυτό είναι κάτι που εμπεριέχει καλά στοιχεία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός δεν λαμβάνει χώρα ουδετέρως αλλά στρεβλώνει την όλη κατάσταση διότι ευνοεί την κινητή φορολογική βάση ε, εις βάρος της λιγότερο κινητής φορολογικής βάσεως. Κατά την άποψή μου λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Άκουσα επίσης όπως και εσείς το άλλο επιχειρήμα για τα περιφερειακά κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη της περιφερείας. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι, αυτό το επιχείρημα, διότι αν κάποιοι Κοιτάξτε, το ότι είναι μια χώρα μικρή δεν απαραίτητα μειονέκτημα. Σίγουρα κάποια γεωγραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν μειονέκτημα. Παραδείγματο χάρη, μια χώρα που έχει χιλιάδες νησιά που πιστεύω ότι δεν περνά κρίση λόγω των υπέροχων νησιών της, παρόλα αυτά έχει το πρόβλημα των πολλών νησιών, αυτό καλύπτεται από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και υπάρχουν δυνατότητες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέσω κρατικών ενισχύσεων. Και το ότι είναι μια χώρα περιφερειακή, κατά την άποψή μου, δεν είναι πραγματικά μια δικαιολογία θεμητή για την έγκριση μέτρων που επιτρέπουν επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισμό. Κάτι που συνδέεται με αυτό που μας είπε η κυρία Φερέιρα δεν γνώριζα την τη θέση του κ. Νόλτς. Είναι και πρόεδρος της ομάδας ε, για τη διοντολογική συμπεριφορά και λέει ότι είναι λιγότερο δυναμική αυτή η φάση. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος. Αν είναι κανείς αισιόδοξο μπορεί να πει ότι αν εξαλειφθεί ο επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός για τις επιχειρήσεις δρέπονται κάποιοι καρποί και ίσως στις αρχικές φάσεις. Οπότε δεν επιτυχάνονται ακριβώς οι στόχοι που θέλουμε. Εξαρτάται και κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα να εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα. Στην αρχική ενσάρκωση της ομάδας του δεντολογικής συμπεριφοράς στο Συμβούλιο παρόλο που είναι ουδέτερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τους διορισμούς που πραγματοποιούνται από τα κάτι μέλη καλωσόρισα την ιδέα το ότι η Βρετανία και ο Υπουργός Οικονομικών Gordon Brown τότε θέλαν να προτείνουν έναν ε, υφυπουργό οικονομικών, έναν πολιτικό εκπρόσωπο του εργατικού κόμματος που προείδρευε της ομάδας και εκείνη ήταν εκπρόσωπος του Gordon Brown στην ομάδα μου. Είδα ότι ήταν ισχυρή, ήταν αποφασιστική. Και ότι θα υπήρχε εκπροσώπηση από την Βρετανία και θα προείδρευε τις ομάδες ήταν κάτι πολύ θετικό για μας. Η Βρετανίδα εκπρόσωπος προείδρευε. Ότι συμμετείχε και το Ηνωμένο Βασίλειο στο όλο εγχείρημα. Αυτό σήμαινε. Υπήρχε και άλλη μεγάλη χώρα, κάτω μέλος, που επίσης είχε πολύ καλό εκπρόσωπο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν υποστηρίζει που υποστήριζε προφανώς την όλη προσπάθεια. Ουδέτερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ με ικανοποίηση είδα ότι προχωρούν τα πράγματα. Δηλαδή είχαμε την Βρετανίδα η κυρία που προείδρευε της ομάδας. Τώρα είναι γενική διευθύντρια για τα φορολογικά. Ε, ε, ο και ο κύριος Νόλς είναι πάρα πολύ ικανός. Να σας δώσω κάποιες συμβουλές κλείνοντας. πώς να δώσουμε όθηση στις πρωτοβουλίες και τα βήματα. Νομίζω ότι προς τα εκεί κινείστε. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Όταν η τελική σας έκθεση θα εκπονηθεί, νομίζω ότι θα είναι πολύ επικοδομητικό αν με αντικειμενική δημόσια παρουσίαση μπορείτε να προσελκύσετε την προσοχή των Υπουργών Οικονομικών και των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων προς αυτή την έκθεση. Και αν θα μπορούσατε σε κάποια φάση, αλλά σύντομα, να μπείτε στο δρόμο της δημιουργίας μια πιο πραγματικής διακυβέρνησης για την οικονομική και νομισματική ένωση. Και να ισχυριστείτε, όπως θα έκανα εγώ, ότι η φορολογική ένωση δεν αφορά μόνο τελειότερους κανόνες για πειθαρχία και για εφαρμογή και συγκράτηση των εθνικών ελλημάτων και χρεών, αλλά πρόκειται και περί της δομής της φορολόγησης των δημοσιονομικών στην Ευρώπη. Η δομή αυτών να οδηγεί σε πιο εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, που είναι οικοδομικός λίθος της οικονομικής ε, και νομισματικής ενώσεως. Όσο κλιμακώνει κανείς, αυξάνει το πολιτικό επίπεδο και το έργο του το ανυψώνει στο σωστό πλαίσιο, δημιουργείται ορμή και όθηση στην όλη προσπάθεια και διατηρείται αυτή η ορμή. Ευχαριστώ κύριε Γερουσιαστά. Θα δώσω το λόγο τώρα στον καθένα παρακαλώ να μιλήσει για δύο λεπτά παρακαλώ. Στα μέλη της ομάδας θα δώσω το λόγο, στους εκπροσώπους των ομάδων. Και εισπάξει μια γενική απάντηση στις ερωτήσεις. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μπορκαρτ Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, έλεγα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γεροσιαστά, είναι μεγάλη χαρά μας, βεβαίως, που είστε σήμερα εδώ κοντά μας, διαθέσιμος για τα λεγεία απόψεων, ως πρώην Επίτροπος Φορολογίας βρεθήκατε σε ένα σημείο τομής που για τη δική μα Επιτροπή βεβαίως έχει πάρα πολύ κρίσιμη σημασία. Θα ήθελα να έρθω σε ένα θέμα σχετικά με την φορολογική κυριαρχία των χωρών μελών πάντοτε πρεσβεύσατε ρεαλιστικές θέσεις και τονίσατε την ανάγκη Εξέτασα παλαιότερες δηλώσεις σας το 1997 βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Είχατε αναλάβει πρωτοβουλία κατά επιβλαβών φορολογικών πρακτικών. Και στην έκθεση Μόντι, που φέρει το όνομά σας, δηλαδή του 2010, περιλαμβάνονται προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές και ιδίως για την ενισχυμένη συνεργασία των χωρών μελών. Σας ερωτώ σήμερα, κατά την άποψή σας, ποιες πρόοδοι επετεύχθησαν έκτοτε. Κάποια πράγματα ήδη είπατε, ίσως όμως μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο. Και ιδίως με τα όσα γνωρίζετε σήμερα, τι θα θέλατε να είχατε προτείνει τότε, ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται ήδη εδώ και μια εικοσαετία με το θέμα. Τι λοιπόν θα κάνατε τότε διαφορετικά ή τι προτάσεις διαφορετικές θα κάνατε τότε. Δεύτερη ερώτηση. Πάλι κάτω από ένα πρίσμα ρεαλισμού ποιους στόχους μπορεί να βάλει ρεαλιστικούς η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις χώρες μέλη για να αντιμετωπίσει σε διεθνές επίπεδο την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Και όταν λέω διεθνές εννοώ παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ Μπορκχαρτ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο Πέτερ Σίμον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Μόντι για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Χαίρομαι που μπορώ να συνομιλήσω μαζί σας για το έργο που επιτελέσατε ως Επίτροπος για τα φορολογικά. Αναφέρομαι ιδίω σε μια δέσμη για το θέμα των ενισχύσεων το πακέτο Monty Cruz το οποίο ξεκίνησε μια πορεία στην Ευρώπη που λίγα χρόνια πριν θα ήταν αδύνατο να το διανοηθεί κανείς για τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών τους. Άλλαξαν λοιπόν πολλά δεδομένα στις χώρες μέλη. Η Κομισιόν εφήρμοσε, επέβαλε το δίκαιο ανταγωνισμού με το πακέτο Monte Cruz και έχει εξασφαλίσει διαφανείς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, λέγοντας ότι κοιτάξτε αυτό είναι συμβατό με δίκαιο ανταγωνισμού και αυτό δεν είναι. Μείνετε λοιπόν μέσα στο πλαίσιο των συμβατών. Ένα εκατοστό να ξεφύγετε, αμέσως θα υπάρξει προσφυγή για παράβαση της συνθήκης. αυτή είναι η τομή όπου οι χώρες μέλη, εφόσον εξετάσει κανείς σήμερα, έχουν τηρήσει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να εφαρμόσει το δίκαιο αυτό για τις ενισχύσεις, εγώ αυτό το βρίσκω πολύ ικανοποιητικό. Θεωρώ ότι θα είναι ορθή η προσέγγιση να μπορεί κανείς ανεπηρέαστος από τις χώρες μέλη να εξετάσει τις δυνατότητες που δίνουν οι συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση αυτές τις δυνατότητες να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλαίσιο που θα είναι δεσμευτικό για τις χώρες μέλη και αν είναι αρκετά φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να το πράξει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να την εμποδίσει. Από τη δική σας εμπειρία λοιπόν, από την εκπόνηση παρόμοιου πλαισίου, βεβαίω σε άλλε συνθήκε τότε, πώς μπορείτε να κρίνετε τώρα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό του δικαίου των ενισχύσεων για να θεσπίσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ανταγωνισμού έτσι ώστε να δεσμεύσει τις χώρες μέλη να τις βάλει σε ένα στενό κορσέ αν με επιτρέπετε έτσι όπως έπραξατε τότε και εσείς στο δικό σας τομέα αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ Πέτερ Σίμων ο κ. Κράσινοδιεύσκη για την ομάδα ECR. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Γερουσιαστή Μόντι που ήρθε εδώ σήμερα. Τρία ερωτήματα σχετικά απλά έχω. Το πρώτο είναι το εξής. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, πράγματι ισχύει ότι η μόνη λύση του προβλήματος ε, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και αφορά αποφυγής, ιδίως από τις διεθνείς ε, επιχειρήσεις και ομιλούς. Αυτή είναι η μόνη λύση, η φορολογική εναρμόνιση δηλαδή συγκέντρωση. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Τέτοιου είδους φορολογική εναρμόνιση. Πράγματι πρέπει να καλύπτει και τους συντελεστές. Τρίτον, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δεν υπάρχουν άλλα μέσα. Να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθείτε μια απλή αρχή. Δηλαδή όπου κερδίζουν τα χρήματά τους, εκεί θα φορολογούνται επιχειρήσεις. Εκεί που γεννάται το κέρδος. Στην Πολωνία γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη ότι γιατί εδώ συχνά ε, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας ε, σε μεγάλες αμερικανικές πολυεθνικέ, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και γαλλικέ γερμανικές εταιρείε ε, στην Πολωνία, στο τομέα τη ελληνική πώληση, δεν πληρώνουν φόρους εκεί που, που, που παράγεται το κέρδος. Ερωτώ δηλαδή μήπω θα έπρεπε να αναζητήσουμε αλλού τρόπου για να ακολουθήσουμε αυτή την πολύ απλή αρχή ε, που και είναι λογική. Δηλαδή να πληρώνουν ο κόσμος το φόρο του εκεί ε, που κερδίζει το εισόδημά του και σε αναλογία με, το, με τα έσοδά του. Συνάδελφος Κόρα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γερουσιαστά Μοντ, χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ σήμερα και έχουμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Καταρχάς, ένα ερώτημα που ίσως μοιάζει με το ερώτημα που έκανε ο κύριος Μπάλτς προλίγο, αλλά θα το επαναλάβω. Έχετε κάνει πολλή δουλειά κατά το παρελθόν ε, για αυτά τα θέματα, μας το επαναλάβατε και τώρα, αλλά τώρα εκ των υστέρων και επειδή βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται η ίδια συζήτηση που είχε γίνει και στη δεκαετία του 90, ε, αν χρειαζόταν να τα ξανακάνετε από την αρχή. Ε, θα τα κάνετε διαφορετικά, θα κάνετε τα ίδια και τι μπορούμε να αποφύγουμε τώρα. Ποιε παγίδε, ε, σε ό,τι αφορά το CCCTB, την κοινωνιοποιημένη βάση φορολογία εταιριών. Συμφωνούμε όλοι ότι ο φόρος πρέπει να πληρώνεται εκεί που έχουμε την προσθέμενη αξία, αλλά και εκεί ξεκινάει η συζήτηση. Ποια είναι αυτή η αξία ακριβώς που πρέπει να Άρα, κατά την άποψή σας, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για την αξία αυτή, διότι στην προηγούμενη πρόταση είδαμε ότι ε, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ε, μια διχοτομία και μια αντιπαράθεση. Και ένα τελευταίο ερώτημα βασίσατε τις ε, εκθέσεις σας και στην ομάδα επαφή σε κάποιες έρευνες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα. Τουλάχιστον αυτές που έγιναν δεκαετία του 90, τις παλιές αυτές δεν θα ήταν χρήσιμο ε, να δημοσιοποιηθούν, να έχουμε πρόσβαση για να διδαχθούμε, να μάθουμε το μάθημά μας. Ε, σας ευχαριστώ την κόρα και τώρα εκ μέρους της Γκουε ο Φάμπιο Ντεμάς έχει το λόγο, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω που ήρθε γιατί ξέρω ότι δεν τον βόλευε και πολύ αυτή η μέρα. Φάμπιο. Thank you, Ευχαριστώ, Αλά. Μόντι, καλημέρα. Αναφερθήκατε στους χαμηλούς καρπούς της ομάδας επαφής του λογικό κώδικα. Καμιά φορά δεν ήταν πρόβλημα ότι οι καρποί ήταν πολύ χαμηλά. Ίσως η ομάδα καθόταν στη σκιά του δέντρου απολαμβάνοντας το φορολογικό παράδεισο. Αυτό είναι αναλόγως πώς τα βλέπει κανείς. Ο κύριος Γιούγκερ είχε συμβάλει τα μάλα για τα φορολογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να τον πείσετε, διότι δεν θα έπρεπε να φοβάται να έρχεται εδώ στην Ειδική Επιτροπή. Μπορούμε να τα κουβεντιάζουμε όμορφα. Τώρα στα σοβαρά. Έχω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη. Αναφερθήκατε στην ομάδα φορολογικής πολιτικής που είχατε προτείνει το 2010. Πόσο σχετική θα μπορούσε να είναι σήμερα να υπάρχει μια τέτοια ομάδα για την φορολογική πολιτική. Δεύτερη ερώτηση. Ο κ. Μοσκοβίτσι είπε ότι προσωπικά θα ήταν υπέρ της δημόσιας πρόσβασης σε ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα rulings και μάθαμε και από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο ότι η πλειοψηφία αυτού είναι υπέρ της πρόσβασης του κοινού στις εκθέσεις κατά χώρα όσον αφορά τις ε, εταιρείε. Συμφωνείτε ότι αυτά τα δύο μέτρα θα ήταν πολύτιμα για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και κυρίως όσον αφορά τον θεμητό φορολογικό ανταγωνισμό. Τρίτον, όταν αναλάβατε σαν επίτροπος υπεύθυνο για τον ανταγωνισμό το 1999 η ε, προσπαθούσε να βρει κατά πόσο επέβαλαν αθέμητη πολιτική τη φορολόγηση π.χ. στα κράτη-μέλη. Και υπήρχαν 24 περιπτώσεις τότε που αναλάβατε που ε, ξεκίνησαν πριν τον Αύγουστο και όταν αναλάβατε εσείς μειώθηκαν πολύ οι υποθέσεις. Μπορείτε να μας πείτε γιατί έγινε κάτι τέτοιο. Τι εμπόδια είχατε συναντήσει τότε. Ευχαριστώ Φάμπιο, εν ονόματι των Πρασίνων η κυρία Εύα Ζολή, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, που είναι εδώ στα δεξιά μας. Η Εύα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γερουσιαστά. Όταν ήσασταν επίτροπος για τα φορολογικά και μετά για τον ανταγωνισμό, ο σχεδιασμός ο φορολογικός, ο επιθετικός, ήδη θεωρείται σαν ένας μεγάλος κίνδυνος. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ε, θα το ανακαλύψουν εκ νέου χάρη στη δουλειά τους των διαφόρων ε, δημοσιογράφων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις υπηρεσίες της κυρίας Βεστάγκερ, μεταξύ του 1999 και του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε την υπόθεση 45 καθεστώτων ή φορολογικών εργαλείων που ήταν προβληματικά. Ανάμεσα στον Ιούλιο του 2004 και Ιούλιο 2014 μόνο 14 περιπτώσεις μελετήθηκαν. Πώς εξηγείτε εσείς με τέτοια διαφορά, πώς εξηγείτε το ότι η Επιτροπή Ευρωπαϊκή Μπαρόσο δεν συνέχισε το έργο που θα εσείς ο ίδιος. Κατά την άποψή σας, στην Επιτροπή μας για, την φο... τον φόρους θα πρέπει να έρθει εδώ για να τον ακούσουμε όσον αυτό το θέμα. Σε μια επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Επιτροπή για τα φορολογικά αναφέρεται ότι πριν το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με μικρό αριθμό tax rulings, διότι από ό,τι φαίνεται τα σήματα συναγερμού εμφανίστηκαν μόλις το 2013. Όταν είσαστε στη θέση αυτή δεν υπήρχαν συγκεκριμένες ενδείξεις όσον αφορά τον προβληματικό χαρακτήρα των tax rulings από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων. Οι συμφωνίες που ήδη συνήθισαν αρχές του 1990 μεταξύ Apple και Ιρλανδίας παραδείγματο χάρη ποτέ δεν είχαν προσελκύσει την ε, προσοχή. Ευχαριστώ Εύα, εν ονόματι του EFTD ο Μάρκο Τζάνι το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον καθηγητή Μόντι. Μια πρώτη σκέψη που αφορά λίγο πολύ αυτό που μας διηγηθήκατε και αυτά που κάνατε στην περίοδο που περάσατε σαν επίτροπος και από ό,τι κατάλαβα το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επιληθεί το πρόβλημα ήταν η έλλειψη μιας πολιτικής βούλησης και ίσως γι' αυτό μετά από τόσα χρόνια ακόμα εδώ συζητούμε και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που δεν θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή όπως είπαν οι συνάδελφοι αλλά πρέπει να είναι σφαιρική όσον αφορά την φοροδιαφυγή. Πρώτη ερώτηση Κατά την άποψή σας, ποια είναι η άποψή σας για το πακέτο που ανακοίνωσε ο Επίτροπος Μοσκοβίτσι. Θεωρείτε ε, ότι η προσέγγιση είναι πολύ ήπια, πολύ soft και είναι μερική διαφάνεια όσον αφορά τις πληροφορίες. Είναι κάτι μικρό για την επίλυση του προβλήματος. Πάνω απ' όλα από αυτή την έποψη η έλλειψη των πληροφοριών είναι κάτι που διαπιστώσαμε εμείς σαν Επιτροπή για τους φόρους ε, έλλειψη στοιχείων για να λύσουμε αυτά τα θέματα και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το προσωπικό των φορολογικών αρχών των εθνικών θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες να αναλύσουν αυτά τα έγγραφα ε, παρά το γεγονός ότι ανοίγουν αυτά τα βιβλία και ανοίγουν τις πόρτες με την αυτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που συχνά δεν αναφέρεται και κατά την άποψή μου όμως είναι σημαντικό και θα πρέπει η Ευρώπη από πλευράς συνθήκων ε, να κινηθεί. Έχει περισσότερα περιθώρια από αυτά που γίνονται από πλευράς. Πρέπει να παρακολουθούν οι συναλλαγές. Οι παράνομες ή παράνομες κάποιας διάστασης περνούν από τις τράπεζες, περνούν από το τραπεζικό σύστημα. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη διαφάνεια, πρέπει να έχουμε πλήρη διαφάνεια του οικονομικού συστήματος για να λυθεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Το σκάνδαλο του Swiss Leaks οι διάφορες αποκαλύψεις του whistleblower Φατσάνη απεκάλυψαν πώς όλα περνούν μέσω των τραπεζών και λείπει αυτή η διαφάνεια. Αν καταφέρουμε να έχουμε διαφάνεια πλήρη όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές, πιθανότατα θα μπορούμε να λύσουμε καλύτερα το όλο πρόβλημα. Σας ρωτώ μήπως θα ήταν καλύτερο και από την άποψη των ευρωπαϊκών συνθήκων να προσπαθήσουμε να κινηθούμε όσον αφορά αυτό το στοιχείο, να κινηθούμε από εκεί την πλευρά, περισσότερο από εκείνη την πλευρά παρά από το δρόμο που ακολουθούμε. Ευχαριστώ Αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κ. Άνεμανς. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κάποια καχυποψία, ε, πρέπει να πω κύριε Μόντι, σήμερα. Είναι και ένας εφημισμός ο φορολογική εναρμόνιση κατά κάποιο τρόπο. θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία. Δεν θέλουμε περισσότερη συγκέντρωση στη σταδιοδρομία σας. Έχετε και εσείς δει ε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάζο μεταξύ αυτών που λέγονται εδώ, έχουμε τα, την πολιτική ορθότητα και αυτά που ακούγονται, αφόρα απέχουν ε, από τις απόψεις των απλών πολιτών η επιτροπή αυτή είναι η επιτροπή Lux Leaks, Lux του σκανδάλου. Γιατί περί σκανδάλου πρόκειται το Λουξεμβούργο. Ήταν το κράτος μέλος ε, από το οποίο ο τότε Πρωθυπουργό και η νύμπα της Κομισιόν οργάνωσε ένα τεράστιο σκάνδαλο ουσιαστικά. Το θέμα είναι Όλο αυτό πρέπει να μας εμπνέει στο να προσθέσουμε στην Ομισματική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και ούτω καθεξής ακόμα ένα ευρωπαϊκό φορέα και θεσμό. Πώς εφαρμόζεται εδώ η αρχή της επικουρικότητας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε, κύριος Πρόεδρος και Ιαστής. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αν και εθίγησαν πολύ άριθμα και ευρύτατα ζητήματα. Ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με το ερώτημα του κυρίου Μπάλτς και πιο γενικά όμως, δηλαδή τι θα μπορούσε να είχε γίνει παραπάνω ή τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικό, διαφορετικά. Ακούστε, στην Ευρώπη, όπως λέει και η Συνδική της Λισαβόνας, θέλουμε να δημιουργήσουμε μία άκρος ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς. Δυσκολευόμαστε όμως να έχουμε μία αγορά ολοκληρωμένη. Επανέρχονται κάποια εθνικιστικά, λαϊκιστικά κινήματα και αντιδράσεις που δεν θέλω να τα σχολιάσω εδώ, όμως αυτά δημιουργούν σίγουρα νέες προκλήσεις στην πτυχή της ολοκλήρωσης της αγοράς. Και ταυτόχρονα η συνδιείσδυση, αν μπορώ να την πω έτσι, των εταιριών, κινήσεις και μετακαταστάσεις εταιριών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει την εντύπωση σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, ε, την εντύπωση και ίσως να είναι και πραγματικότητα ίδια, ότι η ολοκλήρωση των αγορών είναι σε βάρος της διατήρησης του κοινωνικού στοιχείου της αγοράς, της οικονομίας της αγοράς. Πώς πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι αληθεύει ότι οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κυβέρνησεών τους λόγω των τόσο διαφορετικών παραδόσεων. Όμως, δεν θέλουμε, τέλος πάντων εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα οι πολίτες όλο και λιγότερο να εκτιμούν και τελικά να μισούν όλο και περισσότερο την ολοκλήρωση των αγορών στην Ευρώπη, διότι αυτή την εξέλιξη την αντιλαμβάνονται ως εχθρό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Γι' αυτό και στην αναφορά που υπέβαλα το 2010 στον πρόεδρο Μπαρόζο, πρότεινα την ιδέα να εξεταστεί από την τότε Κομισιόν και ίσως και να ισχύει ακόμη, να είναι επίκαιρο ακόμη το θέμα, να εξεταστεί λοιπόν το εδεχόμενο μιας μεγάλης συμφωνίας ε, των αγορών και του κοινωνικού τομέα. Πώς δηλαδή τα κοινωνικά ε, στοιχεία και τα στοιχεία της αγοράς μπορούν να, συγκεντρωθούν και να συνενωθούν σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Το Λουξεμβούργο και άλλες χώρες από πολιτιστικής και πολιτικής πλευράς ε, ενδιαφέρονται ίσως περισσότερο για τις αγορές από ότι για το κοινωνικό επίπεδο, για να τα πω πιο απλά. Ε, Βρετανικά νησιά βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, κεντρική Ανατολική Ευρώπη είναι κρατημέλη και άλλα μεγάλες πυρετικές χώρες, μέλη της Ευρωζώνης κυρίως, που η Γαλλία, στο τοπικό, το χαρακτηριστικό παράδειγμα, που είναι πιο προσιλωμένη στο κοινωνικό στοιχείο. Και βλέπουμε κάποια καχυποψία ε, ενίοτε την πλήρη αυτή ολοκλήρωση των αγορών και την οικονομία της αγοράς. Εγώ όμως φοβούμαι ότι μια ανταγωνιστική ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να έχουμε μόνο αν συμφιλιώσουμε καλύτερα αυτές τις πτυχές, διότι δεν μπορούμε να παρετηθούμε της διάστασης της ολοκληρωμένης αγοράς, γιατί έτσι θα απολέσουμε έδαφος σε ό,τι αφορά την και της οικονομίες κλίμακας. Ούτε όμως μπορούμε να παρατηθούμε και των βασικών στοιχείων του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε η Κομισιόν κάποια μέρα να προτείνει στα κράτη-μέλη να δεχθούν ένα deal, μια συμφωνία, όπου οι υπέρμαχοι της αγοράς να έχουν μεγαλύτερη ολοκλήρωση των αγορών η αγορά υπηρεσιών, για παράδειγμα, οικονομία, ενέργεια, επαγγέλματα. Θεωρητικά μέχρι στιγμής είναι αυτά. Να τα προχωρήσουν αυτά τα κράτη αυτά, αλλά να βοηθήσουν ώστε να αποτραπεί η κατάσταση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Και να υπάρξει, ας πούμε, αυτό το αντάλλαγμα, δηλαδή να υπάρξει ένα φορολογικού συντονισμού για να μην διαβρωθεί από το φορολογικό ανταγωνισμό, ε, να μην διαβρωθούν τα φορολογικά έσοδα και να μπορούν να καλυφθούν κοινωνικέ ανάγκες. Να γυρίσω πίσω στο χρόνο που δεν είναι και τόσο πάντα επικοδομητικό συγχείρημα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα πάντως ε, να επιλέξω τι συγκεκριμένα δεν πήγε καλά από τεχνικής πλευράς. Αυτή η ενδεχόμενη μόχλευση όμως από μια νέα, από ένα νέο συμβόλαιο αν θέλετε Ευρωπαϊκή Συμβίωση είναι κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί. Σε σχέση με το ερώτημα του κυρίου Πέτερ Ζήμου, μιλήσατε και για το πακέτο Monty Cross, Das for Zorge αν το προφέρω καλά. Χαίρομαι που λέτε ότι ήταν χρήσιμο αυτό το πακέτο και αφού ήταν και επειδή μίλησα πριν για το πώς μπορούμε να καθησυχάσουμε τους υπουργούς οικονομικών, τέτοιου είδους ε, διευκρινήσεις κάποιων αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις, για τις υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, αυτό ήταν πάρα πολύ καθησυχαστικό για τη Γερμανία συγκεκριμένα, και πιο συγκεκριμένα για το επίπεδο των περιφερειών και των κρατηδίων που για δεκαετίες ένιωθαν ότι απειλούνται από ιδέες που δεν υπήρχαν καν στο μυαλό των ε, επιτρόπων ε, ότι θα επιτεθούν κατά του κοινωνικού στοιχείου και αυτό το ακούγε κανείς σε εκπομπές ε, και το διάβαζε στον τύπο. Υπήρχαν χώρες προρομαντικές και συναισθηματικές ε, και όλες αυτές οι χώρες έχουν τα φαντάσματά τους κατά κάποιο τρόπο και ίσως ε, τα κοιμήσαμε αυτά ε, με το πακέτο μας τότε, το πακέτο Monte Cruz. Τώρα δεν ξέρω μπορούμε να δώσουμε τις ίδιες διευκρινήσεις ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σήμερα ε, και πάντα, ε, στο πλαίσιο του φορολογικού ανταγωνισμού. Πάντως αυτά τα οποία θέλει να πετύχει ο Νίνα αρμόδιος για φορολογία επίτροπος με βρίσκουν σύμφωνο και είμαι πολύ αισιόδοξο κάτι που διατρέχει πολλές παρεμβάσεις. Δεν θέλω να φέρω και δεν, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα όλου του που το ανέφεραν, αλλά υπάρχει μια θετική διαφορά τώρα σε σχέση με το τι έγινε πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή, ε, μεσολάβησε η δημοσιονομική κρίση που είχε πολλά αρνητικά, αλλά έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και έκανε και την ομάδα των 20 και των ΩΣΑ να σημειώσουν πρόοδο, να ανησυχήσουν και να προχωρήσουν σε μέτρα για την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων και υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλά από ευρωπαϊκής πλευράς και γενικότερα. Άρα Νομίζω ότι πλέον είναι πιο πρόσφορο σήμερα το έδαφος για μια διεθνή συνεργασία που αποσκοπεί στην κατάργηση των ακραίων στρεβλώσεων που έχουν να κάνουν με την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Τώρα, κατά πόσο χρειάζεται απαραίτητο αναρμόνιση των αφορικών συντελεστών, ίσως όχι, όπως είπαμε και πριν. Ε, αυτό που θα πρότεινα όμως εν γέννη είναι, και με βέβαιος ότι και ο κύριος Μοσκοβισή το έχει υπόψη του, με ή χωρίς μία νεοσύστατη ομάδα πολιτικής, να συνεργαστεί στενά με τα διεθνή βήματα συζήτησης, όπου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι κάλυψα τις παρατηρήσεις του κύριου Κρασνοβεύσκη κάπως έτσι και της κυρίας Κοροβανίμ. Α, κόρα, μάλιστα. Της κόρα, καλύτερα, ναι, για να είμαστε πιο απλοί. Τώρα το τον κύριο Ντεμάση και την κυρία Ζολή. Πάρουμε μαζί τον κύριο Ντεμάζη και την κυρία Ζολή Πρέπει να εξετάσω τα στοιχεία, διότι η κυρία Ζολή έχει την τάση να επενεί την περίοδο κατά την οποία υπήρξε επίτροπος ανταγωνισμού διότι υπήρχε μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που εξετάστηκε από πλευράς κρατικών ενισχύσεων φορολογικών ενισχύσεων 45 και μετά είδαμε ένα είδος μείωση, απεργίας ούτως υπήν. Ο κ. Ντεμάζη με ρωτά κατά πόσο μπορώ να απαλλαγώ από την κατηγορία που δεν την έχω δει ακόμα. Να δω τα στοιχεία. Ότι ήτανε, υπήρχε μεγάλη ενεργητικότητα όσον αφορά την καταπολέμηση των ενισχύσεων. Τα στοιχεία σας. Μέχρι τον Αύγουστο του 1999 και την ακόλουθη περίοδο αναφέρονται σε κρατικές ενισχύσεις ή φορολογικών κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα στις μου, η Γενική Διεύθυνση υπεύθυνη τον ανταγωνισμό ερεύνησε 24 κρίσεις κρατικών ενισχύσεων, φορολογικών ενισχύσεων, κρατικών ενισχύσεων ή φορολογικών κρατικών ενισχύσεων. Απάντηση κρατικών ενισχύσεων για θέματα φορολόγησης και μετά ο αριθμός ε, μειώθηκε. Θα κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Θα υπάρξει διαφάνεια, είναι η απάντηση του κυρίου Μόντι. Κύριος Τζάνι. Βέβαια είναι θέμα πολιτικής βουλήσεως και η πολιτική βούληση θα πρέπει να υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι το εγχείρημά σας θα συμβάλλει τα μάλα στην δημιουργία κάποια ενοχλήσεως εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Θα βρεθούν οι πολιτικοί σε δυσχερή θέση αν δεν δείξουν την ανάλογη πολιτική βούληση. Αν θεωρώ ότι το πακέτο του Επιτρόπου Μοσκοβίτση αν είναι πολύ ήπιο, σαν δέσμη μέτρων, από αυτά που μου περιέγραψε δεν σχημάτισα τέτοια εντύπωση. Τέλος, μεγαλύτερη διαφάνεια, κύριε Τζάνι, όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές, δεν θα διευκόλυνε την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Σίγουρα ναι. Αυτό ισχύει και στα κράτη-μέλη. Αυτά κάθε αυτά. Γι' αυτό όταν ήμουν επικεφαλής Ιταλική κυβερνήσεω θέλαμε να αυξήσουμε και αυξήσαμε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ένα από τα βασικά μέτρα που θεσπίστηκε το Δεκέμβριο 2011 ε, συνέβαλε στο να υπάρχει διαφάνεια των ε, τραπεζικών συναλλαγών για τις, ταξικές, για τις φορολογικές αρχές. Κύριε Σάνεμαντς μετά. Αναφερθήκατε στο LuxLeaks, είπατε ότι είναι σκάνδαλο, αλλά ποια ήταν η ερώτησή σας? Ε, επικουρικότητα. Πιστεύω ότι η επικουρικότητα έχει μεγάλο ρόλο να παίξει στην Ένωση μας και μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή διαφόρων πολιτικών. Πριν από κάποια χρόνια Μία πολιτική που πάντα ήταν το αποκλειστικό φρούριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είναι η πολιτική ανταγωνισμού, αποτέλεσε αντικείμενο τεράστιας διαθροτικής μεταμόρφωσης μέσω μεταρρυθμιστικών εξυγχρονισμών και το πνεύμα της επικουρικότητας πολλές αρμοδιότητες δόθηκαν σε δίκτυο διακυβέρνησης που απαρτίζεται από τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κέντρο. Πιστεύω ότι η επικουρικότητα σημαίνει ότι και αρμοδιότητες άλλες ίσως πρέπει να απαιτείται να συγκεντρωθούν και κάποιες πτυχές φορολογικές τώρα, σε αυτή τη φάση, δεν θα πληρούσαν τα κριτήρια της επικουρικότητας για να παραμείνουν εντελώς αποκεντρωμένες και ίσως χρειάζεται μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης. Ευχαριστώ κύριε Γερουσιαστά, κύριε Πρόεδρε που απαντήσατε στο σύνολο των ερωτήσεων που σας ετέθησαν. Ουσιαστικά μας υπενθυμίσατε πέρα από τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία απαντήσατε, μας επιθυμήσατε εν γέννη ότι όλα αυτά είναι στο επίκεντρο των πολιτικών επιλογών. Οι αποφάσεις που αντιστοιχούν στο θέμα αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις. Εν την πλήρη ενία της λέξης και αν θέλουμε να προχωρήσουμε πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση σε όλα τα κράτη-μέλη. Απαιτείται ομοφωνία όσον αφορά τα φορολογικά και παραμένει εθνική αρμοδιότητα, πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν την, την κυριαρχία όσον αφορά τα θέματα φορολόγησης, θα πρέπει όμως να υπάρχει πολιτική βούληση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Εργάνων, βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό έλεγε η κυρία Ζολή και ο κ. Τομάζη Αυτά ανέφεραν όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Σε κάποια φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μεγάλη πολιτική βούληση και σε κάποια φάση αυτή η βούληση απεδυναμώθη. Βούληση του Κοινοβουλίου. Και εκεί αυτό είναι δική μας ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γερουσιαστά. Ευχαριστώ πολύ. Mes chers Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε, ε, μάλλον ας παραλάβουμε τώρα τις εργασίες μας, λέει ο πρόεδρος ε, Λαμασούρ. Έχουμε τώρα δύο προσωπικότητες, ε, των οποίων θα ακροαστούμε. Περιμένω να ξανακαθίσουν οι δύο συνεισηγητές που αποχαιρετούν τον ε, πρόεδρο Μόντι. Κυρία Ελίζα και Μιχαήλ, παρακαλώ. Ελίζα Μιχαήλ. Ελίζα Μιχαήλ, do you want to take the floor or... Ελίζα uh, και Μιχαήλ, θα θέλατε, ή μάλλον τώρα θα ακούσουμε την κυρία Ρίδινγκ. Θέλετε να θέσετε ερωτήσεις πριν από την παρέμβασή της ή να ακούσουμε πρώτα. Καλύτερα να ακούσουμε, λέει να ακούσουμε πρώτα τι έχει να πει, γιατί μετά θα προκύψουν από αυτά ερωτήσεις. Σας παρακαλώ όμως κάντε ησυχία. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Τόβε Μαρία Ρίδινγκ που είναι Policy Advocacy ε, Manager του, του οργανισμού. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν η κυρία που θα καταθέσει τη μαρτυρία να καθίσει δίπλα σας ε, στα έδρανα του Προεδρείου γιατί είναι δύσκολο να θέτουμε ερωτήσει στην πλάτη της. Ο πρόεδρος Λαμασούρ. ας καθίσει ο, εκεί όπου βρίσκεται η κυρία Ρίτινγκ, δηλαδή στην πρώτη σειρά εδράνων. Αν θέλετε κυρία Ρίντινγκ σας παρακαλώ πρώτα παρουσιάστε τον οργανισμό σας, γνωρίζετε το αντικείμενο των συζητήσεών μα, όπως και ο κύριος Ντελτούρ, άλλωστε έχετε συμμετάσχει στις συναντήσεις μας από την αρχή. Αν ε, θα θέλατε λοιπόν για λίγα λεπτά να καταθέσετε την μαρτυρία σας ενδεχομένως και συστάσεις και μετά θα δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές και του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Κύριε Ρίτινγκ, έχετε εσεί τον λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο τη επιτροπή σα για την πρόσκληση να έρθω εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Χρέος και την Ανάπτυξη, Eurodad, είμαστε στο πλαίσιο του δικτύου ε, για τη δικαιοσύνη ένα μέρος από, που απαρτίζεται από πάνω από 50 οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς στα ζητήματα, παρακολουθούμε την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμιο. Διότι τώρα έχουμε μια παγκόσμια συμμαχία για τη φορολογική δικαιοσύνη και συνεργαζόμαστε και με εταίρους από τον Νότο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για το ζήτημα που συζητούμε σήμερα, δηλαδή τη διεθνή διάσταση. Θα αναφέρω όμως και τις λύσεις που θα πρότεινα. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να πω κάτι για τη σημασία του να έχουμε μία έρευνα και παρακολούθηση της υπόθεσης LuxLeaks που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ένα σκάνδαλο που σόκαρε και άνοιξε τα μάτια σε πολλούς. Έχουμε περάσει από μια δημοσιονομική οικονομική κρίση, απολυτότητα, έχουμε απώλειες θέσεων εργασίας, μείωση ε, και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, χρηματοοικονομική αβεβαιότητα. Και μετά από όλα αυτά αποκαλύπτεται έφνης ότι εκατοντάδες πολυεθνικές επιχειρήσεις ε, είχαν ε, κρυφές συμφωνίες με το Λουξεμβούργο που τους επέτρεπε να έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα φωλικών συλλεστών μέχρι και σε γελίος, γελία χαμηλά επίπεδα της άξιος του 1%. Μπορεί να φαίνεται ε, στο μάτια της κοινή γνώμης παράξενο ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη έρευνα, παρακολούθηση, ε, δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για αυτούς που φαίνεται ότι ήταν αναμεμειγμένοι, δεν υπήρξε καμία ανάληψη ευθύνη, ούτε και μια αξιόπιστη υπόσχεση αλλαγή. Οι εταιρείε που συμμετείχαν φαίνεται ότι συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους και ακόμη και τώρα δεν ξέρουμε τι φόρους πληρώνουν και επίσης έχουμε και μια συνεχή ροή σκανδάλων που ε, γίνονται πρωτοσέλιδο και που αφορούν περισσότερες εταιρείες, περισσότερες κυβερνήσεις και σαφώς όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ λάθος. Ο ο άνθρωπος ο οποίος ε, ηγείται του Λουξεμβούργου στην εποχή που υπεγράφουν αυτές οι ειδικέ ε, ε, αποκλειστικέ συμφωνίε εξελέγει σε ένα από τα πιο ισχυρά αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Είναι δηλαδή επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για την ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποτίθεται ότι θα προτείνει νομοθετικές αλλαγές για να διορθώσει το σύστημα. Ίσως να είναι καλές οι προθέσεις του, δεν τις έχουμε δει όμως ακόμη. Τώρα, στα μάτια τη κοινή γνώμης, η κατάσταση κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει πιο εύκολα κατανοητή, ε, ιδίω όταν σε ένα μήνα από τώρα το Λουξεμβούργο θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η Προεδρία αλλάζει χέρια κάθε έξι μήνες. Σε καμιά, ε, περίπτωση όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε ότι είναι σαν να έχουμε βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα στην προκειμένη περίπτωση. Και επίσης θα ξεκινήσουν ε, ε, και κάποιες ε, δίκες στο Λουξεμβούργο με στόχο δύο πληροφοριοδότες και έναν δημοσιογράφο μεταξύ αυτών που εξέθεσαν το σκάνδαλο. Τα άτομα αυτά που το μόνο έγκλημα που έκαναν ήταν να μας πούν την αλήθεια κινδυνεύουν τώρα να μπουν στη φυλακή για χρόνια. Και εδώ πια είναι ώρα να διαρωτηθούμε σε τι κοινωνία ζούμε. Αυτοί οι άνθρωποι αποκάλυψαν ότι οι κοινωνίες μας χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ. Και τελικά τι συνέβη, σημαίνει να τους, ε, το μόνο που συνέβη ήταν ότι μηνύθηκαν και θα δικαστούν. Ενώ στο μεταξύ οι πολυεθνικές εταιρείες, οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις που ήταν υπεύθυνοι φαίνεται ότι τη γλιτώνουν χωρίς καμία επίπτωση και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται ότι διευρύνεται η εξουσία τους και κάποιοι εκλέγονται και σε κορυφαίες θέσεις, αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να ε, κλείσουμε τα μάτια μας στο ότι εδώ μιλάμε για μια ορολογιακή βόμβα που πλήττει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Το να γνωρίσουμε τα LuxLeaks δεν θα ε, οδηγήσει μακριά αυτή την ορολογιακή βόμβα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται πλέον να είναι η καλύτερη, η, μεγαλύτερη ελπίδα των πολιτών ότι τουλάχιστον ένας θεσμός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αφήσει την κατάσταση να συνεχιστεί. Και χαιρό, ε, μάλλον λυπόμαστε πολύ που εμποδίζουν οι πολυεθνικές το έργο αυτής της Επιτροπής σας, γιατί αρνούνται να έρθουν εδώ, αρνούνται να συνομιλήσουν μαζί σα, αλλά υπάρχουν και ευρωπαϊκέ κυβερνήσει που δεν θέλουν να έρθουν εδώ για να συζητήσουν το θέμα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα μεγαλώσει την αποφασιστικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσει τον αγώνα του, να εκθέσει την αλήθεια, να μεταρρυθμίσει όλο αυτό το σύστημα και να εισαγάγει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα, τη λογοδοσία και τη φορολογική δικαιοσύνη. Και βέβαια να θεσπίσει και ένα πλαίσιο προστασία για του πληροφοριοδότε και σύντομα ελπίζω να ξυπνήσει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διεθνή διάσταση, δυστυχώς δεν έχουμε μόνο στην Ευρώπη ε, την κατακραυγή για τα θέματα της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής πολλά στοιχεία, πολλές ενδείξεις έχουμε ότι τα προβλήματα αυτά πλήττουν τις αναπτυσσόμενες χώρες πολύ περισσότερο από ότι εμάς, τι ανεπτυγμένε. και στις αναπτυσσόμενες χώρες η συζήτηση για αυτό το θέμα, τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροέ κλιμακώνεται. Πρόσφατα είχαμε την έκθεση του πάνελ υψηλού επίπεδου με πρόεδρο τον Τάμπο Μπέκη, έως ε, πρόεδρο ε, της Νοτιοαφρικής. Και εκεί ε, φάνηκε ότι η Αφρική σήμερα χάνει περισσότερα χρήματα λόγω των παράνομων ροών από αυτά τα οποία παίρνει υπομορφή μορφή βοήθειας και από αυτή την ε, σκοπιά ε, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ήταν τόσο δύσκολη η προσπάθεια καταπολέμησης και εκρίζωσης της φτώχειας. Η έκθεση Μπέκη επίσης ε, λέει ότι είναι κάπως αντιφατικό για τις αναπτυγμένες χώρες να συνεχίζουν να παρέχουν τεχνική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική ενώ ταυτόχρονα διατηρούν φορολογικούς κανόνες που επιτρέπουν την αφέμαξη των πόρων αυτής της υπήρου μέσω των παράνομων χρηματοοικονομικών ε, Δεν λειτουργούν τα παγκόσμια πρότυπα φορολόγησης. Αυτό το βλέπουν πλέον ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αρχίζουν να βλέπουν ότι τους κοστίζει και σε πόρους και αρχίζουν να διερωτώνται πώς αναπτύσσονται αυτά τα ε, πρότυπα. Μήπως αποφασίζονται και κλεισμένα των θυρών στον ΩΣΑ, στο Παρίσι, μια διαδικασία που πάνω από 100 αναπτυσσόμενες χώρες αποκλείονται, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό. Έχουν λοιπόν τώρα καταθέσει μια πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη από τις όμενες χώρες να υπάρξει μια φορολογική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι χώρες και όπου εκεί θα μπορέσουν να βρεθούν πραγματικά παγκόσμιες λύσεις. Πρόσφατα το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση αυτή και είμαστε γνώμονες γι' αυτό. Όμως αυτό που δεν μας αρέσει είναι το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αρνούνται να δεχτούν την πρόταση αυτή προς το παρόν. Είναι πραγματικά πορεία άξιων. Ευρωπαϊκέ κυβερνήσει που περηφανεύονται για το πόσο δημοκρατικέ είναι, αυτέ οι χώρε και αυτέ οι κυβερνήσει να προασπίζονται το δικαίωμα μια αποκλειστική λέσχη χωρών να αποφασίζουν για του κανόνε που που θα ισχύουν για όλου του άλλου. Οι κυβερνήσει των ευρωπαϊκών χωρών τη Ένωση υποστηρίζουν ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε ε, συμμετέχουν ε, στην διαδικασία BEPS του ΩΣΑ και ότι λαμβάνονται υπόψη ανησυχίε του. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι λίγε από αυτέ τι χώρε έχουν προσκληθεί σε ορισμένε από τι συναντήσει, ενώ πάνω από 100 χώρε παραμένουν αποκλεισμένε και ενώ υπήρξαν διάφορε προτάσει πέρυσι για το πώ μπορούν να προωθηθούν τα συμφέροντα των πιο φτωχών χωρών και θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διαδικασία BEPS, όλες αυτές τις προτάσεις απορρίφθηκαν. Από τον σαν ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, σε αυτό θα καταλήξω. Τέλος θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι είναι πιο αποτελεσματικό να αποκλειστούν οι περισσότερες χώρες από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ωστόσο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο πυρήνας του προβλήματος είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους οι κυβερνήσεις και γι' αυτό έχουμε κρίση στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λύσεις, πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία όπου πάει κόσμος φυλακή επειδή είπε την αλήθεια για το πόσους φόρους πληρώνουν οι πολυεθνικές. Γι' αυτό χρειάζεται δημόσια υποβολή εκθέσεων αναχώρα για να δούμε τι πληρώνουν τελικά πραγματικά οι εταιρείε και όλοι είμαστε ε, και όλοι θέλουμε να στηρίξουμε τις ε, προτάσεις για αυτή την ε, αναφορά αναχώρα. Χρειάζεται επίσης ε, μια οδηγία για την προστασία των πληροφοριοδοτών και χρειαζόμαστε και ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεν μπορούν ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις τεράστιες πολυεθνικές που δεν πληρώνουν τους φόρους τους. Δεν μπορούμε να έχουμε εταιρείε που χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η παιδεία, το κράτος δικαίου, υποδομές, αλλά τα κέρδη τους να τα ε, αφήνουν ε, σε φορολογικούς παραδείσους και να μην συνεισφέρουν στην ε, πληρωμή για αυτές τις υπηρεσίες. Και το τελευταίο είναι ότι εάν θέλουμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα πρέπει να έχουμε μια αρχή που θα αποτρέπει από τα μονό κράτη-μέλη να καταστρέφουν τη φορολογική βάση άλλων κρατών. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση τη περιβαλλοντική ρήπανση. Για τα χημικά, για παράδειγμα, γενικώ αποδεκτό είναι ότι δεν μπορεί μια χώρα να ε, ρίχνει τα χημικά της ε, σε μια άλλη ε, χώρα και υπάρχει προστασία. Ή για τους γενετικούς πόρους υπάρχει σύμβαση που λέει ότι μόνο αν η χώρα υποδοχής ή εγκατάσταση πολυεθνικής, μόνο αν αυτή λοιπόν η χώρα συμμορφώνεται σε διεθνή πρότυπα, μπορεί να συμμετέχει η εταιρεία της σε άλλες δικαιοδοσίες. Και ελπίζω στις 10 Ιουνίου να ψηφιστεί αυτή η διάσταση που είπα της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για τις προτάσεις σας και για τη δουλειά που κάνατε. Κάνατε πολλή δουλειά σαν οργανισμός που είναι σημαντικότατο για μας και χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος που μπορούμε να ωφεληθούμε από την σοβαρή σας συνεισφορά. Για τις λεπτομέρειες, είπατε ότι το Κοινοβούλιο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο βέλτιστο βαθμό την ευκαιρία και να καλύψει τα κενά που υπάρχουν. Αναφερθήκατε σε κάποια κενά, τις εκθέσεις κατά χώρα, την ανάγκη να προστατευτούν οι πληροφοριοδότες. Τι άλλο έχετε στο πρόγραμμά σας που μπορείτε να μας προτείνετε επεξεργαζόμαστε το θέμα της κοινή ενωπημένης εταιρική φορολογικής βάσης και να έχουμε ε, κάποια μαύρη λίστα για νομοθεσίες ευρωπαϊκές που δεν μπορούν να συνεργαστούν. Πώς, μπορείτε, πώς μπορούμε να το ε, εφαρμόσουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε το πλαίσιο αυτό των rulings και των διαφόρων πρακτικών. Αν έχετε κάποια άλλα στοιχεία στα οποία θα θέλατε να επεκταθείτε, θα ήταν ε, σημαντικό να γίνει. Παρακαλώ μπορείτε να συνοψίσετε τα στοιχεία που μπορέσατε να ε, συλλέξετε για τον αντίκτυπο που έχουν τα διάφορα γεγονότα στις γειτονικέ χώρες, τα φαινόμενα spillover και εντός και εκτός Ευρώπης. Τέλος, μπορείτε να εξηγήσετε λεπτομερέστερα ποια στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας με τους φορολογικούς παραδείσους. Τι ρόλο παίζουν οι φορολογικοί παράδοση στο βαθμό που μπορείτε να το εξηγήσετε στην όλη διαδικασία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει. Και τι μπορούμε να πετύχουμε πάνω σε αυτό μόνο μέσω ε, διεθνών διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ Ελίζα. Μάικλ Τόραν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ρίντινγκ για την παρουσίαση. Θα ήθελα να εστιαστώ επί των στοιχείων που συλλέγεται και δημοσιεύεται. Πολύ σημαντικό το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συλλέγουν στοιχεία. Το ότι είναι υπέρ της διαφάνειας. Θα είχα την καλοσύνη να μας πείτε ποια εμπόδια υπάρχουν όσον αφορά τη συλλογή των στοιχείων. Ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε και αντιμετωπίζετε. Έχετε κάποια παραδείγματα όπου μπορούμε να δούμε γιατί πιέζεται για μια άλλη βάση δεδομένων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα που έχω να σας θέσω. Ευχαριστώ. Προτείνω να κάνουμε αυτό που κάναμε. Να δώσουμε το λόγο σε εκπρόσωπο της κάθε ομάδας και μετά, κυρία μου, μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Για το ΕΛΚ, ο κύριος Τόμας Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρίντινγκ, αναφερθήκατε στην κρατική χρέωση, στο δημόσιο χρέος δηλαδή, αναπτυσσόμενων χωρών. Είπατε επίσης ότι υπάρχει μια, συμμαχία, μια συμμαχία συγγνώμη, για την φορολογική δικαιοσύνη. Αυτό βέβαια πρέπει να έχει και μια παγκόσμια διάσταση. Στον ευρωπαϊκό χώρο και ιδίω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Αναφέρθηκε πριν η έκθεση Μόντι στη συζήτηση που διεξήχθη. Επίσης στην Επιτροπή Οικονομικών, όπου εδώ υπάρχουν και ορισμένα μέλη τη, μιλούμε πάντα για την αποξήρανση των φορολογικών παραδείσων. Βεβαίως η πρόοδος εκεί είναι πολύ αργή διότι πολλές χώρες δεν συμβαδίζουν, δεν συνεργάζονται. Πολλοί μας είπαν αυτά που λέτε ε, δεν αρκούν. Κοιτάξτε, κάνουμε προσπάθειες. Τώρα, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορολογικών αρχών θα πρέπει να είναι αυτόματη. Και για τις, χώρες, ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να ισχύσει αυτό. Δεύτερο, έχουμε το κόνσεπτ του ΟΟΣΑ tax inspectors χωρίς σύνορα. Εάν συμμετάσχουμε τώρα εκεί ή αν προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε και τις χώρες μέλη, κατά πόσον θα είναι δυνατόν να συμμετάσχουν και οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες κατοφλίου. Τρίτο, υπάρχει σε μια έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών για λογαριασμό της Επιτροπής Ανάπτυξης μια αξίωση. Λέμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην συνεργάζονται πλέον με χώρες οι οποίες δηλώνουν ότι δεν είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν μαζί μας για φορολογικά θέματα. Αυτό θεωρείται ότι είναι κάτι που στερείται ουσίας, είναι απλώς ευχολόγιο, ενώ εμείς θέλουμε να σταματήσουμε την φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, καθώς και την μετατόπιση των κερδών. Θεωρείτε ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν κάποιες ουσιώδεις αλλαγές ή θεωρείτε ότι το όσα έχουμε κάνει ως τώρα είναι υπερβολικά λίγα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Κοφούντ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θαυμάσια παρουσίαση. Ευχαριστώ και για το έργο σας εδώ. Είμαι ακριβώς πίσω σας. Για το έργο που κάνετε, για τον εντοπισμό δηλαδή ε, κενών στην νομοθεσία και στη διεθνή νομοθεσία αλλά και στη διεθνή φορολογική νομοθεσία. Είναι σημαντικό το έργο που ε, πράτεται και κάτι αναγκαίο. Βεβαίως και η Επιτροπή μας εδώ θέλουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να πάυσει αυτός ο καταστροφικός φορολογικός ανταγωνισμός. Επιτρέψτε να σας κάνω λίγες ερωτήσεις. Και πρώτα, οι περισσότερες από τις συστάσεις σας συμβαδίζουν με αυτά που λέμε εδώ. Για παράδειγμα, η υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Είδαμε όμως ότι ορισμένοι δεν συμφωνούν. Δεν θέλουν να αλλάξουν τις πρακτικές τους. Με το επιχείρημα συγνά ότι αυτό οδηγεί σε μειονεκτήματα μέσα σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ποια είναι λοιπόν, ποιες προτάσεις μπορεί να έχετε, αφενός βέβαια μπορούν να επιβληθούν με αξαναγκαστικό τρόπο μέτρα, αλλά τι, ποια μέτρα θεωρείτε ότι θα έχουν τις ε, ε, εντονότερες επιπτώσεις και στις κυβερνήσεις για να προκαλέσουν τις αλλαγές στα θέματα αυτά. Και το άλλο τώρα για τις εκθέσεις αναχώρα, country by country reporting. Ακόμα και αν γίνει αυτό και λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις διάφορες εταιρείε από τη δική σας σκοπιά, τι είδους πλαίσιο μπορεί να μας βοηθήσει για να ξεκλειδώσουμε τις πληροφορίες αυτές, διότι θα είναι πολλές οι πληροφορίες αν έχουμε country by country reporting. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε οι πληροφορίες αυτές να είναι χρήσιμες για να σταματήσουν αυτές οι αθέμητες φορολογικές πρακτικές. Τέλος, ποια είναι η άποψή σας για τον ΩΣΑ, για τις πρωτοβουλίες ε, δηλαδή, για τη μετακίνηση των κερδών κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Μπέρντ Λούκε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής της ομάδας ECR. Θα μιλήσω γερμανικά, λέει ο κύριος Λούκε. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω στην υποβολή εκθέσεων αναχώρα, country by country reporting. Πρώτη ερώτηση. Συχνά προβάλλεται η αντίρρηση σε αυτό το country by country reporting ότι μπορεί, μπορούν ή μάλλον θα χρειαστεί να αποκαλυφθούν και ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες μιας επιχειρήσεως. Ερώτηση, συμφωνείτε ή ενδεχομένως ποιο θεωρείται ότι μπορεί να είναι το ελάχιστο των πληροφοριών που θα πρέπει να δημοσιεύονται από επιχειρήσεις, ώστε να διαθέτουμε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με το σε ποιο βαθμό φορολογούνται οι επιχειρήσεις, να μπορέσουμε επίσης να εντοπίσουμε φορολογικούς παραδείσους και θεωρείται ότι μεταξύ των πληροφοριών αυτών θα συμπεριλαμβάνονται και ευαίσθητες πληροφορίες ή μπορεί αυτό να αποφευθεί. Δεύτερον, αν θεωρείτε και εσείς ότι οι πληροφορίε αυτέ ενδεχομένω δεν είναι καν τόσο ευαίσθητες. Μπορούν βεβαίω να επικύλουν οι απόψει και από την πλευρά των επιχειρήσεων μπορεί να κρίνεται διαφορετικά. Το ερώτημα είναι, μπορεί τουλάχιστον ένα μέρος του σκοπού του country by country reporting να επιτευχθεί με την ε, διάθεση των πληροφοριών ανωνύμως. Να μην απαιτείται δηλαδή να αποκαλύπτουν οι επιχειρήσεις με ποιο τρόπο φορολογούνται τα διάφορα τμήματά τους που είναι κατεστημένα σε άλλες χώρες, αλλά να υποχρεούνται οι φορολογικές διοικήσεις στις διάφορες αυτές χώρες να, θέτουν, να διαθέτουν τα δεδομένα αυτά ανώνυμα, βέβαια θα πρόκειται για πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεις και αυτό είναι το ερώτημά μου πλέον, δεν θα μπορούν πλέον να εντοπίζονται οι επιχειρήσεις αυτές, ώστε η ένστασή τους ότι πρόκειται για ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες δεν θα ισχύει πλέον. Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η πρόταση αυτή. Αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ τον φιλελευθέρων. Η κυρία Γκουλάρ μου φαίνεται δεν είναι παρούσα. Και Φάμπιο Ντεμάση από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ρίντεν που είστε εδώ μαζί μας. Πρώτη ερώτηση. Ασχοληθήκατε και με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κρίνεται ότι υπάρχει επαρκής πρόοδος στα πλαίσια του ΟΣΑ και των άλλων πρωτοβουλειών και των πολυμερών βημάτων συζητήσεων για τη μετώπιση του προβλήματος της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι πολλοί ύποπτοι ξεπλένουν το χρήμα τους στο Λουξεμβούργο και στερούν ε, το φόρο που θα έπρεπε να πληρώσουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς το βλέπετε με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Τρίτον, ήμασταν στο Λουξεμβούργο, συνομιλήσαμε τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας και μας είπε οι φορολογικές μας αρχές καμιά φορά ειδοποίησαν τη Γερμανία και τη Γαλλία για ασυνήθη κέρδη, πολύ μεγάλα κέρδη που δηλώθηκαν στο Λουξεμβούργο και δεν αντέδρασαν. Κάποιοι υπουργοί οικονομικών λοιπόν κοιμόταν τότε οι φορολογικές αρχές τους. Αυτό είναι το υπόβαθρο. Θεωρείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να λαμβάνει η χώρα με διαφάνεια, βέβαια να μην αποκαλύπτονται πολύ ευαίσθητες πληροφορίες που δεν έχουν σχέση με τη φορολόγηση. Είπε ο κ. Μοσκοβισή ότι είναι υπέρ αυτού. Η ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς πρόσβαση του κοινού, τι αξία θα είχε. Και όσον αφορά την καταχώρα έκθεση, το Κοινοβούλιο της Ολλανδίας υπερψήφισε την πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες. Θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση του κοινού ούτω ώστε τελικά να ξυπνήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Φάμπιο για τους πράσινους. Εύα Ζολή, Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ που ήρθατε εδώ σήμερα και μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας, τη μεγάλη σας εμπειρία και την αξιολόγησή σας σχετικά με το τι χάνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες λόγω των φορολογικών προβλημάτων και ακούσαμε και στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα για το 2009. Ενδιαφέροντα αυτά διότι ίσως να χάθηκαν πολύ περισσότερα χρήματα στις παράνομες χρηματοπιστωτικές ροές από τις χώρες αυτές από ό,τι δέχτηκαν σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πολύ καλό να αξιολογήσουμε πόσα χρήματα έχασαν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προβούν σε μία αξιολόγηση των διαφόρων φορολογικών καθεστώτων. Καλώς. Έχουμε αγγλικά, γαλλικά. Ήταν έκπληξη ίσως που μίλησα νορβηγικά. Λοιπόν, να επαναλαμβάνω την ερώτηση. Σύμφωνα με μια έκθεση νορβηγική, οι αναπτυσσόμενες χώρες χάνουν 10 φορές περισσότερα από τις παράνομες χρηματοδοτικές ροές από αυτό που παραλαμβάνουν σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Ξέρω ότι η Eurodata έκανε μία αξιολόγηση και θα ήθελα να μας πείτε ποια ποσά ανακαλύψατε στην αξιολόγησή σας. Και έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των φορολογικών καθεστώτων τους επί των αναπτυσσομένων χωρών. Δηλαδή να μας πείτε σαφώς ότι για κάποια δισεκατομμύρια που αντλεί η Ολλανδία από το φορολογικό της καθεστώς, ε, σε τι απώλεια οδηγεί αυτό τις αναπτυσσόμενες χώρες. και ποια στοιχεία θεωρείται σημαντικά για να βοηθήσουμε καλύτερα αναπτυσσόμενες χώρες να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους, το fair share, το δίκαιο μερίδιό τους όσον αφορά τους πόρους τους. Ευχαριστώ Εύα για αυτή την παρέμβαση, την πολύγλωση. Καταλάβαμε πολύ καλά την ερώτηση. Για το EFDD, ο Μάρκο Τζάνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία που είναι παρούσα και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνει η οργάνωσή της, στην οποία ανήκει. Την καλώ λοιπόν να, να, να πιέζει το ώστε οι πολιτικοί να λαμβάνουν υπόψη τα τεράστια προβλήματα υπάρχουν, όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το σημερινό θέμα και εγώ όπως και ο Φάμπιο ενδιαφερόμαστε να ξέρουν ποια είναι η άποψή σα για, για τη δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάνω απ' όλα, αν αυτή η διαφάνεια, αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών είναι πραγματικά ο μηχανής Θεός, αυτός που θα λύσει όλα τα προβλήματα της φοροδιαφυγής, είναι απλώς ένα μικρό, ένα ελάχιστο βήμα μια μικρή βάση από την οποία ξεκινήσουμε και επιμένω επί της ερωτήσεως που έκανα προς τον γερουσιαστή Μόντι. Ίσως ένα σημείο επί τον οποίο επικεντρωνόμαστε πολύ λίγο. Το τραπεζικό σύστημα, επαναλαμβάνω, όλες οι χρηματοδοτικές συναλλαγές, οι νόμιμες ή οι μη νόμιμες περνούν από το χρηματοδοτικό σύστημα. Σήμερα δεν επιτρέπεται στην φορολογική αρχή να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίε. Πρώτη διαφάνεια πρέπει να επικρατήσει εκεί. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τι συναλλαγέ και το τραπεζικό σύστημα. Από αυτή την άποψη θα ήταν πολύ πιο εύκολο να κινηθούμε γιατί έχει την πολιτική δύναμη και τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσει τις χώρες και τις τράπεζες που δεν δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Παραδείγματο χάρη δεν δείχνουν ή αποσύρουν την αδειοδότηση από μια τράπεζα ή όμιλο τραπεζών που δεν συμμορφώνεται. Θα ήταν ένα μέτρο απλούστατο, χρήσιμο και αποτελεσματικό. Τώρα όσον αφορά ένα άλλο είδος επενδύσεων. Πολύ συχνά ε, γίνονται λίγες επενδύσεις. Η λιτότητα δημιούργησε περικοπές και, ε, ε, και λειτουργούν λίγο τα συστήματα συλλογής πληροφοριών και πληροφορική για να γίνει για να δούμε πώς υπάρχει διαφυγή από τον ΦΠΑ θα έπρεπε να υπάρχει ένα πραγματικό μητρό, ευρωπαϊκό μητρό των επιχειρήσεων πληροφορίε ομοιόμορφε να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ για να καταπολεμήσουμε τη διαφυγή από το ΦΠΑ. Τώρα, όσον αφορά τι τρίτε χώρε, ε, πιστεύω ότι θα ήταν δυνατόν, πιστεύω ότι ήταν δυνατόν να επιληθούν τα προβλήματα με τι τρίτες χώρε και τι αναπτυσσόμενες χώρε όταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταφέρνουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα μεταξύ μας με ένα συντονισμό πολιτικό με ένα συντονισμό μεταξύ χωρών πολύ ισχυροτέρων σε διεθνή βήματα και στον όσα από ότι είναι αναπτυσσόμενος. Ευχαριστώ. Κυρία Ρίντινγκ, έχετε το λόγο αν θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, αν μπορείτε να είστε σύντομοι σας παρακαλώ. Ναι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε συντομία στα πολλά ερωτήματα. Καταρχάς, αν έχουν γίνει αρκετά ήταν ένα ερώτημα. Αναφέρθηκαν διάφορα ζητήματα σήμερα, για παράδειγμα η ομάδα ε, για τον ε, κώδικα. Εμείς προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους θεσμούς και πρέπει να σας πω ότι αυτή η ομάδα επαφής για τον κώδικα, κώδικας, έτσι τους αρέσει να αυτό αποκαλούνται, ε, συνέρχονται μυστικά και δεν μας επιτρέπουν να μάθουμε τι συζητάνε. Έκανα μια παρουσίαση PowerPoint πριν από κάποιο καιρό και όλες οι επιζήμεις, λέει, οι φορολογικές πρακτικές στην Ευρώπη ε, δεν υπάρχουν πλέον, ε, έχουν εξαλειφθεί, αλλά αν δει κανείς αυτό το PowerPoint ε, θα δει ότι μάλλον είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα αυτά που γράφει, άρα ανησυχώ με αυτό το contact group και επειδή δεν ξέρω τι κάνουν δεν μπορώ και να σχολιάσω τι κάνουν. Σε ό,τι αφορά το δέσμο μέτρων για τη διαφάνεια που ε, προτείνει η Κομισιόν. Υπήρξε ένα πρώτο τέτοιο πακέτο διαφάνεια στην Άνοιξη και τώρα περιμένουμε το δεύτερο. Αλλά το εαρινό πακέτο δεν νομίζω ότι βοήθησε κανέναν, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε εμείς ανταποκρινόμαστε με μια δεσμέτρο για τη διαφάνεια. Το προφανές ερώτημα είναι διαφάνεια. Ποια είναι η νέα πληροφορία ε, που θα μπορεί να δει γνώμη. Και η απάντηση είναι καμία. Διότι ουσιαστικά προσδιορίζουμε τον όρο διαφάνεια. Διαφάνεια δεν σημαίνει κάτι που μπορεί να το δει ο κόσμο, αλλά σημαίνει πράγματα τα οποία κάποιε φορολογικέ δίκε και όχι όλε, ορισμένε φορολογικέ δίκε θα μπορούν να βλέπουν. Δεν βοηθάει αυτό το παιχνίδι. Αυξάνει την έλλειψη εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι ακριβής η επικοινωνία σε ό,τι αφορά αυτές τις δέσμες μέτρων, η ανταλλαγή αυτών των φορικών αποφάσεων τύπου tax ruling είναι το ελάχιστο βήμα και δεν θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, ό,τι αφορά τον ΩΣΑ και ΩΣΑ, έκανε μια ανακοίνωση τύπου πέρσι λέγοντας ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα για προς τα προς διαφάνεια. Ενώ ήταν σοχαριστικά αυτά που γράφανε, ότι όλες οι εκθέσει αναχώρα πρέπει να είναι πιστευτικές. Αυτό λέγανε σε αυτή την ε, εκθεσή. Ένα πολύ μεγάλο βήμα που έγινε προ τα εμπρό έγινε χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οδηγία Περικεφαλαικών Απαιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δημόσια αναφορά αναχώρα για τι τράπεζε. Παίρνουμε τι πληροφορίε για τι τράπεζε και εφαρμόζεται τώρα αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Τα κρατη πάνε στον ΩΣΑ και να υιοθετήσουν μια σύσταση η οποία θα λέει ότι οι πληροφορίες αυτές τώρα θα πρέπει να γίνουν εμπιστευτικέ ή να πούνε ε, ότι αυτό θα βοηθήσει και τη διαφάνεια. Λοιπόν, ας αρχίσουμε ε, να είμαστε ειλικρινεί και πραγματικά ε, για πράγματα τα οποία είναι εμπιστευτικά να μην μιλάμε για διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τα θέματα των αναπτυσσομένων χωρών, προσπαθούμε πράγματι να εκτιμήσουμε τις απώλειες και υπάρχουν ε, διάφορα νούμερα. Αλλά υπάρχει πλήρης έλλειψη στοιχείων, δεδομένων. Και εδώ έρχομαι σε αυτή τη, το, το country by country reporting, που κάποιοι θεωρούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Ουσιαστικά πολύ βασικά ερωτήματα τίθεται. Δηλαδή, η Coca-Cola πόσο πληρώνει, ε, πόσους φόρους πληρώνει στη Δανία για παράδειγμα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πόσες πόσους υπαλλήλους έχει, τι τζίρο έχει. Αυτό που θέλουμε να δούμε τι είναι, είναι ποια είναι η οικονομική δραστηριότητα της εταιρεία και να τη συγκρίνουμε με τους φόρους που καταβάλει. Και μετά βλέπουμε τις χώρες που είναι φορολογική παράδειση και τι πληρώνει εκεί, ε, τι κάνει η Coca-Cola ή τι κάνει η McDonald's, ε, πόσους υπαλλήλους απασχολούν και τι φόρους πληρώνουν. Δεν είναι πιστευτικά αυτά τα στοιχεία. Για όλες τις εθνικές εταιρείες Πράγματι, δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Είναι δημόσια, δεν μπορούν να κρυφθούν πίσω από διασυνοριακέ διευθετήσει και διακανονισμού. Δεν μπορούν να κρύψουν τα νούμερα αυτά. Είναι διαθέσιμα αυτά τα νούμερα. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να είναι δημοσιοποιημένε όλε οι φορολογικές πληροφορίε, γιατί το ίδιο ισχύει και για τους ιδιώτες. Δεν λέμε ότι όλα τα στοιχεία που πρέπει να είναι ε, δημόσια, αλλά εδώ μιλάμε για το τι κάνουν οι πολυεθνικές. Δεν έχω ακούσει ούτε ένα λογικό επιχείρημα γιατί να πρέπει να είναι όλα μυστικά και απόρριτα. Και έρχομαι τώρα στο, στην προσπάθεια να υπολογίσουμε τις απόλυσεις στις αρψόμενες χώρες. Πολύ λίγα γνωρίζουμε για το τι κάνουν σε αναψώμενες χώρες οι πολυεθνικές. Ε, πόσα χρήματα βγάζουν και αυτό ισχύει για όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Αυτό που βλέπουμε ε, είναι απλά προσπάθειες. Εμείς κάνουμε προσπάθειες και έχουμε κάποια νούμερα που βλέπουμε από αυτά ότι τουλάχιστον το λιγότερο ε, είναι ίσο με την απτυξιακή βοήθεια το ποσό αυτό της και σίγουρα είναι και πολύ πιο σημαντικό σε πάση περιπτώσει. Τώρα για, τις, για τα Ηνωμένα Έθνη, τι μπορούμε να κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κάνουμε. σω θα ήταν ένα δώρο στη συζήτηση αυτή. Το να μην είμαστε κλεισμένοι, κλειδωμένοι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να μπει στη μαύρη λίστα ούτε η Ολλανδία ούτε το Λουξεμβούργο, γιατί είναι κράτη-μέλη τη Ένωση. Άρα, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η διαδικασία να μπουν σε μαύρη λίστα κάποιες χώρες, είχε ως αποτέλεσμα να μπουν σε κάποιες τυχές ε, μαύρες λίστες κάποιες χώρες αναπτυσσόμενες, ενώ το προφανές πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Ένωση πέρασε παρατήρητο. Άρα οι διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, ώστε να συζητήσουμε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ εσωτερικά στην οικογένεια της Ένωσης, αλλά σε ένα άλλο πλαίσιο θα ήταν κάτι ευκταίο ώστε να μην είναι το Λουξεμβούργο μια ειδική χώρα κατά κάποιο τρόπο που δεν μπορεί να συζητηθεί. Θα ήταν κάτι τέτοιο αναζωογονητικό λοιπόν. Βέβαια είναι δύσκολο να γίνουν τέτοιου είδου ε, διεθνεί διαπραγματεύσει. Είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί όμω στο παρελθόν. Ότι δηλαδή όταν αρχίζει μια χώρα να χάνει δισεκατομμύρια ευρώ, όπω συμβαίνει, αρχίζει να είναι πρόθυμη τι πολυεθνικέ επιχειρήσει να τι εκδιώξει από την επικράτειά τη να πει σε μια πολυεθνική δεν θέλουμε να κάνεις ε, δουλειές εδώ, όπως είδαμε με τους γενετικούς ε, πόρους, αν δεν τηρούνται κάποιοι κανόνες. Άρα θεωρώ ότι φτάνουμε στη φάση που αυτό ε, το βλέπουμε ως ρεαλιστική δυνατότητα. Μόνο η Κίνα και η Βραζιλία έχουν φορολογικά συστήματα που είναι δύσκολα για τις πολυεθνικές. Αυτό θα οδηγήσει σε διπλή φορολόγηση και δεν ξέρω αν θα λύσει το πρόβλημα γιατί δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Πάντως κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπιστούν τις οικονομίες τους και νομίζω ότι θα βλέπουμε όλο και περισσότερες μονομερείς ενέργειες. Το φορολογικό σύστημα αυτό δεν θα είναι από κανέναν ε, επιθυμητό, αλλά θα υποχρέωσει και τις πολυεθνικές να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν γίνονται αυτά τα σκάνδαλα. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή απόπειρα ε, να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά μπορώ να σα πω ότι οι εκτιμόμενε απώλειες ε, των εψωμένων χωρών ε, δύσκολα και με πολλού τρόπου μπορούν να μετρηθούν, αλλά όπω και αν τι μετρήσαμε φτάσαμε πάντα σε πολύ ψηλά νούμερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα η μαρτυρία σα. Είναι σαφέ ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο θετικό στόχο που θέλουμε όλοι αν δεν έχουμε μια πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, των stakeholders όπως λέμε, και όλων όσων αποκάλυψαν, μέτρησαν το πρόβλημα και ασκούν πίεση και ε, κρατάνε και συγκρούσει την κοινή γνώμη, σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Πρόοδος όμως υπάρχει. Χρειάστηκε να έχουμε αυτή τη δημοσιονομική κρίση, ώστε σε επίπεδο G20, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή, να αποφασιστούν ε, κάποιες γενικές κατευθύνσεις οι οποίε υλοποιούνται παντού στον κόσμο. Dot Frank στι ΗΠΑ. Πολιτείες, έχουμε 20-30 ε, κανονισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι τέλεια βέβαια τα πράγματα, αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα, έχουμε και το τραπεζικό απόρριτο. Μετά από προσπάθειες ετών ήρθε ε, το τραπεζικό απόρριτο και η σύμβαση φάκτα είχε το ρόλο της. Και ένα από τα πιο σημαντικά όπλα, όπως επιβεβαιώσαμε και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, ε, όπως επιβεβαιώσαμε στις ε, αποστολές και στις οποίες διοργανώσαμε σε κάποια κράτη-μέλη, είναι ότι κανένα από αυτά τα κράτη δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο να χάσει την καλή του φήμη. Από τη στιγμή που ενημερώνει την κοινή γνώμη και όλος ο πλανήτης και όλοι οι οικονομικοί χρηματοπιστωτικοί παράγοντες ε, είναι ενήμεροι, μια χώρα ανεξάρτητο μεγέθου που θέλει να προσελκύσει επενδυτέ και θέλει να είναι χρηματοπιστωτικό κόμμος, δεν μπορεί να είναι το μαύρο πρόβατο του συστήματο. Αν είναι όλα τα πρόβατα μαύρα σε ένα σύστημα, αν σε ένα σύστημα όλοι δεν ε, μπορούμε να ξέρουμε τι χρώμα τέλο πάντων έχουν τα πρόβατα, ίσως να μπορεί να περάσει αυτό. Αλλά όταν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να αποκαλύπτουμε το χρώμα του προβάτου, τα πράγματα εξελίσσονται. Έστω και με βράδυς ρυθμού, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίντινγκ. toute la de saluer votre intervention et sans transition. Λοιπόν, θα δώσω παρευθύ το λόγο στον τελευταίο ομιλητή μας, στα πλαίσια της ακροάσεως μας, διότι τα άλλα μέλη είχαν προβλήματα ανεξαρτήτως θέλησής Ο κ. Αντουάν έχει το λόγο. Κύριε Ντελτούρ, έχετε περίπου ένα πεντάλεπτο, θα παρουσιάσετε την θέση σας και μετά, αν έχει την καλοσύνη, θα απαντήσετε στις ερωτήσεις, τις διάφορες που θα τεθούν. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ούτε την προέλευση της Επιτροπής, ούτε το στόχο και το πνεύμα των εργασιών μας. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Θα ήθελα να διαβάσω ένα κείμενο και προέβλεψα ένα δέκα λεπτά. Ζητώ εκ των προτέρων, λοιπόν, συγγνώμη. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή για τα φορολογικά που με προσεκάλεσε. Δεν θέλω να επεκταθώ μακρόν στην παρέμβασή μου για τις αποκαλύψεις LuxLeaks, γιατί γνωρίζετε τις γενικές γραμμές νομίζω εργάστηκα σε ένα μελαγό γραφείο ελέγχου στο Λουξεμβούργο που ανακάλυψα την ε, τακτική του tax ruling που είναι κάτι θεμητό λόγω της νομικής ασφαλείας, ασφαλείας δικαίου που επιφέρει το περιεχόμενο κάποιου εγγράφου με συνεκλώνηση. Αυτές, αυτά τα σκάνδαλα περιγράφουν λεπτομερώς σε ένα φορολογικό σχεδιασμό ε, πολύ επιθετικό σε επίπεδο βιομηχανικό Λοιπόν, οι πρακτικέ εφαρμόζονται από πολλέ πολυεθνικέ και είναι επιζήμιε και καταλήγουν σε περιπτώσει όπου υπάρχει σχεδόν έλλειψη φορολόγηση, μια κατάσταση που θεωρώ ο πολίτη ότι είναι απαράδεκτη. Όχι μόνο οι επιχειρήσει εκμεταλλεύονται τα κενά των εθνικών νομοθεσιών, αλλά αρκετά κράτη-μέλη αναπτύσσουν πραγματικέ στρατηγικέ προώθηση φορολογικών καθεστώτων που θέλουν να συλλάβουν τη φορολογική βάση των γειτόνων. Από την άποψή μου, αυτό που δημιουργεί πρόβλημα δεν είναι τόσο η πρακτική του tax ruling, αυτό τεχνικέ Αποφυγή των φόρων περιγράφει το έγγραφο. Και εκλήθησαν από τον ελεγκτή, από τους ελεγκτικούς φορέ. Α, πιο αργά για τις διερμηνείς, λέει ο μιλητής. Εκλήθην από τον έλεγχο όσον αφορά την κυκλοφορία των εγγράφων να εξετάσω διότι υπήρχαν και προβλήματα φορολογικών διαφορών από τους διαφόρους φορείς αν τελικά απεκαλύπτεται από ανταγωνιστή κάποιο έγγραφο ή από τις ξένες φορολογικές αρχές τέλος του 2010 πλην παρετηθώ, αποφάσισα να αντιγράψω αρκετές εκατοντάδες tax ruling που ήταν απλώς ένα κομμάτι το, της εφαρμογής του μέτρου. Ποτέ δεν είχα πρόθεση να δημοσιοποιήσω όλα αυτά τα έγγραφα, όμως τα διαβίβασα σε ένα δημοσιογράφο με στόχο να ευνοήσω δημόσια συζήτηση από αυτού. Ε, πιστεύω ότι τα κίνητρα είναι πολύ κοντά σε εκείνα που κινητοποίησαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει αυτή την ειδική επιτροπή, διότι αν ερευνάτε αυτή τις, ε, αυτά τα τις φορολογικές πρακτικές το κάνετε διότι θεωρείτε όπως και εγώ ότι παρά την υποτιθέμενη νομινότητά δεν είναι εντελώς ε, νόμιμες. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η ύπαρξη της Επιτροπής ΤΑΞ ε, αντιπροσωπεύει μια πλευρά, μια αναγνώριση του δημοσίου ενδιαφέροντος για τα έγγραφα που συνέχισα να βγάζω από τη σκιά και από την άλλη πλευρά σαν μια δικαιολόγηση των κινδύνων που ανέλαβα εγώ όπως γνωρίζετε, πατέρασα το αντικείμενο ε, δικαστικών ε, ε, διώξεων που μου δείξαν να δικαινήσω μια ποινή πενταετή και να πληρώσω πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Το Λουξεμβούργο επιβεβαιώνει ότι ήθελε να συνεργαστεί και να προωθήσει την φορολογική διαφάνεια, αλλά θεωρεί ότι είναι η αυτή, οι διώξει αυτές είναι νόμιμες. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις εκείνοι που, ε, που ειδοποιούν και η ενυπέρωση του κοινού είναι ένα κινητήρα ε, για μια πολιτική δράση. Διάφορες προσωπικότητες δήλωσαν στον τύπο ότι είναι πολιτικά άδικο και ηθικά ε, ασύλληπτο ότι ένα διάβημα του πολίτου προς το κοινό όφελος ε, του ευρωπαϊκού λαού αποτελεί αντικείμενο δικαστικών διώξεων. Λοιπόν, θεώρησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα νομικό πλαίσιο που να προστατεύει εκείνους που δίνουν του πληροφοριοδότε και να υπάρχει μια ευρεία, ένας ευρύς ορισμός όπως συμβουλεύει και το, ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Με έχουν κατηγορήσει ε, μάλλον ότι το σχέδιο οδηγίας πιστεύω ότι ε, είναι απειλή για τους δημοσιογράφους και για τους πληροφοριοδότες και ιδιωτικά συμφέροντα θα επικρατήσουν έτσι των δημοσίων συμφερόντων. Εξάλλου, κάποιε αναλύσει προσωπικέ έχω να μοιραστώ μαζί σα όσον αφορά τα φορολογικά θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή τη και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω ερωτήσει σα. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία μου στο Λουξεμβούργο δεν είναι περίπου παρά μόνο διετή όσον ε, ελεγκτή ε, και δεν με κάνει ειδικό όσον αφορά τα φορολογικά θέματα, αλλά οι απόψει μου εκπροσωπούν μόνο αυτέ ενό πολίτου απλού. Και γι' αυτό δράτω με τι ευκαιρίε να προβώ σε ανταλλαγέ απόψεων με εσά, να σα πω εντάξει πόσο σημαντικό είναι η Επιτροπή Τάξ να είναι μαχητική και τολμηρή έναντι των εμποδίων που θα αντιμετωπίσει και θα αναφερθώ σε δύο σημεία εντάχει. Καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι μια επιτροπή εξεταστική που τη θέλουν πάνω από το 1 τέταρτο των Ευρωβουλευτών θα επέτρεπε να απαιτηθούν έγγραφα και να προσκληθούν άτομα. Διαπιστώνουμε σήμερα ότι ο αριθμός των προσκλήσεών σας απερίφθησαν, το διαπιστώνουμε σήμερα και κάποια κράτη-μέλη επιτρέπουν στον εαυτό τους να μην δώσουν όλες τις πληροφορίες που τους ζητάτε. Γνωρίζουν την υποφασιστικότητα κάποιων μελών αυτής της ειδική επιτροπής για να κινηθούν οι πολιτικές γραμμές και να τιμηθεί η φιλόδοξη εντολή Ελπίζω σήμερα ότι πιο ε, και από εσά ε, έχουν επίγνωση των διακυβευμάτων αυτών για τα φορολογικά στην Ευρώπη. Το δεύτερο σημείο μου αφορά την φορολογική δικαιοσύνη ή μάλλον τη φορολογική αδικία των οποίων, ε, το, το, το, οποίο το εύρος βλέπουν και διαπιστώνουν διάφοροι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είναι τίποτα άλλο από το να διατηρηθεί ε, το η συνδετικό συστός των δημοκρατιών μας και η κοινωνική σύμβαση. Πολλοί ε, ανησυχούν για την ελκυστικότητα της Ευρώπης. Να τηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα των κρατών μελών. Είναι με στρατηγική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες και οδήγησε τελικά στην παρούσα κατάσταση. Σύμφωνα με τον Τόμας Πικετή, ο, φόρος ε, των εταιριών απειλείται να εξαφανιστεί μέχρι σε, μέσα 10-20 χρόνια. Αυτή η Επιτροπή την υποστήριξη του κοινού και άλλων πολιτικών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι ένα σημείο ε, καμπής για να εξεταστούν οι διάφορες στοιχείες που απαιτείται. Λοιπόν, τα συμφέροντα τα διάφορα εμποδίου στη φορολογική διαφάνεια, ε, γίνονται πιο επαχθείς διαδικασίες και αναπτύσσεται ε, η, συζήτη, η περιπλοκότητα των τεχνικών συζητήσεων υπέρ κάποιων ε, ειδικών για τα φορολογικά σε ένα πλαίσιο όπου διποφέρουν οι ευρωπαϊκοί λαοί λόγω περικοπών θα ήταν παρακειδεμένο οι θεσμοί, ε, οι θεσμοί να συμβιβαστούν όσον αφορά το θέμα αυτό το φορολογικό για να προστατεύσουν κάποια συμφέροντα. Τέλο, η ανάπτυξη τη απασχόληση δεν είναι ένα καλό λόγο για να περτηθούμε από το πολιτικό θάρρο όσον αφορά τα φορολογικά θέματα. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει εν γέννη δεν έχουν πρόσβαση στα περίπλοκα σχήματα που τα έχουν οι μεγάλε επιχειρήσει των πολλών χωρών. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει υπόκειται σε προφανή στρέβλωση ενώ ε, δημιουργούν πάρα πολλοί θέσει εργασίες. Επιτρέψτε μου να κλείσω αντιστρέφοντα του κανόνε, θέτοντα ένα ερώτημα, αυτό του ερώτημα ενό ανησύχου Ευρωπαίου πολίτε. Χωρί τα φορολογικά έσοδα των επιχειρήσεων, ποια θα είναι η φιλοδοξία των δημοσίων πολιτικών στο μέλλον. Θα έχει νόημα να εκλέγουμε πολιτικού υπευθύνου που δεν έχουν τίποτα παρά μόνο μια πολύ ε, ισχνή εξουσία εσείς θα πρέπει να ρυθμίζετε τελικά τις πολιτικές ε, και οικονομικές εξουσίες όταν αντιβαίνουν ε, στα συμφέροντα του κοινού καλού. Ελπίζω ότι αυτή η διαπίστωση είναι κοινή για σας και ότι αυτή η Επιτροπή θα μπορεί τάχιστα να ε, καταλήξει σε κάποια αποτελέσματα υποδειγματικά και φιλόδοξα. Λοιπόν, θα κάνουμε κάποια σχόλια και μετά θα δώσουμε το λόγο στους διαφόρους εισηγητές. Γιατί δημιουργήσαμε μια, γιατί δημιουργήσαμε μια εξεταστική επιτροπή. Το θέμα που συζητάμε σήμερα δεν είναι αρμοδιότητα κοινοτική, γι' αυτό δημιουργήσαμε έρευνα, αλλά εξεταστική. Και νομικά δεν είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί θέματος αρμοδιότητας ευρωπαϊκής, ε, όπως είναι η κοινωνική πολιτική, η πολιτική συνοχής, η προστασία των καταναλωτών, μπορώ να δημιουργήσω μια ερευνητική επιτροπή, μπορώ να συγκαλέσω μια τέτοια, είτε υπαλλήλου να χρησιμοποιήσω πολιτικού ω μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών ή κρατών μελών που εφαρμόζουν τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Η φορολογία είναι αρμοδιότητα εθνική αποκλειστικά. Δεν μπορώ να συγκαλέσω με τέτοια επιτροπή, δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν να έρθει. Αλλά μπορώ να καλέσω. Μπορώ να ε, κάνω να έρθουν μέσω προσκλήσεως θέσατε την περίπτωση κάποιων επιχειρήσεων που καλέσαμε οι οποίες δεν ήρθαν πολύ καλά αυτές που δεν έρχονται τελικά δηλώνουν ενοχή εκείνες που δεν έρχουν δεν τολμούν να έρθουν να εξηγηθούν μπροστά μας και παρατηρώ και δράτω με τις ευκαιρίες του σχολείου που κάνατε, διότι υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωση εδώ δημόσια συνεδρίαση. Παρατηρώ λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις στις οποίες είπαμε ότι θα θέλαμε να έρθουν προς ενημέρωση, μάλλον να έρθουν σε επαφή με τους υπουργούς τους αρμόδιους για τη φορολογία στις χώρες. Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, με την κυβέρνηση, με μέλη της κυβερνήσεως, με την Επιτροπή Οικονομικών του Εθνικού Κοινοβουλίου που παρακολουθεί το όλο πρόβλημα να συναντήσουμε τους ντόπιου stakeholders εμπλεκόμενους, τους μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τους πληροφοριοδότες, τους whistleblowers, τους δημοσιογράφους. Να συναντηθούμε επίσης με εκπροσώπους των Big Four, των μεγάλων ε, συμβουλευτικών φορέων. Όλοι τελικά δέχτηκαν και οι ελβετικές αρχές. Μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δέχτηκε και άλλες ε, κυβερνήσεις με τις οποίες είμαστε επαφή τώρα, θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο αργότερα, θα κινηθούν παρομοίως και είμαι πεπισμένος ότι κάποιοι από εκείνους που εν πρώτης απάντησαν αρνητικά τελικά θα οδηγηθούν στο να αλλάξουν γνώμη. Βλέπω ότι πολλές μεγάλες πολυεθνικές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους από τούδε και στο εξής να έχουν φορολογική έδρα σε όλες τις χώρες που ασκούν δραστηριότητα και να διοργανώσουν μια ημερίδα ανοιχτών θυρών. Κάλεσα σήμερα τις επικεφαλής των πολυεθνικών, ώστε αυτή η ημερίδα των ανοιχτών θυρών ε, εν μέρη να γίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσία Εάν το δεχτούν αυτό θα μπορέσει να διεξαχθεί μια συζήτηση που θα οδηγήσει στους ανταγωνιστές της πολυεθνικής εταιρείας να κάνουν παρόμοια πράγματα και αν αρνηθούν αυτό θα μειώσει στο μηδέν ε, τη βούλησή τους που προέβαλαν να σεβαστούν τη φορολογική δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Θα φανούν ότι είναι απλώς λόγια αυτά. Έχουμε πολύ ανίσχυρα νομικά μέσα, αλλά τα πολιτικά μας μέσα είναι πάρα πολύ ισχυρά αν κινηθούμε στο πνεύμα που θα μας διαπνέει και στα πλαίσια των πληροφοριών που μας δώσατε και των απαντήσεων που θα δώσετε. Πρώτα απ' όλα στους εισηγητές και μετά στα μέλη μας. Καταρχάς, η Ελίζα Φερέρα έχει το λόγο. Merci bien d'être parmi nous. Euh, Ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν ε, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι αν δεν είχαν υπάρξει τα Lux Leaks. Παρότι είχε υπάρξει μεγάλο πρόβλημα ε, με την υποβάθμιση της δικαιοσύνης και φορολογική αδικία, σας ευχαριστούμε πιστεύω και που βγάλατε στο φως ε, αυτό που ήταν καλά κρυμμένο. Τρία ερωτήματα. Πρώτο, σε πολλές ανακοινώσεις και τα λοιπά έχετε πει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν επίθεση ε, στην εταιρεία, αλλά ο μηχανισμός ήταν αυτό που θέλατε να εκθέσετε, να αποκαλύψετε. Τώρα λοιπόν που έχουμε τα εργαλεία και προσπαθούμε τέλο πάντων να προσπαθούμε να βρούμε τα εργαλεία για να κλείσουμε να σπάσουμε αυτούς τους μηχανισμούς με τη φορολογική βάση και τα φορολογικά είσοδα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να αλλάξει πραγματικά η κατάσταση. Δεύτερο ερώτημα. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την προστασία των πληροφοριοδοτών. Στο Λουξεμβούργο πραγματικά ε, όταν πήγαμε, αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στη δική σας περίπτωση και μας απάντησαν ότι τα προβλήματα που θα είχατε απέρεαν από τις διατάξεις του αστικού δικαίου. Γιατί ήταν ε, η σύμβαση που είχατε με την εταιρεία. Και αυτή είναι στην ε, ρίζα του προβλήματος. Διότι είχατε την υποχρέωση ψευτικότητας της εχεμήθειας αναλάβει. Δεν είναι θέμα λοιπόν ακριβώς ε, πληροφοριδιωτών. Αλλά τι συμβάσει έχετε υπογράψει. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να γίνεται με μεμονωμένες συμβάσεις ή συνολικά να υπάρχει μια προστασία των πληροφοριδιωτών. Τρίτο ερώτημα. Και αυτό σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο και με ε, την ανησυχία μου. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων εντός επιχειρήσεων, όπως ο Κούπερς άλλων ή άλλων που είναι σύμβουλοι σε θέματα φορολογικά. Και εδώ βλέπουμε ότι ε, στηρίζουν, υπάρχουν τεχνικές συμβουλές ε, και εδώ ακόμη και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν και σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι πολύπλοκο. Πώς μπορούμε εμείς να εγγυηθούμε το ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν θα παίζουν σε όλα τα ταμπλό. Και με τις επιχειρήσεις και με που θέλουν ουσιαστικά να περιορίσουν τις κινήσεις σε αυτό το φορολογικό ανταγωνισμό. Και αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που δεν είχατε το χρόνο στην πρώτη σας παρέμβαση, ευχαριστώ να σας ακούσουμε. Merci Elisa. Ευχαριστώ, Michael Teurer. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Δελτούρ, σας ευχαριστώ πολύ που ε, ήσασταν πρόθυμος να έρθετε στην Επιτροπή μας και για μένα ως εισηγητή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είστε εκ των προσώπων εκείνων που είναι γνωστά ως καταγγέλλοντες, ως whistleblower, που επέτρεψαν με τις καταγγελίες τους την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις οδήγησαν στην αποκάλυψη ε, θεμάτων σε διαστάσεις που πολλοί δεν φαντάζονταν. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε περισσότερο ποια εντύπωση είχατε εσείς ως συνεργάτης μιας φύρμας συμβούλων. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ είναι το εξής. Οι διάφορες εταιρείες συμβούλων προσεγγίζουν τις χώρες μέλη και ζητούν συγκεκριμένες φορολογικές ρυθμίσεις ή συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή εμφανίζουν, προτείνουν τις ε, φορολογικές αυτές ρυθμίσεις οι διάφορες χώρες μέλη ή οι σύμβουλοι που έχουν ειδικέ γνώσεις προσεγγίζουν τις εταιρείε ή πρόκειται τελικά για ένα συνδυασμό όλων αυτών των πτυχών. Δεύτερη ερώτηση, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε για λόγους νομικούς. Από τη δική σας υποκειμενική άποψη, πώς γινόντουσαν οι χειρισμοί μέσα σε αυτή την επιχείρηση. Διάβασα συνέντευξή σας στον τύπο, που λέτε, όπου λέτε ότι όχι μόνο ο εργοδικός σας εργοδότης, αλλά και άλλοι πράττουν παρόμοια. Υφίσταται δηλαδή κάποια πίεση, υπάρχει κάποια πίεση η οποία δίνει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες ή οι ίδιοι συνεργάτες καταλήγουν με δική τους πρωτοβουλία σε πρόταση κάποιων λύσεων που επιτρέπει στις ε, εταιρείε να μειώνουν πάρα πολύ τα φορολογικά τους ε, ε, έξοδα, τις φορολογήσεις τους. Και πότε εντοπίσατε παραβιάσεις δικαίου. Λάβατε υπόψη το ενδεχόμενο να καταγγείλετε τα πράγματα στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Δηλαδή, αντί να πάτε να βρείτε κάποιον δημοσιογράφο, σκεφτήκατε να πάτε στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα. Και αν το σκεφτήκατε, τι σας απέτρεψε από το να το πράξετε. Πού δηλαδή εντοπίζετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταγγέλλοντες. Γιατί δεν πηγαίνετε στις αρμόδιες αρχές. Εκεί που πήγαμε μας είπαν κατ' επανάληψη, μα υπάρχει η δυνατότητα να ε, απευθυνθούν οι καταγγέλλοντες στις αρμόδιες διοκτικές αρχές. Ορισμένοι βέβαια μας είπαν ότι έκαναν την προσπάθεια αυτή, δεν οδηγήθηκε όμως ε, η υπόθεση σε δίωξη κατά των επιχειρήσεων, αλλά σε δίωξη κατά των ίδιων των καταγγελόντων. Γι' αυτό και νομίζω ότι απαραίτητη είναι και η προστασία των δικαιωμάτων των ίδιων των καταγγελόντων. Ευχαριστώ. Νίτερ του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα που ήρθατε. Θα γνωρίζετε ότι πριν από λίγες ημέρες η Amazon είπε ότι θα εγκαταλείψει το φορολογικό της σύστημα του Λουξεμβούργου και θα αρχίσει να πληρώνει πραγματικούς φόρους. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Και βεβαίως μετά από την σημαντικότατη πίεση του κοινού. Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Ή ε, θεωρείτε ότι θα είναι πολύ περισμένο το εύρος αυτών των αντιδράσεων. Δεύτερον, διαφάνεια πολύ σημαντική για την βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας ε, των φόρων. Ως πρώην ελεγκτής, auditor, πού βρίσκεται ότι βρίσκονται τα όρια της διαφάνειας. Γιατί ταυτόχρονα μιλούμε για διαφάνεια. Τι είδους έγγραφα που να έχουν σχέση με τη φορολόγηση θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνονται προσβάσιμα στο κοινό και ποια έγγραφα θα πρέπει να εξυπηρετήσουν την καλύτερη φοροεισπρακτική ικανότητα των χωρών. Επίσης, δεν πρόκειται για επιχειρήσεις ή συμβούλους ή ε, λογιστές. Δεν είναι αυτοί δηλαδή που δημιούργησαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα προέρχεται από την περιπλοκότητα των φορολογικών ρυθμίσεων. Κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει τις φορολογικές ρυθμίσεις χωρίς την υποστήριξη ειδικών. Μας είπαν ορισμένοι ειδικοί ότι το καλύτερο θα ήταν να στοχεύσουν στην φορολόγηση των ιδιωτικών εισοδημάτων καθώς και της κατανάλωσης και να ξεχάσουν τον φόρο των επιχειρήσεων. Πώς το βλέπετε αυτό, γιατί μου φαίνεται αρκετά επαναστατική προσέγγιση. Merci, pour le groupe Ευχαριστώ, Αναλύς Ντότς, ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα, γιατί νομίζω Μου ότι δείξατε μεγάλο θάρρος. Και οι πράξεις σας οθούνται από μια ιδέα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Uh, να το πω καλύτερα στα αγγλικά ε, γιατί διευκολύνει. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και βεβαίως και τις προσωπικές συνέπειες που υποστήκατε. Ήταν πολύ θαραλέο το βήμα σας. Μάλλον τα πηγαίνατε πολύ καλά και είχατε μπροστά σας μια πολύ ελκυστική σταδιοδρομία και όμως τα καταλήψατε αυτά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Μίλησα τώρα για το σχέδιο οδηγίας για το επαχειρηματικό απόρριτο. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά γιατί θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να ε, αποδειχθεί προβληματικό για τους καταγγέλλοντες στο μέλλον. Δεύτερο, Προωθούνται κάποια μέτρα τώρα μέσα στην οδηγία κατάχρηση αγοράς στο δεύτερο επίπεδο για προστασία που θα παρέχεται στους καταγγέλλοντες όταν πρόκειται δηλαδή για insider trading. Και εκεί βλέπουμε ότι παρόλο που σημειώνεται αντίσταση από τις χώρες μέλη, είναι δυνατόν να επιβάλλουν τα μέτρα αυτά με διάφορους τρόπους σε διάφορες χώρες μέλη, αλλά και με σεβασμό των ε, νομικών περιστάσεων στις διάφορες χώρες μέλη. Ποιες είναι οι απόψεις σας και για ορισμένους από τους μηχανισμούς που μπορούν να επιβάλλουν τις προστασίες αυτές στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν έχετε κάποιες ιδέες σχετικά, Αντιλαμβάνω βέβαια ότι είναι περίπλοκο το θέμα που θίγω. Τέλος, έχουμε συζητήσει για κώδικες διοντολογίας για τους ε, φοροτεχνικούς συμβούλους και όταν μιλήσαμε και με τους μεγάλους τέσσερις μας είπαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεσμοθετήσουμε τίποτα γιατί υπάρχουν κώδικες διοντολογίας. Όμως η δική σας περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης αυτών των κωδίκων διοντολογίας και ότι επίσης αυτοί δεν επιβάλλονται ορθά. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν κάποιες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να σφίξουν λίγο τα πράγματα, να υπάρξει ένας κώδικας διοντολογίας, για παράδειγμα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή απαιτήσει που να εφαρμόζει διάφορες χώρες μέλη. Γιατί από την μαρτυρία σας που μόλι άκουσα, φαίνεται ότι αυτό που σας ζητείτε ήταν να κάνετε πράγματα τα οποία άγγιζαν τότε και αυτό αναγνωριζόταν μέσα στην επιχείρησή σας. Και αυτό βεβαίως αντίκειται στην άποψη των περισσότερων για το τι είναι διοντολογικά αποδεκτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Αντελίζ. Αυτή την τελευταία σας ερώτηση την έθεσα και στους εκπροσώπους των μεγάλων τεσσάρων και δεν μου απάντησαν. Βεβαίως θα εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο την δική σας ενδεχόμενη απάντηση. Φάβιο Ντεμάζη, Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ. Αλλά η σχέση μου με τον πρόεδρο είναι καλή, αλλά θα χρησιμοποιήσω λίγο από το χρόνο μου για να φέρω μια αντίρρηση. Θα υπήρχε χρόνος και θα υπήρχε και χώρος να δημιουργηθεί μια ερευνητική επιτροπή, διότι γνωρίζουμε ότι το και κοινοτικό δίκαιο παραβιάζεται εδώ και δεκαετίες. Μας τα είπαν αυτά και στις διάφορες επισκέψεις μας και θα ήταν δυνατόν και άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αντιδράσει. Θα μπορούσε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιδράσει. Δεν υπήρξε όμω η πολιτική βούληση. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Δεύτερο, ο Αλάν Λαμασούρ τόνισε ότι όσοι δεν προσέρχονται αναγνωρίζουν την ευθύνη του Ενδιαφέρομαι να μάθω αν θα προσέλθει ο κύριος Γιούνκερ με άλλα λόγια. Τώρα, ερωτήσεις προς κύριο Ντελ Τούρ, τον οποίο, τον οποίο ευχαριστώ που προσήλθε και βρίσκω σκανδαλώδες ότι ο κ. Γιούνκερ πίνει τον καφέ του στην, ε, εδώ κοντά στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ εσείς τελείτε υποδίωξη. Η οδηγία για την προστασία του επαγγελματικού απορρίτου χαρακτηρίζει την δυνατότητα των Ευρωπαϊκών Επιτροπών, ε, των ε, εταιριών, των εταιριών να μπορούν να διευρύνουν αυτό που θεωρούν ότι καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρριτο, μειώνοντας έτσι την προστασία των δικαιωμάτων των κατακελόντων. Πώς βλέπετε τώρα ε, την διαδικασία που κινείται εναντίον σας και που ως άλλος πόντιος πιλάτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νύπτει τα σχήρας της. Δεύτερο, θα ήθελα να μάθω εάν θα υποστηρίζατε στην ψηφοφορία για την οδηγία για, για τα δικαιώματα των μετόχων να συμπεριληφθεί και διάταξη για το country by country reporting, κάτι το οποίο φαίνεται να μην πρόκειται να γίνει μετά από επιθυμία ορισμένων πολιτικών ομάδων εντός του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Φάμπιο, θα επανέλθουμε. Ε, των διαφορών αυτών. Εννοώ με τον Πρασίνων. Μολύς Κοτκάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με κάθε σεβασμό να επανέλθω σε αυτό που είπατε προηγουμένως για το βαθμό των εξουσιών που έχουμε. Συμφωνώ ότι είναι πολιτικές οι εξουσίες και όχι νομικές. Η πολιτική επιρροή όμως εξαρτάται πολύ από το ποιος έρχεται, ποιος είναι μάρτυρας, και όταν οι επιχειρήσεις αποφάσαν να μας περιφρονήσουν, σαν Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσουμε, να αυξήσουμε τις εξουσίες μας, να τους απαιτήσουμε να έρθουν, να έχουμε δικαστική τέτοια εξουσία για να μπορούμε να καλούμε μάρτυρες. Αλλιώς πιστεύω ότι υπονομεύουμε την εξουσία μας και τη δύναμη να δράσουμε με τον τρόπο που απαιτείται. Προχωρώντας τον Αντουάν, λυπούμε, λοιπόν, βλέπω μόνο το πίσω μέσα του κεφαλιού σου, Αντουάν, τέλος πάντων, συγχαιρετώ. Καταρχάς, ευγνωμοσύνη και αλληλεγγύη εκφράζω προς εσένα για το θάρρος που έδειξες και καλώς ήρθες στην Επιτροπή σήμερα. Βέβαια, είμαστε σε γραφειοκρατική σύνθεση σήμερα, χωρίς εσένα θα συνέβαινε αυτό. Πολλές, ε, πολλούς πόρους έχουμε στη διάθεσή μας λόγω των δράσεών σου και σε ευχαριστώ για αυτό. Είναι σημαντικό να εστιαστούμε επακριβώ ε, όσον αφορά αυτά που έκανε στου καταγγέλων. Ποια είναι η εμπειρία σου. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάποιε προσωπικέ ερωτήσει, αν δεν σε πειράζει. Ενδιαφέρον το ταξίδι σου για κάποιον που εργαζόταν σαν ελεγκτή και να γίνει κάποιο που αποφάσισε να κινηθεί προ κοινόν όφελο και αντιμετωπίζει ποινική δίωξη, ποινικέ διώξει λόγω των πράξεων του. Δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση προφανώ. Μπορεί να εξηγήσει όμω πώ αισθάνεσαι. Διότι ελάχιστοι προφανώ κινούνται όπω εσύ. Πολλοί έχουν πληροφορίες για παρατυπίες, αλλά πολλοί λίγοι δρούν όπως εσύ. Πολλοί έχουν το θάρρος, μπορεί να μας πεις περισσότερα. Επί τεχνικής σε η ομάδα των Πρασίνων πρότεινε να δημιουργηθεί μια πύλη διαδικτυακή, ούτως ώστε οι καταγγέλλοντες να μας δίνουν πληροφορίες για το κοινό καλό, με πλήρη ασφάλεια και μυστικότητα. Δεν θα φοβούνται για νομικές κινήσεις εναντίον τους. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου είπε ότι υπάρχουν προβλήματα με αυτό και έχουμε πολύ λιγότερη ασφαλή. Έχουμε λοιπόν email με κάποια ρήτρα που αναφέρει περί, θέματα περί επαλλαγής υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Λοιπόν, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών για το κοινό καλό, τι μπορεί να μας πεις πάνω σε αυτό, τέλος. Μπορεί να μας πεις αν υπάρχει άλλος τρόπος που μπορούμε να στηρίξουμε και σε ένα και άλλους καταγγέλλοντες κάλυψα κάποια τεχνικά θέματα. Μπορείς να μας δώσει λεπτομέρειες για συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη μπορούμε να σου διαθέσουμε. Ας πούμε εγγύηση απασχόλησης, εσόδων ή κάποιες νομικές συμβουλές που μπορούμε να προσφέρουμε. Ευχαριστώ μόλι. Για το EFTD ο Μάρκο Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εν ονόματι όλων των Ιταλών, ειλικρινών Ιταλών και εκείνων που ψηφίζουν το κίνημα των πέντε αστέρων για αυτό που έκανε ο Αντώνιντε Λετούρ και για εκείνα που κατήγγειλε, διότι σήμερα με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε διεθνέ επίπεδο, το θέμα τη φοροδιαφυγής από πλευρά των πολυεθνικών είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργεί τέτοια στέβλωση του ανταγωνισμού που είναι απίστευτη και εμεί από πρώτο χέρι τα βλέπουμε όλα αυτά πηγαίνοντα στι διάφορε περιοχέ των χωρών πώ είναι απελπισμένο ο κόσμο και η κοινή γνώμη Πώ είναι με αυτό το παιδί με αυτό τον... και όχι με την πολιτική, με του πολιτικούς που μετά θα ψηφίσει η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπω είναι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δείχνοντα ότι δεν άκουσε τίποτα. Δεν άκουσε καθόλου τους πολίτες που από αυτή την πλευρά προσπαθούν να ανακαινήσουν τους θεσμούς οι πολίτες. Η απάντηση που λαμβάνεται μέσω αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης όσον αφορά την παλαιά πολιτική είναι η νέα πηγή των νέων κινημάτων και λυπούμε διότι τελικά πολλά νέα κινήματα οδηγούν σε ακραίες θέσεις που δεν οδηγούν σε αλλαγές σε θέσεις όπως είναι τα κινήματα της άκρας δεξιάς. Θε θα σας ρωτήσω, αισθάνεστε ως πολίτης αυτή την τοποθέτηση ήθελα να δώσω στη συζήτηση ότι εκπροσωπείστε από τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον άνθρωπο που σαν πρόεδρος της Ευρωομάδας επέβαλε στη λιτότητα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα και ταυτόχρονα δημιούργησε αυτό το σύστημα της φοροδιαφυγής σε μια χώρα μισό εκατομμυρίου κατοίκων με μια έκταση πολύ μικρή δημιουργώντας όλο αυτό το μηχανισμό επαφών με τα εξασφαλιστικών εταιριών πολυεθνικών τραπεζών ε, και χωρών που είναι ένοχες που δεν εφάρμοσαν σωστά τους κανόνες μεταξύ τους για να αποφευθεί η δημιουργία του συστήματος. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε μαζί σας και πάντα θα έχετε την ανοιχτή πόρτα του κινήματός μου για να καταγγέλλετε αυτού του είδους τις ε, πρακτικές. Ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο κύριος Δελτούρ. Ε, Πόσο χρόνο έχω στη θέση μου, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα ο πρόεδρος, όπως είπε και η κυρία Ρίντινγκ. Όπως μάλλον μπόρεσε η κυρία Ρίντινγκ μέσα σε 10 λεπτά να απαντήσει. Μάλιστα, θα προσπαθήσω και εγώ να περιουστώ σε λεπτό, στο βαθμό του δυνατού ή των δυνατοτήτων μου. Βασικά με τη σειρά της ερωτήσεις, αλλά είναι δύσκολο να είμαι ευσύνοπτος, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω. Πράγματι υπογράμμισα ότι οι πρακτικές που καταγγέλλω και εγώ είναι συστημικές. Και ήθελα να πω με αυτό ότι δεν θέλουμε να κατονομάσουμε και να καταγγείλουμε μόνο κάποιες εταιρείε ή κάποια κράτη όπως έγινε από τον τύπο και τα υπόλοιπα μέσα. Ποια θα ήταν η λύση τώρα απέναντι σε αυτό το συστημικό πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό άπτεται περισσότερο της ε, πολιτικής. Ε, υπάρχουν προτάσεις επιτάπητος. Ε, είπα στην πρώτη μου παρέμβαση ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός δεν βοηθάει να λυθούν τα προβλήματα. Και οι λύσεις περιφορολογικής αρμόνισης δηλαδή, όπως έχει ακουστεί, προβάλλονται ή αυτή η πρόταση για την ενοποιημένη βάση φορολογίας με βάση την πραγματικότητα και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η λύση πιστεύω ότι θα έβαζε ένα τέλος στην εκμετάλλευση όλων των τεχνικών κενών και αδυναμίων. Πρόεδρος, ε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή είστε ειδικό, λέτε ότι από τεχνικής πλευράς αυτή η λίστα ήταν εφικτή. Τι άποψη έχετε Εντάξει, υπάρχει το πολιτικό θέμα, αν θα γίνει όχι, αλλά δεν είμαι ειδικό, ε, λέει ο κύριο Ντελτούρ, ε, ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι ειδικό, γι' αυτό και δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειε ότι αυτά τα φορολογικά, γιατί εργάστηκα ω ελεγκτή για δύο χρόνια, όπω σα είπα, και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο ικανοί από εμένα. Ο Ρίσα θα ήταν. Ε, ο Ρίσαρτ Μέρφυ, συγγνώμη, θα ήταν πολύ καλύτερα να ήταν εδώ, δεν μπόρεσε να έρθει. Τέλο πάντων, εγώ δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω. Ε, τώρα, για την προστασία των καταγγελών των πληροφοριδοτών και κατά πώς θα πρέπει οι ρήτρες εχεμήθειας ψευτικότητας να περιοριστούν στις συμβάσεις εργασίας. Ίσως υπάρχουν κάποια περιθώρια πρόοδου, αλλά ε, δεν ξέρω αν είναι ο σωστός δρόμος. Υπάρχουν α, ανάγκες για εχεμήθεια Κάποιο μου είπα πρέπει να οδηγηθούμε στην πλήρη διαφάνεια. Όχι, δεν είμαι υπέρ. Εγώ δεν θα ήθελα όλα μου τα έγγραφα να μπαίνουν ε, στο διαδίκτυο και να είναι προσβάσιμα σε όλους, γιατί υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία που είναι εμπιστευτικά και το αναγνωρίζω, έχασα από τον έλεγχο των εγγράφων μου. Είμαι υπερήφανος βέβαια για, για τον αντίκτυπο, όπως είναι και η δημιουργία αυτής της Επιτροπής, αλλά υπάρχουν υποχρεώσεις χεμήθειας ε, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σε ό,τι αφορά τώρα την προστασία των καταγγελόντων και πληροφοριοδοτών. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας πραγματικά εγώ είμαι αντικείμενο ποινική δίωξη αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ένα ενδεχόμενο και αυτό κάποιες εξαιρέσεις στη Γαλλία, αλλά θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια αρχή που κατά κάποιο τρόπο δέχεται αυτές τις πληροφορίες με ανώνυμο τρόπο και κάνει μια διαλογή ε, για το αν μια πληροφορία είναι σημαντική για το δημόσιο συμφέρον ή όχι και ορίζει και τον ε, συνομιλητή. Αν με ρωτάτε γιατί δεν στράφηκα στις δημόσιες αρχές, η απάντηση είναι ότι πολύ απλά, με βάση τις πληροφορίες που είχα στη διάθεσή μου, οι πρακτικές που κατήγγυλα δεν ήταν παράνομες τεράστια η συζήτηση. Χάρη και στι δικέ σας εργασίε. είδαμε Υπάρχει αυτή η κύκλιο του 77 που μιλάει για μια και ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν και οι έρευνες ε, τη ε, Κομισιόν ε, σε, για κάποια holding κτλ. Άρα, ναι μεν υπόκειται σε συζήτηση, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές που είναι νόμιμες, θεμητές, τι να καταγγείλει κανείς. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει κάνει κάποια πρόταση για την προστασία των πληροφοριδιωτών. Είναι ευρύτατο ο ορισμό του whistleblower. Είναι αυτό ο οποίο αποκαλύπτει πληροφορίε για το γενικό συμφέρον. Είναι ένα ευρύ, ένα γενικό ορισμό. Δεν πάει πιο μακριά. Έχουμε Ουσιαστικά ένα πλαίσιο προστασίας που προβλέπουμε για περιπτώσεις παράβασης. Δεν είναι το ίδιο αυτό. Εδώ μιλάμε ότι με την αποκάλυψη των πληροφοριών, στην Επιτροπή σας το είδαμε αυτό, με την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών πράγματι προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Δεν μιλάμε για κάποια παράβαση, αλλά για αποκάλυψη πληροφοριών. Ε, πάρα πολλές ερωτήσεις ε, μου ετέθησαν, δεν μπορώ να τις απαντήσω σε 10 λεπτά. αν επιχειρήσεις θα έρθουν σε επαφή με τα κράτη-μέλη ή κάποιοι μεσάζονται ή τα κράτη-μέλη κάνουν marketing, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Εσείς μπορείτε να αναλύσετε έπειτα αν κάποια κράτη ε, που είναι κάπως σαν φορολογική παράδειση πρέπει να κάνουν ε, κάποια να έχουν μια συγκεκριμένη επικοινωνική στρατηγική. Υπήρξαν και άλλη κάποια άλλα γραφεία ελέγχου που εμπλέκονται ε, στο LuxLeaks. Φαίνεται λοιπόν από όλα αυτά ότι ήταν συστημική πράγματι η όλη πρακτική. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες στα σχόλιά μου για τις πρακτικές αυτών των ε, γραφείων ελεγκτών. Υπάρχει η ε, δικαστική διαδικασία και η εξέταση που έχει ξεκινήσει. Απλά επαναλαμβάνω ουσιαστικά αυτά που έχουν πει άλλοι και διαπιστώνουν ότι κάποιες φορές ε, υπάρχουν κάποιοι που παίζουν σε διπλό ταμπλό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά για μένα πάρα πολύ δύσκολο να το σχολιάσω σε βάθος. Τώρα για τον κώδικα ηθικής δαντολογίας ή καλών πρακτικών, αν πρέπει να προχωρήσει περισσότερο. Είμαι ρεαλιστής. Η ηθική δεν είναι η προσέγγιση. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από μια επιχείρηση να εθετήσει πρακτικές ηθικές. Συμφωνώ με την κοινότητα των πολιτών. Μια επιχείρηση τι λόγο ύπαρξης έχει, την αναζήτηση του κέρδους. Για να το κάνει αυτό με τρόπο ηθικό, ε, πρέπει η πολιτική να βάλει κάποια όρια. Ένα κώδικα ηθική και δεοντολογία απλά θα δείξει κάποιε ασυνέπειε στι συμπεριφορέ των επιχειρήσεων, αλλά δεν νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ε, υποχρεώσουμε τι επιχειρήσει. Ο πρόεδρο διακόπτει. Αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό το σημείο, οι εκπρόσωποι αυτών των γραφείων ε, λεκτών ε, που ακροαστικά μας είπαν και μάλιστα ήταν περήφανοι ότι έχουν ο καθένας το δικό τους κώδικα ηθικής διοντολογίας. Άρα θέσαμε το ερώτημα. Και γι' αυτό σας το και σε εσά πολύ το ερώτημα. Αυτή η προσέγγιση για ένα κώδικα διοντολογία ηθικής που θα είναι κοινό για όλο τον κλάδο και όλο το επάγγελμα, όλου του επαγγελματίε του κλάδου, αν αυτό θα ήταν αποτελεσματικό. Εσεί μα απαντάτε ότι για σας όχι, δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ε, όπου εργαζόσασταν ο κώδικας ηθικής διοντολογίας ε, ήταν ε, ένα με αναφοράς, ήταν γνωστός, τον ελάμβαναν υπόψη στην καθημερινότητα, στη συμπεριφορά τους οι διάφοροι ή όχι. Απάντηση. Η απάντησή μου δεν μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία μου γιατί ήταν πολύ περιορισμένη λόγω του πλαισίου και επειδή δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να εκφραστώ. πιο πολύ την άποψή μου θα σας πω παρά ότι έχω εγώ εμπειρία. Ε, δεν είναι δεσμευτικός ένας κώδικας. Ε, ουσιαστικά μιλάμε για μια επικοινωνία. Τι δείχνουμε προς τα έξω, τι συμπεριφορά περνάμε προς τα έξω. Αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε ε, η συγκεκριμένη συμπεριφορά με ένα τέτοιο κώδικα ηθικής. Ε, Τώρα. Bon, il y a un, Ένα μέλος επιτροπής σας υπογράμισε το κουράγιο που έδειξε και είπε γιατί τόσοι λίγοι ε, συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Να σας πω πολύ απλά λόγω των ε, συνεπειών που τις οποίες φύσταμε και εγώ σήμερα. Γι' αυτό και χρειάζεται ένα πλαίσιο προστασίας στους πληροφοριοδότες, διότι εκατομμύρια εργαζόμενοι ε, βλέπουν συμπεριφορές ε, αντίθετες ε, με την ε, ηθική τους, με την έννοια της ηθικής που τους χαρακτηρίζει. Το θέμα είναι ότι θέλω να δώσω τις πληροφορίες αυτές αλλά χωρίς να υποστούν τις συνέπειες που υφίσταμαι εγώ σήμερα. Αν γίνει αυτό, αν υπάρχει αυτή η προστασία, θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Οι δημοσιογράφοι, οι δημόσιες, αρμόδιες δημόσιες αρχές διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Δύο λόγια για την οδηγία για το επαγγελματικό απόρριτο, επιχειρηματικό απόρριτο μάλλον. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες γιατί δεν εργάζομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άρα δεν γνωρίζω ακριβώς πώς έχει συζήτηση. Αυτό που μπορώ εγώ να δώσω ως μαρτυρία είναι ότι με κατηγορούν για παραβίαση του επιχειρηματικού απορρίτου. Υπάρχει στο Λουξεμβουριανό δίκαιο αυτή η ε, ρήτρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. και σίγουρα μπορεί κανείς να διωχθεί γι' αυτό, δηλαδή για παραβίαση του επιχειρηματικού απορρίτου, περιορίζει ε, τη δράση των πληροφοριοδοτών. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και αν έχουμε πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρέ. Αλλά η ίδια η φύση της οδηγίας έρχεται σε αντίθεση με τη δράση τουλάχιστον των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω πολλά για αυτό το σχέδιο οδηγίας, δεν καταλαβαίνω ακριβώς το νόημα πάντως. Ήδη υπάρχουν ε, κανόνες για την ε, πνευματική διοκτησία αν η απειλή είναι η κυβερνοτρομοκρατία, δεν ξέρω κατά πόσο μια οδηγία αλλά θα αλλάξει τα δεδομένα και το επιχειρηματικό απόρριτο πράγματι απειλεί άμεσα ε, δράση σαν αυτή ε, στην οποία προέβηνε εγώ και άλλοι πληροφοριοδότες. Γνωρίζουμε τι δυσκολίες έχουν και οι δημοσιογράφοι για να ασχοληθούμε κάποια θέματα οικονομικά. Άρα ε, παρακολεί το έργο τους η ύπαρξη αυτού του απορρίτου, του χειρηματικού απορρίτου. Για τη δική μου τώρα κατάσταση συγκεκριμένα, όπως σας είπα, ε, διώκομαι ποινικά. Δεν θέλω να επεκταθώ βέβαια. Ε, καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που συνεπάγεται βέβαια αυτή η δίωξη. μπορεί να μου παρασχεθεί σίγουρα υποστήριξη με διάφορους τρόπους ε, και στο πολιτικό επίπεδο και ήδη η πρόσκληση που μου απευθύνεται είναι συμβολική ε, ως χειρονομία και από εκεί και πέρα βέβαια Φυσικά χωρίς να περαστεί δικαιοσύνη που πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αλλά καλό είναι να υπενθυμίζουμε την ε, ε, χρησιμότητα ε, της δράσης μου. Αντιπρόεδρος Εύα Ζολή νομίζω θέλω να κάνει μια ερώτηση. Να ευχαριστήσω τον Αντών Λατούρ για την ε, κίνηση που έκανε, που επέτρεψε να δείξουμε πόσο εγκατάλειψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη μάχη και παρά την κρίση ε, έπρεπε να μας το επενθυμίσει και χρειάστηκε το LuxLeaks και ο Αντουάν Λετούρ ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή και να μπορέσουμε να θέσουμε τα διάφορα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μπαρόζο δεν αντέδρασε στα tax rulings πιο νωρί, ενώ υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία. Ήθελα να σα το πω δημοσία. Θέλω να πω ότι είστε πάρα πολύ σημαντικό για περισσότερη δικαιοσύνη στον κόσμο. Ευχαριστώ. Μάικλ Τόρερ, έχετε κι εσείς κάποιο σχόλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντελτούρ και να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε να μου πείτε εάν χρειάζεται ο κύριος Δελτούρ περισσότερο χρόνο να εξηγήσει κάτι μήπως θα έπρεπε να του δώσουμε το χρόνο. Ίσως και μετά την συνεδρίαση αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλει να μας δώσει ο κύριος Δελτούρ θα μας ενδιέφερε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ ο Φάμπιο. Ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευελιξία σήμερα. Να χρησιμοποιήσουμε ευελιξία για τον κύριο Ντελτούρ είναι και συμβολικά σημαντικό. Ξέρουμε τι, τι περνάει. Όσον αφορά τα σχόλια του κυρίου Ντελτούρ, θέλω να του πω ότι στις κατευθυντήριες γραμμές για τα μυστικά των επιχειρήσεων θέλει να επεκτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τι καλύπτουν τα επαγγελματικά μυστικά ε, και ίσως το τρόπο να μην προσφέρεται η προστασία στους πληροφοριοδότες. Όσον αφορά την προστασία, λέει ο Πρόεδρος, των καταγγελόντων, των πληροφοριοδοτών, διαβεβαιώνουμε τον κύριο Ντελτούρ και όχι μόνο εκείνον προσωπικά, αλλά και εκείνους που θα ήθελαν να κινηθούν παρομοίως ότι το Κοινοβούλιο ήδη έχει τοποθετηθεί μέσω ψηφοφορίας όσον αφορά την αρχή του αιτήματο που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τεθεί επιτάπητος μια πρόταση για προστασία των πληροφοριωτών. Οι εισηγητές θα δουν κατά πόσον πέραν αυτής της αρχής που ήδη στήριξε το Κοινοβούλιο θα προτείνουν στην έκθεσή τους να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο αίτημα που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία από αυτού στο Κοινοβούλιο και όπως δείξατε και ο ίδιος, αν και εσείς και άλλοι έχετε προσκληθεί στην αυτή την Επιτροπή, ε, είναι διότι επικρατεί αυτό το πνεύμα που σας ανέφερα. Η Άννα Γκόμερς έχει κάποιο σχόλιο να κάνει. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ σαν βουλευτής να σας στηρίξω, σας θεωρώ πραγματικά σημαντικότατο αποφασιστική σημασίας η καταγγελία σας. Να σας ρωτήσω, αποκαλύψατε ότι υπήρχαν ε, συμφωνίες, tax rulings, έχουμε και είχαμε σειρά και άλλων ωφελιών για τις ε, ε, επιχειρήσεις κατά περίπτωση φορολογικές απαλλαγές που εχορηγούνται από τις κυβερνήσεις σε ποιο βαθμό όλα αυτά είναι σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις κινήσεις των επιχειρήσεων όπως αυτή στην οποία εργαστήκατε. Ποιες σχέσεις υπήρχαν μεταξύ επιχειρήσεως και κυβερνήσεως και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ρωτήσω μετά, διότι είχαμε περιπτώσεις όπως το SwissLeaks όπως καλείται τώρα. Έχαμε και τη λίστα Λαγκάρντ ή τη λίστα Λίστενστάιν. Και οι κυβερνήσεις ε, δεν έκαναν τίποτα. Οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν κινήθηκαν. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η φορολογική αμνηστία που χορηγείται είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις οι μεγάλες τέσσερις και άλλες κινούνται για να νομιμοποιούν τα κέρδη από την φοροποφυγή από το tax dodging. Και σε ποιο βαθμό αυτές οι επιχειρήσει όπως οι μεγάλες τέσσερις, οι Big Four, παρεμβαίνουν και πιέζουν τις κυβερνήσεις να χορηγήσουν φορολογική αμνηστία στη χώρα μου. Είχαμε μία περίπτωση το 2005, μία το 2010, μία το 2012 επί πολύ βολικό για να καθαρίσουν τα κέρδη των ανθρώπων από την τράπεζα Espíritu Santu, χάρη. Και τέλος, το θέμα των ελευθέρων λιμένων. Το Λουξεμβούργο είναι Freeport, όπως και η Ελβετία. Και Σιγκαπούρη και λοιπά. Και μου λένε ότι τώρα όλο και περισσότερο είναι πιο προσελκυστικό να προσφεύγει κανείς στο Freeport για να αποθηκεύει χρεόγραφα αξιόγραφα για κάποια σειρά ετών και να μην πληρώνει φόρους. Σε ποιο βαθμό και αυτό είναι σχετικό, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζετε. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Υπερβάνος Πέρες στα γρήγορα παρακαλώ. Δύσκολο, δύσκολο να ξεκινήσω χωρίς να συγχαρώ όλο το έκανε. Νομίζω ότι είναι σωστό και κατανοητό αυτό και θεμητό. Το προσωπικό σας θάρρος συμβάλλει σε συλλογική προσπάθεια σημαντική. Από αυτή την πλευρά λοιπόν έχετε όλη τη στήριξή μας και πράγματι συγκλονιστήκαμε όταν βρεθήκατε στριμωγμένος και το είπα το ίδιος ότι κατά κάποιο τρόπο ότι χρησιμοποιήθηκαν τα έγγραφα και δευτήκατε. Αλλά στο τέλος τελικά έβγαινε κάτι καλό. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματική δυσκολία. Αναφερθήκατε στο μονοπάτι αυτό που ακολουθήσατε, ότι θα μπορούσε, είπατε, να δημιουργηθεί μια δομή που να προβαίνει σε μια δίθηση των πραγματικών από τους ψεύτικους πληροφοριοδότες. Τι πρέπει να δημοσιοποιηθεί και τι όχι. Και πράγματι υπάρχει δυσκολία εδώ. Ε, είναι το ίδιο επιχειρήμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί όταν δεν θέλει να δημοσιοποιεί κάποια στοιχεία. Είσαστε στην αρχή του προβληματισμού σας, φαντάζομαι, και εμείς θα πρέπει να δείξουμε κάποια φαντασία για να δούμε ποια δομή θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματική δυσκολία όμως. Ε, μπορούμε να συζητούμε εσαΐ διαφορετικά το επαγγελματικό μυστικό. Σε κάποια επιχείρηση θεωρείται ότι κάποια πράγματα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. Πραγματικά είμαστε στα όρια κάποιων πραγμάτων, στα σύνορα. Τι πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα της επιχείρησης, πώς μπορεί να συναλλάσσεται και τι θα πρέπει να δημοσιοποιείτε. Και αληθεύει περισσότερο στα, ε, σε αυτά που είναι ε, γραπτά. Το ανέφερε κάποιος συνάδελφος. Τι γίνεται σε επαφές που έχει με επιχείρηση με την εφορία, πώς διοργανώνεται η όλη υπόθεση και τι προβλέπει η νομοθεσία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία διασύνδεση όλων αυτών και εμείς ως νομοθέτες είμαστε εδώ ε, προσπαθώντας να συλλάβουμε κάτι πολύ δύσκολο. Αν θέλουμε να μπορούμε να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα πρέπει να κάνει στο μέλλον, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Με αυτή τη μελέτη λοιπόν ε, προβαίνουμε σε ένα, κάνουμε ένα στάδιο. Καμιά παλιά ασχολιόμασταν με την απάτη και με την απάτη, εδώ με τη βελτιστοποίηση. Πώς μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα πράγματα. Δηλαδή η βελτιστοποίηση μπορεί να είναι αντίθετη προς το γενικό συμφέρον. Ίσως πηγαίνω πολύ μακριά. Και περισσότερο εμείς θα απαντήσουμε παρά εσείς. Αν έχετε κάποιες σκέψεις όμως που συνδέονται όχι με τη μεγάλη σας εμπειρία, με τη μεγάλη σας γνώση πολλών πτυχών του θέματος, αυτό θα μας βοηθήσει και εμάς ε, ως νομοθέτες να βγάλουμε μια άκρη. Μάλιστα. Κύριε Τελτούρ, αυτές οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις έχουν κάποια απάντηση από πλευρά σας, κάποιο σχόλιο. Σε αρκετές ερωτήσεις δεν μπορώ να απαντήσω. γιατί δεν έχω τη σχετική εμπειρία. Τα θέματα που αφορούν την φορολογική αμνηστία, τα Freeport, δεν είμαι στη θέση να δώσω απαντήσεις εγώ. Βεβαίω. Υπάρχουν στρατηγικές άλλες πέραν των tax rulings. πιστοποιητικά και άλλα, τα οποία ουσιαστικά ισοδυναμούν με απουσία φορολόγησης. Γι' αυτό και έλεγα εντάχει στην παρουσίασή μου ότι το tax ruling για μένα πρέπει βεβαίως να αποκαλυφθεί σαν στρατηγική, σαν πρακτική, αλλά υπάρχει ολόκληρο ένα ζήτημα του συνόλου των πρακτικών που αξιοποιούνται. Εκεί, σε αυτό το θέμα πρέπει να γίνει αναλυφθή δράση. Και πρέπει να ε, ενσκύψουμε και στο νόλο, στην όλη προβληματική της φοροαποφυγής. Αυτό νομίζω είναι η καρδιά του προβλήματος. Πρέπει δηλαδή να αναλυθεί όλο αυτό το περίπλοκο ε, σύστημα για να εξασφαλιστεί αφενός η διαφάνεια, αφετέρου η αποτελεσματικότητα της πολιτικής εξουσίας. Και αυτό είναι θεμελιώδο σημασία για μένα. Γιατί όλες αυτές οι πρακτικές σημαίνουν αποφυγή του δημοκρατικού διαλόγου, της δημοκρατικής πρακτικής. Οι πολιτικοί έχουν σαν ευθύνη να το αποφύγουν αυτό χωρίς να θέλουμε βέβαια να απλοποιούμε ή να υπεραπληστεύουμε. Πρέπει να κοιτούμε τι είδου ε, άνθρωποι βρίσκονται πίσω από αυτά και τι είδου συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτούς. Στο επιχειρηματικό απόρριτο, παραδείγματι, τι νόημα έχει και τι εξυπηρετεί το η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλέγματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αναλογιστείτε τι είδου συμφέροντα εξυπηρετείτε. Τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης ή των επιχειρήσεων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ε, αντιφατικά μεταξύ τους ή ασύμβατα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο λησμόνησα σε σχέση με το Amazon, χωρίς να θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στην υπόθεση αυτή, αλλά γενικότερα στην στάση ορισμένων πολυεθνικών όταν βρίσκονται ενώπιον της καταγγελίας ότι έχουν επιθετική φορολογική πρακτική. Απαντούν λοιπόν, α, εμείς πληρώσαμε τόσους φόρους και ούτω καθεξής. Και εκδηλώνεται από πλευρά των επιχειρήσεων αυτών η γενεοδορία ότι θα πληρώσουμε τόσους φόρους, το ταδεκράτος και το καθεξής. Φαίνεται δηλαδή σαν να ε, είναι δωρίας η καταβολή των φόρων. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ξεπερνάμε τα όρια. Δηλαδή, τηρώντας αυστηρά τους νόμους με ορισμένε συνθήκες, μπορούμε ακόμα και να ξεφύγουμε από τη φορολόγηση. Γι' αυτό για μένα η μπαλά δεν είναι τόσο στο γήπεδο των επιχειρήσεων, όσο και αν ε, ε, αυτές καταγγέλλονται, διότι αυτές απλώς στείλουν τον νόμο. στη συνέχεια πως πρέπει να κωδικοποιηθεί η κατάσταση, η απουσία νομοποίησης, η επιθετικότητα αυτής της ε, φορολογικής πρακτικής. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Αναλύσουμε όμως ε, τα πραγματικά ποσοστά φορολόγησης, νομίζω ότι θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Αυτό άλλωστε καταγράφει και ο τύπος. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πραγματικά περιπτώσεις σοβαρών καταχρήσεων. Τελικό δε μήνυμα είναι η απουσία εσόδων φορολογικών που να προέρχονται από επιχειρήσεις και υπάρχουν σαφή δείγματα σε αυτό. Πρόεδρε. Αυτό το παράδειγμα μας έδωσε και Μάικλ Τόιρερ πριν. Δηλαδή αυτό που πλήρωνε μια μεγάλη επιχείρηση, μάλλον τα κέρδη μιας μεγάλης επιχείρησης στην Γερμανία, τα πληρώνει ως ΦΠΑ στη χώρα που έχει τη φορολογική της έδρα. Κύριε Δελτούρ, έχετε να προσθέσετε τίποτα. Δεν θέλω να σας ε, εμποδίσω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Πάντως ε, θα κρατήσουμε επαφή και το ίδιο ισχύει και με την κυρία Ρίντινγκ και όλους ε, τους καλεσμένους μας που κατέθεσαν τη μαρτυρία τους στην Επιτροπή μας και οι δύο μας συζητητές θα είναι σε μόνιμη επαφή μαζί σας. Μάλιστα, δημιουργήσαμε και μια ιστοσελίδα για ανταλλαγή απόψεων με όλους εκείνους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις ή που να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες. Μάλιστα, ε, με δύσκολους ε, νομικούς όρους και συνθήκες, γιατί Είπατε πώ μπορούμε να φανταστούμε ένα νομικό πλαίσιο που να προστατεύει του πληροφοριοδότες, του καταγγέλλοντε. Η διαφορά μεταξύ των βουλευτών και των δημοσιογράφων έγκυται στο ότι ε, δεν έχουμε εμείς το προνόμιο να μπορούμε να μην αποκαλύπτουμε τις πηγές μας, να τις κρατάμε μυστικές. Οπότε, αν κάποιος ε, μας κοινοποιήσει κάτι, καταγγείλει κάτι μέσω της ιστοσελίδας ε, γραπτός. Καταγγείλει κάποιες πρακτικές παρόμοιες με αυτές που καταγγείλατε εσείς. Δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος του από μία δικαστική αρχή. Δηλαδή, Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να κρατήσουμε την ανωνυμία και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε τη γνησιότητα όλων αυτών των εγγράφων που μας υποβάλλονται. Μας ενδιαφέρει και η γνησιότητα των εγγράφων και φυσικά η εξακρίβωση της αλήθειας όλων αυτών των περιστατικών και των γεγονότων που καταγγέλλονται. Πάντως όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε πιο διεξοδικά. Μήπως θα μπορούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μια επιφορτισμένη αρχή, μόνιμη αρχή με το θέμα αυτό. Γιατί η Επιτροπή μας είναι προσωρινή. Πάντως διαπιστώνουμε ότι και σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε άλλους, αυτό που έγινε εν θερμό ή μετά την πρώτη, μετά το πρώτο σοκ από τις μαρτυρίες και τις καταγγελίες, το έργο που θα γίνει, που γίνεται στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής και ενδεχομένως και το νομοθετικό έργο μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και ενδεχομένως κάποιες διεθνείς συμφωνίες που ευελπιστούμε ότι θα καταρτιστούν επί τη βάση των συστάσεων του ΟΣΑ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και να μην επανέλθουμε μετά από μια σύντομη περίοδο σε ακόμη πιο καταδικαστές πρακτικές. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η ε, ομιλία του κυρίου Μόντι και η αναγγελία που έκανε ότι είχε πρωτοστατήσει σε νομοθετικέ πρωτοβουλίε για να διορθωθεί μια κατάσταση που είχε διαπιστωθεί ήδη πριν από μία εικοσάετια και στην αρχή υπήρξε κάποια βελτίωση, αλλά μετά από 20 χρόνια διαπιστώνουμε ότι καταλήξαμε στα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους ε, πολιτικούς στόχους που είχαμε θέσει πριν από 20 χρόνια. Τώρα, αν αυτή τη φορά καταφέρουμε να πείσουμε όλες τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα να υπογραφεί μια διεθνή συμφωνία για να ε, καταλήξουμε σε μια δίκαιη, διαφανή φορολογική κατάσταση και να πατάξουμε αυτές τις πρακτικές, θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό που δεν θα εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες περιοχές του κόσμου για ένα προσωρινό διάστημα, αλλά παντού και στο Σας ευχαριστώ πάντως για την παρουσία σας, τα, τα, τη μαρτυρία σας και πραγματικά να σας επενέσω γιατί εγκαινιάσετε ένα νέο είδος και ένα νέο ε, χαρακτηριστικό του πολίτη να κάνει κάποιες καταγγελίες αναλαμβάνοντας την ευθύνη και ε, αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες και εκκινώντας μια συζήτηση που μετά εξαρτάται από εμά ε, να την προωθήσουμε και να ανταπεξέλθουμε στο νομοθετικό μας έργο για να βελτιώσουμε την νομική κατάσταση. Ευχαριστώ. Mes chers collègues, alors, nous... Αγαπητοί συνάδελφοι, Επαναρχόμαστε στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης τώρα, τα διάφορα δηλαδή, που προβλέπουν ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχω ανακοινώσεις σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών για τη συνέχεια των εργασιών μας. και επίσης για τις επόμενες μας συνεδριάσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανάλογα με τις εξελίξεις των εργασιών και σε συμφωνία με την Οικονομική Επιτροπή και τους α, διακεκριμένους εισηγητές Ανελίζα και Μάιερ, διαπιστώσαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουμε τη συλλογή των πληροφοριών και των συστάσεων και την ολοκλήρωση το, των, της έκθεσής μας. Γι' αυτό και με εντολή των συντονιστών ζήτησα παράταση της εντολής μας, που κανονικά θα εξέπνε στα μέσα Αυγούστου, ζήτησα παράταση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου για την Επιτροπή Τάξε, ώστε το Νοέμβριο, στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου, να υποβληθεί η έκθεσή μας ε, προς Οπότε, στο χρονοδιάγραμμα μας θα προβλέψουμε μέχρι το καλοκαίρι την ολοκλήρωση της συλλογή των πληροφοριών, της των αποστολών και των επισκέψεων. Έχουμε 18 Ιουνίου αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα δούμε ε, τι θα προγραμματίσουμε ανάλογα με και τις πληροφορίες που θα λαμβάνουμε στο, στο σελίδα. Η έκθεση στα αγγλικά θα είναι έτοιμη πριν τις θερινές διακοπές και στις υπόλοιπες μεταφράσεις μετά μέχρι το τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να έχουμε τη συζήτηση ε, της έκθεσης, υποβολή τροπολογιών, εξέταση τροπολογιών, έγκριση στην Επιτροπή Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στην Επιτροπή. Και δώσαμε στις 28 κυβερνήσεις, γιατί από το σκάνδαλο Λίξ που αφορούσε μία χώρα και μόνο, επεκτείναμε ε, το θέμα στις υπόλοιπες 27 και δώσαμε στις 28 κυβερνήσεις μέχρι τις 31 Μαΐου να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο το γραπτό. 9 ε, κυβερνήσεις ε, απάντησαν εμπρόθεσμα. Θα φροντίσουμε και οι υπόλοιπες να στείλουν τις απαντήσεις και θα σας ενημερώσουμε στο μέτρο που θα τις λαμβάνουμε. Αύριο θα γίνει εργαστήριο από το Policy Department, από το Τμήμα Πολιτικών Α, παρουσία ε, εμπειρογνωμών για τη φορολογία και πανεπιστημιακών. Σεμινάριο, workshop με θέμα τα tax rulings. Δυστυχώς ε, δεν θα είμαι παρόν, αλλά σίγουρα κάποιος αντιπρόεδρος θα είναι για να προεδρεύσει. Είπαμε για τις αντιπροσωπείες που θα στείλουμε, τις επισκέψεις. Τώρα, το επόμενο πολύ σημαντικό πολιτικό μας ραντεβού, και σας το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό, αναμένεται για τις 17 Ιουνίου. Στείλαμε επιστολή στις 28 κυβερνήσεις, στείλαμε επιστολές και στα 28 κοινοβούλια, τα εθνικά, στις αρμόδιες επιτροπές, τους επιτροπές οικονομικών συγκεκριμένα, καλώντας ε, όσους ενδιαφέρονταν για τις εργασίες μας να λάβουν μέρος αυτές ε, με όποιο τρόπο επιθυμούν. Και τους καλέσαμε όλους σε μία δημόσια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 17 Ιουνίου. Και σας στείλαμε πριν λίγες μέρες mail ζητώντας σας να συνεννοηθείτε με τους συμπατριώτες σας για να έχουμε μεγάλη συμμετοχή και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μέχρι τώρα λάβαμε επιβεβαίωση από πάνω από τα μισά κοινοβούλια για τη συμμετοχή στην διάσκεψη αυτή. 18 κράτη-μέλη επίσης έχουν απαντήσει με 6 προέδρους επιτροπών ε, οικονομικών από τα Εθνικά Κοινοβούλια και επιβεβαιώθηκε και η παρουσία του κυρίου Μιουέ που ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και ήταν και εισηγητής ε, μιας ε, αποστολής διερευνητικής παρόμοια τη δική μας πριν από έξι μήνες θα έρθει λοιπόν ο πρόεδρος αυτής της ερευνητικής αποστολής από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. καλέσαμε και την κυρία Χότζ, δεν ξέρω αν το επιβεβαίωσε, γιατί δυστυχώς για μας δεν επανεξελέγει στο Westminster. Ήταν όμως πρόεδρος στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Η ομόλογος του κυρίου Τόιερ δηλαδή από την προηγούμενη Βουλή των Κοινοτήτων και οργάνωσε πολύ σημαντικές δημόσιες ακροάσεις επί της θητείας της. Μία δημόσια ακρόαση για την Google, για παράδειγμα, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αξιοσημείωτη. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Χότς και άλλες ε, εθνικές βουλές είχαν οργανώσει παρόμοιες έρευνες. Η Ουγγρική Βουλή, για παράδειγμα, θα στείλει εκπρόσωπο. Η Βουλή της Κύπρου, πολύ σημαντική χώρα για το θέμα αυτό. Οπότε η 17η Ιουνίου θα είναι πολύ σημαντική ημέρα, ορόσημο. Οπότε σας υπενθυμίζω την πρόσκληση και παρακαλώ κοινοποιήστε το στις, στους Επιτροπών Οικονομικών των Εθνικών σας Κοινοβουλίων για να δώσουν το παρόν και φυσικά και στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Άλλο σημαντικό ορόσημο, 23η Ιουνίου. Κάποιες εκράσεις που δεν έγιναν σήμερα λόγω προσωπικών προβλημάτων των καλεσμένων έχουν ε, αναβληθεί για αργότερα. Επίσης, είχαμε και επιφυλάξεις έως και απόρριψη μερικών μεγάλων επιχειρήσεων που είχαμε καλέσει στις ακροάσεις μας και που μέχρι τώρα κολλησιεργούν. Βέβαια αυτό δεν μας ε, αποθαρρύνει επουδενή. Μάλιστα και εγώ και μερικοί από εσά ε, εκδώσατε και ανακοινωθέντα τύπου δήλωσα ότι όσους προσκαλούμε και απορρίπτουν την πρόσκληση ουσιαστικά έμεσα ομολογούν την ενοχή τους ή αφήνουν να εννοηθεί ότι έχουν πληροφορίες που δεν θέλουν να κοινοποιήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ε, επιχειρήσεις που διώκονται είτε δικαστικά είτε σε ιονή δικαστικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε δικαστικές διώξεις από τις χώρες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τις έχει στο στόχαστρο για συμφωνίες καρτέλ κατάχρησης δεσπόζουσα θέση. Και εκεί λογικό είναι να μην θέλουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις για να μην χρησιμοποιηθούν εις βάρος τους οι δηλώσεις τους. Αλλά στον κατάλογο που έχουν συντάξει οι συγητές μας και τον οποίο έχουν εγκρίνει οι συντονιστές, εμείς είπαμε τουλάχιστον έξι ε, πολυεθνικές να καλέσουν από διάφορες χώρες, από διαφορετικούς τομείς, δύο αμερικανικές πολυεθνικές, τέσσερις ευρωπαϊκές πολυεθνικές, κάποιες τις κλασικής οικονομίας, άλλες της ψηφιακής οικονομίας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα πράγματα. Ο στόχος μας δεν είναι να δηλώσουμε ότι καλέσαμε την τάδε επιχείρηση γιατί είναι εκ των προτέρων ύποπτη. Αλλά θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε πώς μια μεγάλη επιχείρηση, μια τράπεζα, μια ασφαλιστική επιχείρηση, μια πετρελαϊκή, μια αυτοκινητοβιομηχανία, μια αεροναυπηγική επιχείρηση, πώς ε, καταρτίζουν τη φορολογική του στρατηγική. Γιατί οι πολυεθνικές έχουν φορολογική στρατηγική φορολογικό προγραμματισμό. Μερικές εθνικές βουλές το κατάφεραν να έχουν τέτοιες ακροάσεις. Θέλω και εμείς να το επιτύχουμε. Και μάλιστα αναφέρω το παράδειγμα της Amazon. Αν τελικά είναι συνεπής με τις δηλώσεις που έκανε η επιχείρηση αυτή, θα πρέπει να είναι η πρώτη που θα έρθει η Amazon να κάνει την ομιλία και να παρουσιάσει τη μαρτυρία της. Δίνοντας το καλό παράδειγμα, και κινητοποιώντας μια χιονοστιβάδα τέτοιων παρουσιών. Όλα αυτά θα γίνουν στις 23 Ιουνίου. Και κατόπιν έχουμε και τις άλλες κυβερνήσεις, τους άλλους υπουργούς. Στείλαμε επιστολή σε 28 κυβερνήσεις και στις 28 κυβερνήσεις. Λάβαμε νέα απαντήσει στο γραπτό ερωτηματολόγιο και επίσης ε, μερικοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Κάποιοι υπουργοί μας είπαν πολύ ευχαρίστως να συνεργαστούμε. Μάλιστα μερικοί είπαν ορίστε περάστε σε εμάς, ελάτε στη χώρα μας. Ε, ο Εσθονός για παράδειγμα υπουργό, η Πορτογαλίδα υπουργό. Άλλοι είπαν ό,τι θέλετε, πολύ ευχαρίστω. Να ακόμη να έρθουμε, να και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συναντήσουμε τους συζητητές, το Προεδρείο σας, τους συντονιστές ή και σε μια δημόσια κρόση ακόμη να παραστούμε. Είχα και εγώ προσωπικές επαφές και οι συγητές μας. Εγώ είχα προσωπική συνομιλία με μερικούς από αυτούς τους υπουργούς και αυτό προσπαθούμε να οργανώσουμε φυσικά με την έγκριση και την εθάριση των συντονιστών είναι να έχουμε ακρόαση με πολλούς υπουργούς ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Πέραν αυτό που θα συναντήσουμε στην πατρίδα τους στο περιθώριο του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ που θα γίνει τον Ιούλιο. Γιατί θα γίνει ένα Συμβουλίο ΕΚΟΦΗΝ τον Ιούνιο, αλλά στο Λουξεμβούργο. Γιατί τον Ιούνιο τα Υπουργικά Συμβούλια γίνονται στο Λουξεμβούργο. Αυτό δεν μα βολεύει και πολύ. Αλλά θα έχουμε στι 14 Ιουλίου Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και εδώ στι Βρυξέλλε. Και μάλιστα στι 13 Ιουλίου το απόγευμα θα συνεδριάσει το Eurogroup. Οπότε αμέσως πριν το Eurogroup σκεφτήκαμε να προσκαλέσουμε μερικούς υπουργούς. Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε έτοιμος. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί και μάλιστα με εξουσιοδότησε να σας το ανακοινώσω. Βέβαια δεν θα θέλαμε να περιοριστούμε σε έναν υπουργό και μόνο. Να καλέσουμε και τον Εσθονό, τον Πορτογάλο, τον τον Πολωνό Υπουργό, που επίσης είναι πρόθυμος να έρθει. Ο Γάλλος Υπουργός είπε ότι αν έρθει ο Γερμανός ομολογός του, θα ήταν θεάρεστο. Και νομίζω ότι πολύ συμφωνούμε. Και μάλιστα ο ίδιος έχει επαφή με τον Γερμανό ομολογό του και εγώ το ίδιο. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί θα ήταν ευχή έργο να παραστήκε εκείνο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα και το θέμα είναι να έρθει και ο, και ο Υπουργός Πάντοβαν, ο Ιταλός. Γιατί μετά το LuxLeaks οι τρεις ε, υπουργοί είχαν συνυπογράψει επιστολή ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία. Και αν δεν κάνω λάθος και ο Ισπανός υπουργό που ε, μας είχε καλέσει στη Μαδρίτη, ο κύριος Λουίς Δεγκίντος, δεδομένης κατάστασης της χώρας του αλλά και ενδεχομένως λόγω των προσωπικών του φιλοδοξιών για το μέλλον μάλλον δεν θα έρθει. Αν καταφέρουμε όμως τουλάχιστον έξι υπουργού να έχουμε, δεν μπορούμε φυσικά να έχουμε το σύνολο του Eurogroup, αλλά τουλάχιστον έξι υπουργού στην ίδια δημόσια ακρόαση για να τους υποβάλουμε ερωτήσεις έχοντας αναλύσει τις γραπτές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και να τους ρωτήσουμε τι γίνεται στη χώρα τους. Βέβαια όλοι θα πούν ότι είναι οι καλύτεροι μαθητές, αλλά δεν είναι όλοι. Επίσης, ε, να τους ε, δώσουμε τη γνώμη μας για το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στο μεταξύ θα έχει υποβληθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα, θα έρθει στις 2 Ιουλίου, άλλο σημαντικό ορόσημο, σε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών, θα μας παρουσιάσει το νομοθετικό της πακέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα τους δώσουμε τις εντυπώσεις μας για το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο δράσης του ΩΣΑ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό λοιπόν για όλους και κυρίως για τους εισηγητές. Τώρα, ο κύριος Στόιρερ ζήτησε το λόγο, ο εισηγητής μας. Έχεις το λόγο, Μίκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε ότι έχω συχνά επικρίνει και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες πάλι ε, και γι' αυτό θα ήθελα να σας συγχαρώ ρητά, Πρόεδρε, γιατί καταφέρατε να κερδίσετε την παρουσία του Γάλλου Υπουργού των Οικονομικών στην Επιτροπή μας. Σας ενθαρρύνω λοιπόν και εσάς και όλους τους, και τους εισηγητές από τις ε, δύο ομάδες να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσκαλέσουμε τους Υπουργούς των Οικονομικών στην Επιτροπή μας. Πρόκειται για ένα θέμα κεντρική σημασία, ένα πολύ σημαντικό θέμα, πρέπει να το συζητήσουμε. Οι πολίτες της Ευρώπης ρωτώνται γιατί δεν έχουμε μπορέσει να εξασφαλίσουμε ή δεν έχουν μπορέσει οι Υπουργοί των Οικονομικών στη διακυβερνητική λύση να βρουν ε, απαντήσει στα προβλήματα αυτά. Αυτό λοιπόν θέλω να υπογραμμίσω και ιδιαίτερα σημαντική για μένα και την ομάδα μου είναι η υπόθεση των προσκλήσεων στις πολυεθνικές, τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εάν δεν ε, καταδέχονται να έρθουν στην Επιτροπή μας, νομίζω ότι το μόνο μπορούμε, ο μόνος χαρακτηρισμός που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι πρόκειται για σκάνδαλο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ε, μία ε, λύση όπου μπορεί να εξασφαλίζει κάθε επιχείρηση όπως θέλει τις καλύτερες δυνατές ε, συνθήκες αλλά όταν έρχεται η ώρα θα πρέπει να αναγνωρίζετε ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το διεθνές πλαίσιο που έχει πλέον διαμορφωθεί να εξηγούν οι Starbucks, οι Emerson, οι Fiat, άλλες επιχειρήσεις πολυεθνικές να εξηγούν όλες αυτές που έχουν εμπλακεί στα Lux Clicks και οι άλλες μεγάλες τράπεζες όπως η Commerzbank ή η Deutsche Bank από τη Γερμανία που έρχομαι εγώ θα πρέπει να έρχονται λοιπόν και να μας εξηγούν τη δική τους προοπτική. Έχετε λοιπόν την αμέριστη υποστήριξή μου, Πρόεδρε και σας ε, παρακαλώ να απευθύνετε και πάλι το αίτημα στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Να επιμείνουμε και να πιέσουμε ώστε να έρθουν εκπρόσωποι των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Επιτροπή μας για να τις ακούσουμε. Ο Πρόεδρος. Βεβαίως. Δημοσιοποιούμε και... Ναι, θα σας δώσω το λόγο, Πίτερ. Δημοσιοποιούμε συστηματικά τις προσκλήσεις που κάνουμε γραπτός και απαιτώ και γραπτή απάντηση και δημοσιοποιούμε και την απάντηση. Και αν δεν υπάρχει βέβαια αλλαγή γνώμης, θα μπορούσαμε να πάμε στο επίπεδο του Προέδρου του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα, Πίτερ. Ναι, θα ήθελα εδώ ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να καθίσταται γνωστό στην κοινή γνώμη ποια είναι η επιχείρηση, ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν δέχθηκαν την πρόσκλησή μας σε ακρόαση. Αυτό όχι μόνο μέσω τη ιστοσελίδα μα, αλλά με έναν τρόπο ο οποίο να είναι πραγματικά προσιτό στην κοινή γνώμη, να ενημερώνεται και να ασκήσουμε με τον τρόπο αυτόν πίεση στις, μικρο... στις ε, πολυεθνικές αυτές επιχειρήσεις ώστε να έρθουν να μας μιλήσουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ αυτό που προτείνω είναι, έχουμε την επόμενη εβδομάδα την σύνοδο στο Στρασβούργο. Αυτό που προτείνω λοιπόν είναι να επαναλάβουμε τη να κάνουμε τη ρελάνς αυτή τη βδομάδα ήδη και να δούμε τις οριστικές απαντήσεις που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο. Και θα κάνουμε και μια ε, συνέντευξη τύπου με τους, με τους συζητητές, ώστε να πούμε ξεκάθαρα εμείς έχουμε στείλει αυτές τις προσκλήσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις που έρχονται και άλλες που ξέρουμε πως δεν θα έρθουν. Και έτσι τα πράγματα θα είναι ξεκάθαρα. Συμφωνείτε, Ελίζα. Ναι, αυτό θα ήθελα κι εγώ ακριβώς. Μόνο μια ερώτηση σε σχέση με τον κύριο Μάριο Σκόλλα. Δεν κατάλαβα αν υπήρξε πρόβλημα μετακίνησης ή αν αρνήθηκε. Δεν κατάλαβα καλά όταν είπατε τα σχετικά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δυσκολίες να τον βρούμε δεν μπορούμε να έρθουμε να... σε επαφή μαζί του. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εμείς του είχαμε στείλει την πρόσκληση στις γνωστές του διευθύνσεις αφήνοντας και μηνύματα στα γνωστά τηλέφωνα και με βάση τα στοιχεία που λάβαμε από δημοσιογράφους και δεδομένου ότι δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του για σήμερα Άρα η σημερινή πρόσκληση ακυρώθηκε στην ουσία, αλλά ισχύει για τις 23 Ιουνίου. Ελπίζω πως μέχρι τότε θα καταφέρουμε να έρθουμε σε επαφή. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πέρα στην συνεδρίαση.